Καλημέρα. Καλώς ήρθατε στην τελευταία μας συνεδρίαση για τον Ιόνιο. Και είναι η τελευταία φορά που καλωσορίζουμε ως προεδρεύοντα του Συμβουλίου τον Ζόλταν Σέφελβεϊ, τον ε, Ούγγρο Υπουργό ανταγωνιστικότητας κάτι το οποίο ξέρω ότι παίρνει πάρα πολύ σε σοβαρά ε, ο κύριος Υπουργός ε, συμμετείχε ενεργά στην Επιτροπή μας και όσοι είχαμε πάει στη Βουδαπέστη γνωρίζουμε πως ε, ήταν και εκεί πέρα πάρα πολύ κινητικός διπνήσαμε μαζί και με την ομάδα του και Ξέρω πως είχε δώσει πάρα πολύ σημαντική όθηση στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί η άποψή μου είναι πως το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας είναι πάρα πολύ σημαντικό αλλά είχε χάσει λίγο το δρόμο του λόγω αβεβαιότητας για την αποστολή του και γιατί βεβαίως υπήρχαν πολλοί και διάφοροι υπουργοί αλλά νομίζω κύριε Υπουργέ ε, δώσατε μια νέα όθηση και ελπίζω η επόμενη υπουργοί να ακολουθήσουν έτσι. Νομίζω και ο Πολωνός σκοπεύει να κάνει το ίδιο. Εκτιμάμε λοιπόν το ότι ήρθατε στην Επιτροπή μας και επί τη ευκαιρία θέλω να ευχαριστήσω δημόσια και την ομάδα σας εδώ στις Βρυξέλλες ειδικά τον πρέσβη τον κύριο Βάς, τον οποίο έχουμε δει πάρα πολύ και την κυρία Κέρτες που σας συνοδεύει σήμερα και ασχολείται με πάρα πολλά θέματα και όπως ξέρετε στις 10 η ώρα η Επιτροπή μας θα εγκρίνει νομίζω μπορώ να πω τη συμφωνία που επιτύχαμε με, τη με την Προεδρία για την οδηγία δικαιωμάτων των καταναλωτών. Πολύ σημαντικό νομοθέτημα. Και βεβαίως ε, αυτό οφείλεται και στην συνεργασία της δικής σας ομάδας μαζί μας για αυτόν τον δύσκολο συμβιβασμό. Και αυτό είναι κάτι που εκτιμούμε. Σας ευχαριστούμε λοιπόν και ελπίζουμε πως θα έχετε την ευκαιρία να κάνετε ένα διάλειμμα καθώς θα αναλάβει άλλη Προεδρία. Οπότε χαίρομαι ιδιαίτερα που σα καλωσορίζω και θέλω να σας παρακαλέσω να μιλήσετε στην Επιτροπή για τις προκλήσεις που έχουμε, να κάνετε κάποιες σκέψεις για το μέλλον. Οπότε έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Ε, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ και θα σας εκφράσω κάποιες σκέψεις για την Προεδρία μας. Ε, ξέρετε, ήταν ε, μια ταραχώδης περίοδος για πολλούς λόγους. Βλέπετε τι συμβαίνει στην Ευρώπη και νομίζω ότι ήταν ταραχώδης περίοδος και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αντιμετωπίζουμε μια περίεργη κατάσταση στην Ευρώπη γιατί νομίζω ότι αν δείτε τι συνέβη την τελευταία δεκαετία κυρίως στην ανταγωνιστικότητα η Ευρώπη έχασε πάρα πολλές ευκαιρίες έτσι λοιπόν έπρεπε να ενισχύσουμε και να προωθήσουμε την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης εδώ παρευρέθηκα πριν δύο μήνες ε, και θυμάμαι ότι ο διευθυντής ε, της ομάδας του χρηματιστηρίου του Λονδίνου είπε ότι κοιμόταν ε, η Ευρώπη και είχε λάβει και ένα υπνοτικό. Έτσι λοιπόν ήταν πάρα πολύ γλαφυρή η παρομοίωση. Εγώ δεν θα το έλεγα τόσο γλαφυρά. Ε, και απλώς ε, θα πω ότι και οι άνθρωποι ε, έγιναν οκνηροί αλλά και οι κυβερνήσεις μπήκαν σε μια παραλόγη διαδικασία. Εγώ νομίζω ότι δεν κατόρθωσαν την τελευταία δεκαετία οι κυβερνήσεις να προωθήσουν τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. Γι' αυτό πρέπει να προωθήσουμε σημαντικές μεταρρυθμίσεις και να ξυπνήσουμε την Ευρώπη. Ξέρω ότι τώρα όλη η προσοχή δίνεται ε, στην ε, διαχείριση της δημοσιονομικής κρίσης, όμως η δημοσιονομική σταθερότητα αυτή καθ' αυτή δεν δημιουργεί θέσεις εργασίας, δεν δημιουργεί παραγωγικότητα, ούτε ανάπτυξη. Έτσι λοιπόν ε, χρειαζόμαστε δημοσιονομική σταθερότητα ε, και πρέπει να ενδυναμώσουμε τις προσπάθειές μας για να ενδυναμώσουμε την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης για να δημιουργήσουμε ένα ευνοϊκό επιχειρηματικό πλαίσιο που μπορούν να ανθίσουν οι επιχειρήσεις και να δημιουργήσουν περισσότερες θέσεις εργασία. Αν δούμε δηλαδή τι χρειάζονται οι επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν, και για να δημιουργηθούν νέες εργασίες έχουμε τέσσερις ε, απαιτήσει ε, που βρέθηκαν και στο επίκεντρο της άσκησης της Ουγγρικής Προεδρίας. Πρόκειται λοιπόν για την ενιαία αγορά, περισσότερη ενιαία αγορά ή λιγότερος κατακαιρματισμός της ενιαίας αγοράς θα έλεγα. Το δεύτερο που χρειάζονται οι επιχειρήσεις ε, και η οικονομία είναι λιγότερη γραφειοκρατία. Πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον όπου μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι λειτουργούν επιχειρήσεις με λιγότερο κόστος, πρέπει να έχουν κατάλληλη πρόσβαση στη χρηματοδότηση, που δεν είναι κάτι τόσο εύκολο ε, και μάλιστα τον τελευταίο καιρό και τέταρτη απέτηση είναι να απελευθερωθεί το δυναμικό καινοτομία των επιχειρήσεων. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με την πρώτη απέτηση περισσότερη ενιαία αγορά και λιγότερος κατακαιρματισμός ε, ε, κατά τη διάρκεια της ε, Ουγγρικής Προεδρίας. Το Συμβούλιο υιοθέτησε την πράξη για την ενιαία αγορά, Single Market Act, και αποφασίσαμε επί 12 σημαντικών προτάσεων που θέλουμε να προωθήσουμε και θέλω να ευχαριστήσω και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που υποστήριξαν το έργο αυτό. Όταν φυσικά βλέπουμε την ενία πράξη για την αγορά, προκύπτουν κάποια ερωτηματικά, αλλά νομίζω ότι η πράξη για την ενιαία αγορά μπορεί να υπερβεί τις προκλήσεις όταν μιλάμε για πολιτική ενιαίας αγοράς Έχουμε και την πρόκληση μόντι, ξέρετε, όχι μόνο υπάρχει κατακαιρματισμό της ενιαίας αγορά, αλλά και της πολιτική για την ενιαία αγορά. Αν δείτε πόσε επιτροπές, επίτροποι ασχολούνται με το θέμα αυτό. Έτσι λοιπόν από πολιτική σκοπιά Δεν είναι βέβαια τόσο άσχημα τα πράγματα. Μπορούμε να εντοπίσουμε τα διάφορα προβλήματα στην ενιαία αγορά, αλλά νομίζω ότι πρέπει να υπερβούμε αυτά τα προβλήματα και να δούμε συνολικά το θέμα της ενιαίας αγοράς. Η δεύτερη πρόκληση που τίθεται στην ενιαία αγορά νομίζω ότι είναι ε, πρόκληση ε, ε, για το διάλογο, δηλαδή χρειαζόμαστε δημόσια υποστήριξη για την ενιαία αγορά. Και η τρίτη πρόκληση όταν μιλάμε για την ενιαία αγορά ε, είναι, είναι μια προσέγγιση που συνίσταται στο εξής, δηλαδή ότι δεν καταλαβαίνει ο πολίτης ε, ότι λείπουν κάποιες σύνδεσμοι, ότι είναι ατελής η ενιαία αγορά, υπάρχουν συμφορήσεις κτλ. Νομίζω ότι πρέπει να εντοπίσουμε τα προβλήματα. Αυτό είναι σημαντικό, αλλά είναι και αποθαρρυντικό ταυτόχρονα. Χρειάζεται να κάνουμε περισσότερα. Η πράξη για την ενιαία αγορά μα δίνει μια καθολική πλατφόρμα για όλα τα θέματα που υπάρχουν επιτάπητο σήμερα. Και υπάρχει κάτι ακόμη που δεν πρέπει να ξεχνάμε. Η ενιαία αγορά έγινε ένα από τα μεγαλύτερα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Ευρώπης. Υπάρχουν πάρα πολλές συζητήσεις για την παγκόσμια θέση της Ευρώπης. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μια τόσο υψηλά ολοκληρωμένη ενιαία η αγορά λείπει στην Κίνα, στη Βραζιλία. Έτσι λοιπόν αυτή είναι η μεγαλύτερη επιτυχία μας και το μεγαλύτερο ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα και βεβαίως είναι κάτι που θα πρέπει να επικαιροποιείται και να ενημερώνεται κάθε φορά. Και η πράξη για την ενιαία αγορά στην περίπτωση αυτή δεν εμβαθύνει απλώς την ενιαία αγορά, αλλά την επικαιροποιεί επιπρόσθετα. Η πράξη για την ενιαία αγορά ε, θέτει, παρουσιάζει τα θέματα που έλαβαν χώρα τα τελευταία 10-15 χρόνια, κυρίω ό,τι αφορά τι ψηφιακέ εξελίξει, το διασυνοριακό εμπόριο κτλ. Έτσι λοιπόν, ε, χαίρομαι πάρα πολύ που η Ουγγρική Προεδρία μπόρεσε να δώσει το πράσινο φως ε, για αυτές ε, τις προτάσεις και προσωπικά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο για αυτό το έργο. Τα, η οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών είναι επίσης ε, πάρα πολύ σημαντική για να αντιμετωπίσει τον κατακαιρματισμό της αγοράς και για να διασφαλίσει τις διασυνοριακές συναλλαγές και επίσης σε κάποιο βαθμό η οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών επικαιροποιεί ο προβληματισμό των όσων συνέβησαν τις τελευταίες δεκαετίες. Αναφέρομαι και στις ε, τεχνικές εξέλιξεις για το εμπόριο. Έτσι λοιπόν, ε, ανυπομονώ για αυτή τη συνεδρία και ελπίζω ότι επίσης θα αποτελέσει μια επιτυχία. Λοιπόν, το δεύτερο στοιχείο που χρειάζονται οι επιχειρήσεις ε, για να αναπτυχθούν και να δημιουργήσουν περισσότερες θέσεις εργασία ε, είναι να απελευθερώσουμε τις ικανότητες ε, και το δυναμικό καινοτομία των επιχειρήσεων. Υπάρχει μία άμεση σχέση μεταξύ της ενός αγοράς και της καινοτομίας. Μιλάμε πάρα πολύ για καινοτομία, αλλά νομίζω ότι η σχέση είναι άμεση όσο πιο πολύ εμβαθύνουμε στην νέα αγορά, ε, ε, τόσο πιο οικονομικά αποδοτικό είναι να επενδύουμε στην κοινοτομία. Σκεφτείτε, αν επενδύουμε ε, στην αγορά και έχουμε μια αγορά με 5 10 εκατομμύρια καταναλωτές, διαφέρει πάρα πολύ. Είναι πολύ πιο αποδοτικός πρωτοκόστος να επενδύει κανείς στην κοινοτομία. Και φυσικά όταν υπάρχει μεγαλύτερη αγορά υπάρχει και μεγαλύτερος ανταγωνισμός. Επομένως αυτό ευνοεί και την καινοτομία. Επομένως βλέπουμε αυτούς τους συνδέσμους. Όταν ε, μιλώ για την ε, τελευταία δεκαετία ή τις ε, τελευταίες ευκαιρίες στην τελευταία δεκαετία βλέπουμε κάτι τέτοιο ιδιαίτερα στην καινοτομία. Δηλαδή η καινοτομία αφέθηκε μόνη της χωρίς καμία υποστήριξη και αρρωγή. Νομίζω όμως ότι αλλάζουν τα πράγματα, αλλάζει η προσέγγιση και κατά τη διάρκεια της Ουγγρικής Προεδρίας. Νομίζω ότι και εμείς επιδείξαμε κάτι τέτοιο. Ίσως ε, θα ακούσατε ε, αυτή τη διάσημη δήλωση του Πρόεδρου Ομπάμα. Ε, είπε ότι ξέρει Χρειάζεται μια στιγμή σαν το Σπούτινικ για να ξαναρχίσουμε. Πρέπει ουσιαστικά να προσφέρουμε καινοτομία και εκπαίδευση στον υπόλοιπο κόσμο. Έτσι λοιπόν πρέπει να προσφέρουμε καινοτομία και παιδεία στον υπόλοιπο κόσμο. Τίποτα το καινούριο δεν υπάρχει εδώ. Οι οικονομολόγοι ξέρουν ε, ακριβώς πάντοτε ότι πρέπει να βλέπουμε τις λεπτομέρειες ε, και όχι μόνο την ευρύτερη εικόνα. Πρέπει να διαδώσουμε τη γνώση. Πού δημιουργεί αυτό το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Γι' αυτό χαίρομαι πάρα πολύ ε, να σας ενημερώσω ότι κατά τη διάρκεια της Ουγγρικής Προεδρίας το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της 9 Μαρτίου έδωσε το πράσινο φως ε, στο ενέο σύστημα για το δίπλωμα βρεσιτεχνία, το οποίο το αναμέναμε πάρα πολύ, ήταν ιστορική στιγμή. Νομίζω ότι δεν ήμουν ιδιαίτερα μετριόφρον ε, όταν ε, κατόπιν από αυτή τη απόφαση ε, είπα στη συνέντευξη τύπου ότι γράφτηκε ιστορία, ήταν ιστορική στιγμή. Και πραγματικά ήταν παράξενο για μας για την Ουγγρική Προεδρία να ζήσουμε μια τέτοια ιστορική στιγμή. Γιατί είδα όλο το ιστορικό και είδα ότι πραγματικά για 15 χρόνια αγωνιζόταν η Ευρώπη για να έχουμε ένα ενιαίο σύστημα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Ε, πολλές φορές περνούσαν και 10 χρόνια και τίποτα δεν συνέβαινε. Όμως ε, κάποια στιγμή την θέσαμε σε εφαρμογή αυτή την ιδέα. Στις 10 ε, Δεκεμβρίου κατά τη Βελγική Προεδρία είχαμε το Συμβούλιο Αντιγωνιστικότητας. Θυμάμαι ότι είχε καταλήξει σε αδιέξοδο και χρειάζονταν 12 χώρες για να ξεκινήσουν προθυμένη συνεργασία. Έτσι λοιπόν στις 9 ε, Μαρτίου είχαμε ε, τις 25 ε, χώρες λιομιλητής που συμφώνησαν στην ενισχυμένη συνεργασία και έτσι γράψαμε ιστορία για τα, για τα διπλώματα ευρεσιτεχνία. Και φυσικά τα διπλώματα ευρεσιτεχνία είναι σημαντικά για την καινοτομία, όχι γιατί είναι πιο απλά και πιο φτηνά, γιατί κάποιοι μας ρώτησαν πόσο πιο φτηνό θα είναι αυτό το νέο σύστημα. Εγώ νομίζω ότι είναι σημαντικό να έχουμε ένα πιο ασφαλές σύστημα σε σχέση με σήμερα γιατί και σήμερα βλέπουμε ότι μπορεί κάποιος ε, να έχει το δίπλωμα πριστεχνία σε μία χώρα και να μην καλύπτεται σε άλλη χώρα και στην άλλη χώρα μπορεί να παραχθεί αυτό το προϊόν. Και έτσι προκύπτουν κάποια νομικά προβλήματα. Δεύτερον, αν ε, έχουμε αυτό το νέο σύστημα διπλώματο ευρεσιτεχνία, ε, που είναι και πιο ασφαλέ από νομική σκοπιά και πιο φθηνό και πιο απλό, υπάρχει και το πλεονέκτημα ότι οι επενδυτέ μπορούν να ελκύσουν ιδιωτικό κεφάλαιο πολύ πιο εύκολα. Και όταν μιλάμε για την καινοτομία και τα κοινά στην καινοτομία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, νομίζω ότι είναι ένα καθοριστικό βήμα. Τώρα εργαζόμαστε επί των εφαρμοστικών μέτρων και δεν είναι και τόσο εύκολα τα πράγματα. Γι' αυτό αποφασίσαμε να έχουμε ένα έκτακτο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας στις 27 Ιουνίου και ελπίζουμε να καταλήξουμε σε μια γενική προσέγγιση επί αυτού των πολύ σημαντικών εφαρμοστικών μέτρων Έτσι λοιπόν, να ακολουθήσαμε το σχέδιό μας στην περίπτωση αυτή και προωθήσαμε το όλο ζήτημα των διπλωμάτων ευρεσιτεχνία. Λοιπόν, όταν μιλάμε για το δεύτερο σημείο, λιγότερη γραφειοκρατία, πώς ε, μπορούν να λειτουργούν ε, λιγότερο δαπανηρά οι επιχειρήσεις. Είναι δυνατό οι πολισίες ε, ε, να εντάσσονται σε ένα σύστημα ε, μικρότερης λογοδοσίας. Και επίσης έχουμε και το κανονισμό SMART και αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα προς τα μπρος Δηλαδή πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα κανονιστικό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις που να είναι λογικό και ε, ευφυές. Τώρα, το Small Business Act ήταν ε, τεράστιο επίτευγμα η πράξη για τις ε, μικρές επιχειρήσεις και νομίζω ότι καλύπτει όλα τα ζητήματα που είναι σημαντικά για τις εταιρείες όχι μόνο θέματα αριθμιστικού πλαισίου, αλλά και θέματα πρόσβαση στη χρηματοδότηση και επίση, βελτίωση σύμφωνα με το θέμα της λεγόμενης διακυβέρνησης, τιμολόγηση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, πρέπει να το σχάρει, γιατί νομίζω ότι το πρόβλημα για τις μικρές επιχειρήσεις δεν είναι ότι είναι μικρές, αλλά ότι είναι μόνες τους. Και αυτό σημαίνει ότι τους λείπει η πολιτική φωνή που χρειάζεται για να επηρεάσουν το κανονιστικό πλαίσιο. Οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν αυτή την πολιτική φωνή, αλλά δεν ισχύει κάτι τέτοιο για τις μικρές επιχειρήσεις. Και νομίζω λοιπόν ότι το Small Business Act, η πράξη αυτή, αλλά και το θέμα της διακυβέρνησης είναι πολύ σημαντικά Αν δείτε λοιπόν όλο αυτό το ζήτημα, τι χρειάζονται οι επιχειρήσεις ε, για να αναπτυχθούν και να δημιουργήσουν περισσότερες θέσεις εργασίας για να εξέλθουν από την κρίση και να είναι ανταγωνιστικά στην Ευρώπη. Νομίζω Όλα αυτά είναι σημαντικά. Έχουμε και το θέμα της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, δηλαδή να βαθύνουμε στην νέα αγορά, να απελευθερώσουμε το δυναμικό της καινοτομία και να μειώσουμε το διοικητικό άχθος για τις επιχειρήσεις. Η Ουγγρική Προεδρία πέτυχε όσα ήταν δυνατό να πετύχει και φυσικά θέλω να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους για τις προσπαθίες τους στην περίπτωση αυτή και Θέλω να ευχαριστήσω και τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ξέρω ότι η κύρια πρόκληση στην Προεδρία είναι πώς να συνεργαστούμε με τους υπόλοιπους παίκτες, δηλαδή με τα κράτη-μέλη, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με την Επιτροπή. Γιατί πρέπει όχι μόνο να συνεργαστούμε, να συνεργαστούμε και τη σωστή χρονική στιγμή. Γιατί αν το Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο ή η Κομισιόν καθυστερούν δύο-τρεις εβδομάδες, δυο δύο-τρει έχουμε τόσο μεγάλη πίεση χρόνου που δεν μπορούμε πλέον να σημειώσουμε επιτυχία. Έτσι λοιπόν, εγώ χαίρομαι πάρα πολύ και θέλω να σας ευχαριστήσω τα μάλα που σε αυτή την περίπτωση η συνεργασία ήταν τόσο καλή ήταν τόσο επιτυχή η συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί χωρί τη δική σα αρρωγή δεν θα μπορούσαμε να έχουμε πετύχει αυτό το σημαντικό βήμα που θέτει την Ευρώπη σε μια τροχιά, σε μια πιο ανταγωνιστική τροχιά από ό,τι πριν. Ξέρετε ότι η Ουγγρική Προεδρία έχει αυτό το σύνθημα «Ισχυρή Ευρώπη», «Strong Europe». Και αν σκεφτώ πίσω στον Ιανουάριο, νομίζω ότι από τότε έγινε πιο ισχυρή η Ευρώπη βήμα το βήμα. σιγά σιγά θα εξέλθουμε από αυτή την κρίση και φυσικά αυτό χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε πολύ περισσότερη ε, ανταγωνιστική Ευρώπη και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που προσωπικά συμμετείχα σε αυτές τις εξελίξεις. Σας ευχαριστώ. Well, thank you very much, um, for your... Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ξεκάθαρες απόψεις σας ε, και τη φιλοδοξία στα σημαντικά για εμάς συζητήματα. Η διαπράξη της ενίας αγοράς και από μας θεωρείται σημαντική και νομίζω πως μπορούμε να αναμένουμε την συνεχιζόμενη στήριξή σας στο Συμβούλιο για μέτρα για να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους ε, τα κράτη-μέλη. Και χάρηκα που αναφέρατε και την εφαρμογή της νομοθεσίας αυτής γιατί καμιά φορά θεωρούμε πως λόγια υπάρχουν, γίνονται αλλά δεν υπάρχουν αποτελέσματα και νομίζω πως εσείς συμφωνείτε μαζί μας πως πρέπει να προχωρήσουμε αυτή την υπόθεση. Έχουμε τώρα γύρω σε μισή ώρα για ερωτήσεις και συζήτηση με τον κύριο Υπουργό. Ποιο θα ήθελε το λόγο. Ο Κυριάκος. Όλοι οι παρόντες. Να ξεκινήσουμε με τον κύριο Τριανταφυλλίδη. Θέλω να ευχαριστήσω τον ε, Υπουργό για τα όσα μας είπε ε, και να ε, κάνω αναφορά και εγώ όπως και εσείς στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί στο θέμα της οδηγίας για την προστασία των καταναλωτών που πιστεύω ότι αυτή η πρόοδος οφείλεται κατά ένα μεγάλο βαθμό και στην Προεδρία. Ε, θέλω να σταθώ σε ένα θέμα που έχει αναφερθεί στην ομιλία του κύριου κύριος Υπουργός, αυτό της ε, καινοτομίας. Η Προεδρία αφιέρωσε μεγάλο μέρος του προγράμματος της στον κομμάτι αυτό της καινοτομίας σε ό,τι αφορά τον ανταγωνισμό και ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και γίνεται αντιληπτό από τα όσα έχει πει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με τη χρηματοδότηση της καινοτομίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο θέλω να μας πει ποιες δράσεις έχει αναλάβει η Προεδρία για το ενιαίο πρόγραμμα πλαίσιο χρηματοδότησης και τι έχει αφήσει ως παρακαταθήκη για να ελοποιήσει το επόμενο τρίο των Προεδριών, δεδομένου ότι προέρχομαι και από την Κύπρο και θα με ενδιαφέρει ιδιαίτερα αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Μια που υπάρχει χρόνος, νομίζω πως ε, μπορεί να απαντήσει την κάθε ερώτηση χωρίς τα κύριος Υπουργός θέλετε να απαντήσετε. Ε, καλύτερα να, να ακούσουμε δύο-τρεις ερωτήσεις, λέει ο κύριος Υπουργός. Όπως προτιμάτε. Κυρία ε, ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ, για την ε, παρουσία σας και για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση των ε, δραστηριοτήτων της Ουγγρικής Προεδρίας. Ελπίζω πως Πολλά από αυτά τα οποία ξεκινήσατε θα τα συνεχίσει η Πολωνική Προεδρία προς όφελος της εσωτερικής αγοράς. Μιλήσατε για το σύστημα των δρεσιτεχνιών. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη για το ότι καταφέραμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα σε μεγάλο βαθμό. Όχι εντελώς, αλλά πάμε προς την σωστή κατεύθυνση για να βρεθεί μια λύση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες ε, έχουν πολύ υψηλό κόστος όσον αφορά την προστασία των ε, ευρεσιτεχνιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε χαίρομαι για το ότι το σύστημα αυτό θα δώσει δυνατότητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να προστατεύσουν τα συμφέροντά τους. Έχω μία ερώτηση. Μιλήσατε για ιδιωτικά κεφάλαια για την ε, καινοτομία. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω πώς σκοπεύετε να προσελκύσετε αυτά τα κεφάλαια και πώς θα τα χρησιμοποιήσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κυρία Κοράτσα Μπίλτ, ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα ήθελα να πω το πόσο εντυπωσιαστήκαμε πολύ από εμάς από την ε, προσωπική σας δέσμευση και την αποτελεσματικότητα της ε, Προεδρίας σας σε σχέση με αυτά που μας υποσχεθήκατε πριν από έξι μήνες. Να ξαναξεκινήσει η η αγορά, να ξανάρθει η οικονομία στο προσκήνιο, ειδικά το θέμα της ανταγωνιστικότητας που ήταν συγκεκριμένο αίτημα επιβελγικής ε, Προεδρίας και όπως εξηγήσατε να φύγουν εμπόδια γραφειοκρατία και να εστιάσουμε στην καινοτομία. Βεβαίω, ο νόμος περί ενιαίας αγοράς και η οδηγία προστασίας των καταναλωτών είναι δύο επιτεύγματα της Προεδρίας σας και είμαστε ευγνώμονες βεβαίω για αυτά. Θα ήθελα να σας ρωτήσω για το θέμα των εμέσων εμποδίων και εθνικών εξαιρέσεων. Είχαμε πάρα πολύ καλό διάλογο μαζί σας και σας ευχαριστώ που δεχτήκατε την Επιτροπή μας στη Βουδαπέστη. Για το θέμα εμπορικών και φορολογικών νόμων, όπως ξέρετε η Σλοβακία πλέον απέσυρε ε, το σχετικό νόμο, όλοι καταλαβαίνουμε την κατάσταση. Θα ήθελα λοιπόν ε, να επαναλάβετε πως πράγματι υπάρχει αυτή η δέσμευση πως τα μέτρα αυτά είναι προσωρινά και σχετίζονται με την κρίση και να μας πείτε πώς έχει τώρα η κατάσταση και θα ήθελα βεβαίω να μας πείτε αν συνεχίζετε να είστε εξίσου ε, υπέρ μιας επανεκκίνησης ενίας αγοράς. Κυρία Πέρες. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε για όλες τις πληροφορίες που μας δώσατε. Εγώ θα ήθελα να θέσω στο επίκεντρο της προσοχής τους πολίτες. Δηλαδή θέλω να θέσουμε στην καρδιά της Ευρώπης τους πολίτες γι' αυτό. Θέλω να θέσω μια ερώτηση, που όμως έχει δύο σκέλη. Καταρχήν, για την Ουγγρική Προεδρία, πού τίθεται η κοινωνική διάσταση στην εσωτερική αγορά και τι σημασία δίνεται στις υπηρεσίες κοινής ωφελίας. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Uh, Κάποιος άλλος. Χάιντι. Όχι, θα θέλατε να απαντήσετε σε αυτές τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Τις δύο πρώτες ερωτήσεις θα τις απαντήσω μαζί. Μία αφορούσε χρηματοδότηση της ε, καινοτομίας και η δεύτερη ως ένα βαθμό. Όταν μιλάμε για την καινοτομία, έρευνα και ανάπτυξη, νομίζω πως έχουμε πάρα πολλές ε, διάφορες ε, πρωτοβουλίες. Τέλος πάντων, υπάρχουν αυτές οι ευφυΐες, εν πάση περιπτώσει, στον καράζ που κάνουν τις εφευρέσεις και ακούμε μετά, βλέπετε, όταν υπάρχει το επιχειρηματικό κεφάλαιο, τι έγινε με το Google, με το Sergey Brin, το Yahoo, με το Steve Jobs κτλ. Um, και διάφοροι άλλοι ήρωες αυτής της υπόθεσης. Ωραία αυτά πράγματα, ωραία ακούγονται, αλλά δεν είναι αυτή βασική, βασικός τρόπος καινοτομία. Η καινοτομία κατά κανόνα βεβαίως κινητοποιείται από τη βιομηχανία που είναι σε επαφή με τους καταναλωτές και θέλουν νέα προϊόντα για τους καταναλωτές. Νομίζω λοιπόν πως η καινοτομία ε, κατά κύριο λόγο δημιουργείται από τις βιομηχανίες και αν ξεπεράσουμε τους τους μύθους που έχουμε κατά νου περί Silicon Valley που ούτως ή άλλως δεν μπορούμε να αντιγράψουμε σε άλλα μέρη του κόσμου και γνωρίζουμε πως ε, η καινοτομία όπως σας είπα δημιουργείται κυρίως από τη βιομηχανία. Το δεύτερο θέμα είναι η χρηματοδότηση. Πρέπει να δημιουργήσουμε λοιπόν ένα ευνοϊκό κλίμα εντό του οποίου μπορεί να επενδύσει η βιομηχανία στην καινοτομία. Και το δεύτερο ερώτημα είναι ε, το ρυθμιστικό ζήτημα και το δεύτερο είναι πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα σύστημα χρηματοδότησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Νομίζω πως αυτό το οποίο είχαμε ε, στην Προεδρία μας πρώτα απ' όλα ήταν η ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος πλαισίου 7 και τα αποτελέσματά της που ήταν πως χρειαζόμαστε ένα πολύ πιο απλό σύστημα υπάρχουν πάρα πολλά και διαφορετικά μέσα και πρέπει να συνδυάσουμε τις προσπάθειές μας και τους πόρους μας και το δεύτερο ήταν σταδιακά να πάμε σε ένα κοινό στρατηγικό πλαίσιο δηλαδή να βρεθούν συνέργειες μεταξύ πολλών χρηματοδοτικών μέσων. Και αυτό σημαίνει όχι μόνο παραδείγματος χάρη να υπάρξουν κάποια χρηματοδοτικά μέσα για την έρευνα και την ε, ανάπτυξη όπως το πρόγραμμα πλαίσιο 7 και πολλά άλλα αλλά να βρεθεί και μια εναρμονισμένη βάση ε, με βάση τον κανονισμό. Θεωρώ λοιπόν πως υπάρχουν δύο τρόποι εδώ πέρα. Πρώτον να δημιουργηθεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον για τη βιομηχανία, για να επενδύσει περισσότερα και αυτό βέβαια σε έναν βαθμό είναι θέμα των κρατών μελών κάποια τα πάνε καλά, κάποια άλλοι όχι τόσο καλά και βεβαίως και στο ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να λυθούν κάποια δήματα και είναι μετά η μετάβαση από το πρόγραμμα πλαίσιο 7 στο κοινό στρατηγικό πλαίσιο η Παρασκευή που μας πέρασε υπήρχε μια πολύ μεγάλη διάσκεψη που ολοκλήρωσε την διαβούλευση με τους ενδιαφερομένους. Ήμουν ε, εγώ εκεί, επίτρεπος ε, Γκίγεν Κουίν. Βεβαίω δεν ε, υπόθηκε τίποτα από τον Επίτροπο περί χρηματοδότησης. Το ζήτημα ήταν να απλοποιηθούν οι προσπάθειες. Και το δεύτερο ερώτημα βεβαίω αφορά του, τους φόρους στην Ουγγαρία. Ναι, είναι ένα προσωρινό μέτρο και μέχρι το τέλος του 2012, δηλαδή 1η Ιανουαρίου δεν θα υφίσταται πλέον. Ε, και συχνά οι επιχειρηματίες με ρωτάνε, δηλαδή προχτές με ρώτησαν, είναι πράγματι και τους λέω ναι, πράγματι είναι θέσφατο, δεν, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Ε, είναι σαφές ε, ε, πως είναι ένα προσωρινό μέτρο. Εάν δείτε λοιπόν τις εξελίξεις και το τι έγινε την τελευταία φορά. Αυτό το μέτρο εισήχθη για πολλούς λόγους. Ένας ήταν η κατάσταση του προπολογισμού, η λεγόμενη φορολογική κρίση που υπήρχε και μας ανάγκασε να λύσουμε αυτό το, το ζήτημα. Και βλέπουμε πως τα μέτρα αυτά απέδωσαν. Ε, υπάρχει χρόνος να περάσουμε τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις και ένας στόχος της μεταρρύθμισης ήταν να έχουμε πιο ευέλικτη αγορά εργασίας. Υπάρχει και σε πολλά έγγραφα στο ευρωπαϊκό επίπεδο ούτως ή άλλως και να γίνει πιο αποτελεσματικό το κράτος. Αυτοί είναι οι δύο βασικοί στόχοι. Αλλά με αυτές τις μεταρρυθμίσεις ε, θα μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε την ουγγρική οικονομία και το χρέος και τα λοιπά χωρίς ε, άλλους εξαιρετικούς έκτακτους φόρους. Αλλά αυτό το οποίο είδα στις συζητήσεις είναι πως ε, βλέπουμε πως τα μέτρα αυτά απέδωσαν. Εάν δείτε το τι προβλήματα είχαμε στην Ευρώπη και το πως ε, η Ουγγαρία προσπάθησε να χρηματοδοτήσει το χρέος της ε, με τρόπο βιώσιμο που μπορεί να το κάνει στην αγορά, στην των ομολόγων. Είναι πολύ χαμηλά τα ασφαλιστικά κινδύνου, οι αναπτυξιακές πρόπτικες είναι ενθαρρυντικές. Τα τελευταία στοιχεία νομίζω της ανάπτυξης δείχνουν πως ε, αυτό το, το τρίμηνο ήταν αυτό με την υψηλότερη ανάπτυξη τα τελευταία πέντε χρόνια. Οπότε βλέπουμε προς βήμα-βήμα υπάρχουν αποτελέσματα. Ξέρω πως ήταν ένα ε, ζήτημα επίμαχο, αλλά ήταν για περιορισμένο χρόνο. Μας έδωσε το χρόνο που χρειαζόμασταν για να επιτύχουμε σημαντικές μεταρρυθμίσεις, γιατί χρειάζεται και χρόνος και στο Κοινοβούλιο Ναι, το να κόβει κανεί είναι απλό. Το να λέει πως θα κόψω μερικά δισεκατομμύρια είναι απλούστατο. Μια υπογραφή χρειάζεται. Αλλά το να δημιουργηθούν βιώσιμα συστήματα και για να έχουμε μεταρρυθμίσει, χρειάζεται χρόνος και αυτός ο χρόνος ήταν για μα σημαντικό. Και τώρα καθώ εφαρμόζουμε αυτές τις ε, μεταρρυθμίσει βημα βήμα-βήμα νομίζω πως ε, μια χαρά θα, θα προχωρήσουμε. Οπότε όπως σας είπα αυτό έτσι είναι και δεν αλλάζει. Λοιπόν, η κοινωνική διάσταση της ε, αγοράς ε, είναι πάρα πολύ σημαντική και βεβαίω εντάξει υπάρχει αυτή η πολύ γνωστή φράση ότι κανείς δεν μπορεί να ερωτευτεί την, την ενιαία αγορά γιατί εντάξει μπορούμε να, να την προωθήσουμε αλλά εάν δείτε αυτά τα 12 σημεία και τα 12 μέτρα στη, στο νόμο περί ενίας αγοράς υπάρχουν κάποιες ε, κοινωνικές ε, επιχειρήσεις με κοινωνική σημασία και κάποια θέματα με κοινωνική σημασία και χρειαζόμαστε και τη στήριξη των πολιτών για την ενιαία αγορά. Καμιά φορά είναι ζήτημα επικοινωνίας γιατί τα πλεονεκτήματα της ενιαίας αγοράς είναι προφανή. Αλλά οπωσδήποτε όταν βεβαίως, ε, ε, κοιτάμε τις ειδήσει, ε, αυτό το οποίο ενδιαφέρει είναι οι κακές ειδήσει, έτσι είναι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Aspect. Καμιά φορά βλέπουμε τις προβληματικές πτυχές μόνο, αλλά νομίζω πως χρειάζεται στήριξη από τους πολίτες της ενιαίας αγοράς και είναι νομίζω κάτι το σημαντικό αυτό στα 12 αυτά σημεία μπορείτε να βρείτε πολλά σημαντικά στοιχεία που αποτελούν την κοινωνική διάσταση της ενιαίας αγοράς. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλει κάποιος να επανέλθει, ή είστε ικανοποιημένοι από τις απαντήσεις. Ωραία. Τότε θα ήθελα και εγώ να αναφέρω κάποια ζητήματα, κύριε Υπουργέ. Εφόσον έχουμε, εφόσον έχουμε χρόνο στη διάθεσή μας, επανέρχομαι σε αυτό τον ενθουσιασμό που δείχνετε για την πράξη για τις μικρές επιχειρήσεις, στο Small Business Act και τι μπορούμε να καταφέρουμε σε αυτό το τομέα. Μήπως έχετε κάποιες ιδέες ε, για το πώς θα μπορούσαμε να ενισχύσουμε τον τομέα αυτό. Έχουμε διατάξει για τις δοκιμές που κάνουμε για τις μικρές επιχειρήσεις, δηλαδή δοκιμάζουμε την νομοθεσία να δούμε ποια επίπτωση έχει η μικρών επιχειρήσεων. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να ασκήσουμε πολύ μεγαλύτερη πίεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι όταν εξετάζουμε τις μελέτες αντικτύπου στην Επιτροπή ΙΜΚΟ, ε, θεωρούμε ότι είναι καλά τα αποτελέσματα, αλλά βασιζόμαστε στην εξή υπόθεση ότι από νομοθετική πλευρά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει να προβλέπεται κάποιο είδους εξαίρεση, δηλαδή αυτόματα ενσωματώνται μία εξαίρεση μέσα στην νομοθετική διάταξη. Ε, και δεν μπορούν να είναι εξαίρεση και όχι ο κανόνα, μικρομεσαίε επιχειρήσει. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να νομοθετούμε έτσι. σω θα μπορούσαμε να το εξετάσουμε αυτό το θέμα από κοινού. Αυτή είναι, αυτή είναι η πρώτη παρατήρηση. Δεύτερη παρατήρηση. Όπως είπατε κι εσείς, απέρχεστε από μια ιδιαίτερα επιτυχημένη προεδρία με μεγάλα επιτεύγματα. Ποιο είναι το μήνυμά σας ε, προς το Κοινοβούλιο. Σε τι θα έπρεπε να εστιάσουμε τις προσπάθειές μας εδώ στην Επιτροπή ΙΜΚΟ για τον επόμενο χρόνο. Μήπως θα είχατε κάποιο μήνυμα να περάσετε στην Επιτροπή μας. So, Απάντηση. Η ενδιάμεση αναθεώρηση της πράξης για τις μικρές επιχειρήσεις είχε μεταξύ άλλων το στόχο του να προσδιορίσουμε, να όριοθετήσουμε αυτό το πρόβλημα και να το εντάξουμε σε ένα γενικότερο πλαίσιο. Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας συνειδητοποίησα ότι χρειάζεται ορισμένες φορές να επαναλαμβάνουμε κάτι παρά τα επιτεύγματά μας, γιατί έτσι εγγράφεται το σημείο στην ημερήσια διάταξη εισαγωγικά. Δεύτερον, αυτά που είπατε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έχουμε, αυτές, ε, έχουμε την ευφυή νομοθεσία, έτσι την αποκαλούμε, με όλες αυτές τις αρχές που προανέφερα. Είναι πάρα πολύ σημαντικές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, και θα έλεγα ότι στην, η καθημερινή ζωή, αν θέλετε, η καθημερινή δουλειά των εθνικών αρχών ε, είναι πάρα πολύ δύσκολη διότι υπάρχουν κάποιες αρχές που πρέπει εμείς να εφαρμόζουμε σε καθημερινή βάση. Ξέρετε ότι στα Υπουργικά Συμβούλια έχουμε πολύ άριθμα προβλήματα και αυτό σημαίνει ότι διαρκώς πρέπει να έχουμε κατά νου αυτές τις ε, συμπεφωνημένες αρχές και να τις εφαρμόζουμε ορθά. Οπότε και η κυβέρνηση και τα κοινοβούλια ορισμένες φορές ε, πέρα από την ε, θέσπιση, την έγκριση νέων νομοσχεδίων έχουν πολύ καθημερινή δουλειά και δεν ενθουσιάζονται όταν καλούνται να εφαρμόσουν ένα κανονισμό που ρυθμίζει τον τρόπο με τον οποίο εργάζονται. Η ίδια η κατηγορία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων παρουσιάζει ιδιαιτερότητες. με του συναδέλφου μου πρέπει να συζητήσω και να πούμε ότι στην ΤΑΔΕ και στη ΔΙΝΑ χώρα 90% ξέρω, των επιχειρήσεων είναι μικρομεσαίες και να κινηθούμε αναλόγως. Οπότε αν εκπονήσουμε έναν ειδικό κανονισμό για το 99% ή το 90% κάποιου πράγματος ε, προκειμένου των επιχειρήσεων αντιλαμβάνεστε πόσο μεγάλο ειδικό βάρο έχει αυτή η κατηγορία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ως προς την ε, απλούστευση του κανονισμού για τα λογιστικά πρότυπα για τις μικρές οικονομικές οντότητες, έτσι, ονομάζονται οι μικρές επιχειρήσεις γιατί δημιουργήθηκε μια νέα κατηγορία που ουσιαστικά δεν υπάρχει, αλλά πρόκειται για εξαιρετικά μικρές επιχειρήσεις, κάτω από 10 εργαζομένους, και τα λοιπά, ε, πρέπει να του επιφυλάξουμε ειδική μεταχείριση. Μα τι είδους ειδική μεταχείριση χρειάζονται. Αυτό είναι το θέμα. Ε, ποτέ δεν ε, συνάντησα κυβερνητικό εκπρόσωπο που να πει όχι εμείς είμαστε κατά. Όλοι λατρεύουν τις μικρές ε, και μεσαίες επιχειρήσεις. Ε, πώς πρέπει όμως να τις μεταχειριζόμαστε. Αυτό είναι το θέμα. Πρέπει να είναι χρήσιμη η υποστήριξη που τους προσφέρουμε και να προσέχουμε όταν δημιουργούμε τέτοιες ε, ε, εξαιρέσεις. Όλε οι αρχέ ε, που διέπουν την νομοθεσία περί μικρομεσαίων επιχειρήσεων, παραλαμβάνω, πρέπει να εφαρμόζονται σε καθημερινή βάση. Δεν είναι εύκολη δουλειά, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει. Υπάρχουν δύο άλλα σημεία που θα μπορούσα να σχολιάσω. Μετά την ε, Ουγγρική Προεδρία, τέλος πάντων μας έχουν μείνει δέκα μέρες, Θεωρώ ότι καλό θα ήταν να επιτευχθεί μια ε, ταχεία συμφωνία για το δίπλωμα Ευρεστεχνίας, γιατί κάναμε εμεί αυτή τη σύσκεψη, αλλά ε, προφανώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η αρμόδια επιτροπή πρέπει να ε, ασχοληθούν με το θέμα. Τώρα η Ευρωπαϊκή Εταιρεία. Φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντικό το ζήτημα και εργαστήκαμε σκληρά. Υπάρχουν κάποια σημάδια που δείχνουν ότι πλησιάζουμε σε μία συμβαστική λύση. Ε, πάντως είναι ραγδαίες οι εξελίξεις, αλλάζουν τα δεδομένα καθημερινά. Ενδεχομένως ε, εδώ θα μπορούσαμε να επιφέρουμε βελτιώσεις σε αυτό το τομέα της Ευρωπαϊκής Εταιρείας ε, με την αρρωγή του Κοινοβουλίου. Θα ενθαρρύνω να κάνετε οποιοδήποτε βήμα ενισχύει την Ευρώπη και ε, ε, υποβοηθά τις επιχειρήσεις ώστε να γίνουν πιο ανταγωνιστικές και να έχουν πρόσβαση στην αγορά, στη χρηματοδότηση και ε, οτιδήποτε μπορείτε να κάνετε για να καταργηθεί το γραφειοκρατικό άχθος θα είναι πρόσφορο. Θέλω να σας υπενθυμίσω και κάτι άλλο ότι τώρα δεν είναι δυνατόν να οικοδομήσουμε ένα τεράστιο πακέτο για να τονώσουμε μόνο και μόνο με αυτό την οικονομία. Αυτό που χρειάζεται να κάνουμε είναι να μειώσουμε, να περιστήλουμε αυτό το γραφειοκρατικό άκθος τόσο ώστε να είναι πιο ελεύθερες και πιο δραστήριες οι επιχειρήσεις. Δυστυχώς δεν είναι η κατάλληλη στιγμή τώρα να ε, φτιάξουμε ένα τεράστιο ογκώδες πακέτο στήριξης, τόνωσης της οικονομίας. Λιγότερη γραφειοκρατία, ε, ε, ενισχυμένη εσωτερική αγορά και καλύτερη πρόσβαση στην καινοτομία και στις νέες τεχνολογίες. Αυτές είναι οι σύμβουλές μου, Πρόεδρος. Σας ευχαριστούμε και πάλι που ήρθατε σήμερα. Με αυτή την ιδιότητα τελευταία φορά έρχεστε στην Επιτροπή, αλλά ελπίζω να παραμείνουμε σε επαφή διότι είστε κι εσείς ε, θειασό της, ε, της εσωτερικής αγοράς, είστε ευπρόσδεκτος, ε, γιατί είναι πολυδιάστατο το θέμα, μην ξεχνάμε και την κοινωνική διάσταση του ζητήματος της εσωτερικής αγοράς. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία για το τέλος της Προεδρίας σας. Ελπίζουμε να καταλήξετε συμφωνία για το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, γιατί είναι ιδιαίτερα σημαίνο το ζήτημα και ε, ευελπιστούμε ότι θα συνεχίσετε να διαδραματίζετε ρόλο στην περιφέρεια, αν θέλετε, του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας, γιατί το αναζωογονήσατε με κάποιο τρόπο μέσα από την Προεδρία σας, του δώσατε νέα ζωή. Σας ευχαριστούμε λοιπόν ε, και σας χειροκροτήσουμε. Καλή επιτυχία για το υπόλοιπο της Προεδρίας σας. Ε, σας δίνω στα Ουγγρικά ε, την έκθεση της επίσκεψής μας στη Βουδαπέστη. Υπάρχουν και φωτογραφίες, έτσι, για σουβενίρ σας το δίνω. Λοιπόν, τώρα θα κάνουμε ένα διάλειμμα πέντε λεπτών. Ε, να σας ε, πω ότι θα έχουμε μία ακρόαση έχει ετοιμαστεί η αίθουσα για μια κρόση. Έτσι λοιπόν, να κάνουν λίγο υπομονή οι συνάδελφοι και να καθίσουν εκεί που καθόνται συνήθω για την ακρόαση. Κατόπιν θα εγκρίνουμε το πακέτο τη δεσμή μέτρων ε, της οδηγίας για τους καταναλωτές και θα συνεχίσουμε με την ακρόαση. Uh, uh, Κυρίες και κύριοι, καθίστε παρακαλώ. Καλώς ορίσατε όλοι. Θέλω να καλωσορίσω όλους όσους ήρθαν για την ακρόση, για τα εξαφρονισμένα τελωνία και την εσωτερική αγορά. Θέλω να καλωσορίσω όλους τους ομιλητές θα ξεκινήσουμε κάπως καθυστερημένα γιατί η Επιτροπή έχει ένα σημαντικό έργο να ελοποιήσει πριν ξεκινήσουμε την ακρόαση και έπρεπε να το συμπεριλάβουμε εδώ για λόγους χρονοδιαγράμματος. Πρέπει να εγκρίνουμε την τελική συμφωνία που ε, σημειώθηκε μεταξύ συζητητή και όδων συγητών με το Συμβούλιο των Υπουργών ε, στην ε, οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών. Και αν συμφωνείτε, θα πρότεινα σε μπλοκ ε, να δούμε το κείμενο του Συμβουλίου. Έχουμε ένα ενοποιημένο κείμενο και επίσης να ψηφίσουμε μάλλον ε, να λάβουμε υπόψη της δήλωσης Προεδρίας ε, για τους πίνακες αντιστοιχίας και τη δική μας δήλωση για τους πίνακες αντιστοιχίας. Αυτά είναι τα δύο τμήματα της συμφωνίας, την οποία καταλήξαμε για τους πίνακες αντιστοιχία. Έτσι λοιπόν, αυτό αφορά τα μέλη της Επιτροπής ε, για την εσωτερική αγορά. Ξέρω ότι είναι μέλη και άλλες επιτροπές εδώ, να μας το πείτε εκ των προτέρων. Θέλω να καλωσορίσω ε, και την κυρία ε, που είναι η την κυρία που είναι η συγγήτρια της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων. Έχουμε και κάποιες σύντομες ε, δηλώσεις από τον κύριο Χάνς Πίτερς Μέιος, ο οποίος έχει αναλάβει το ρόλο του για για τη ο κύριο ΣΒΑΠ, και από την κυρία Γκέπαρτ. Και η κυρία Γόλης θέλει να πει κάτι, μάλιστα, δεν θέλει. Ε, επομένως, να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Αν έχετε τις κάρτες σας, θα υλοποιήσουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία για ε, να έχουμε και το αρχείο. Λοιπόν, ας ακούσουμε λοιπόν τον ε, κύριο Χανς Πίτερ Μάιερ που έχει αναλάβει το ρόλο του συγκητή. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, εκπροσωπώ τον Ανδρέα Σφάμπ, ο οποίος χθες και σήμερα λόγω ενός προγραμματισμένου ταξιδιού απουσιάζει, οπότε σας ευχαριστώ των προτέρων για την ε, διάθεση συνεργασία ε, που έχετε επιδείξει. Να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο, τη Γραμματεία και βεβαίω την Προεδρία του Συμβουλίου και την Κομισιόν. Έχουμε συνολικά ε, επιτύχει κάποιες υποχρέωσεις πληροφόρησης. Καταφέραμε στο κεφάλαιο 5 να επιτύχουμε σημαντικά σημεία όπως τα predict boxes. Επίσης στο κεφάλαιο 4 όπου έχουμε νέα και θετικά στοιχεία που γίνονται νομικά δεσμευτικά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Επίσης το κύριο μέρος της οδηγίας στο κεφάλαιο 3 για συμβάσεις ε, εξ αποστάσεως ε, και στην πόρτα του σπιτιού καταφέραμε να δημιουργήσουμε μεγάλη ασφάλεια για τον καταναλωτή και για τις μικρές βιοτεχνίες. Για το θέμα του κόστους ε, τα είπαμε και χτες, θεωρώ πως υπάρχει μια ξεκάθαρη ρύθμιση στο κείμενο και στην εφαρμογή οπωσδήποτε η Κομισιόν θα φροντίσει να υπάρχει σαφήνεια. Οπωσδήποτε το Κοινοβούλιο θα επιθυμούσε κάποια πράγματα παραπάνω σε ορισμένα σημεία. Θεωρώ όμως πως ένας, αυτός ο συμβιβασμός ε, είναι ε, αποδεκτός από όλους και όπως ξέρετε συμβιβασμός σημαίνει αμοιβές υποχωρήσεις. Ήτανε σε αυτή την περίπτωση θετικό το ότι όλοι ήταν υπέρ της συνένεσης και του συμβιβασμού. Γι' αυτό μπορέσαμε να βελτιώσουμε το κείμενο το αρχικό της Κομισιόν και του Συμβουλίου. Αγαπητοί συνάδελφοι, πεπισμένος πως και με μια δεύτερη ανάγνωση δεν θα είχαμε καλύτερο αποτέλεσμα μπορούμε ως ομάδα του ΕΛΚ και ως συγητής να συμφωνήσουμε με αυτό το κείμενο και σας παρακαλώ να το εγκρίνετε. Η κυρία Γκέπχαρτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και εγώ όλους συμμετέχοντες για τη δύσκολη δουλειά. Υπήρχαν μεγάλες διαφωνίες όπως ξέρετε αλλά θεωρώ πως το αποτέλεσμα το οποίο επιτύχαμε είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο μπορούμε να δεχτούμε δεν είχαμε συμβασμούς που δεν μπορεί να δεχτεί κανείς. Αυτό το οποίο βρίσκω πάρα πολύ σημαντικό είναι το κομμάτι για την υποχρέωση πληροφόρησης έτσι ώστε ο πολίτης να ξέρει ε, σε τι δεσμεύεται όταν αγοράζει κάτι. Αυτό επιτύχαμε και νομίζω πως έχουμε επιτύχει μεγάλη πρόοδο. Πάρα πολύ θετικό είναι πως ε, συμπεριληφθεί και ο ψηφιακός ε, τομέας που αρχικά δεν ε, προβλεπόταν και ξεκαθαρίσαμε πως στις αγορές στο ίντερνετ καταφέραμε να έχουμε μια λύση η οποία σημαίνει πως δεν θα πρέπει να έχουν γίνει επιλογές εκ των προτέρων και θα πρέπει βεβαίως η συνολική τιμή να αναφέρεται πριν οριστικοποιηθεί η αγορά, οπότε έχουμε μια νομική ασφάλεια για τον καταναλωτή. Γι' αυτό μπορώ σήμερα πράγματι να συστήσω στην ομάδα μου να συμφωνήσει με αυτό τον θετικό συμβιβασμό. Uh, um, Ευχαριστώ. Υπάρχουν και άλλοι σκιώδεις εδώ. Θα ήθελα, παρακαλώ να είστε σύντομοι. Κύριος Ροσφόρ, καταρχήν, ευχαριστώ Πρόεδρε, πολύ γρήγορα. Η ομάδα μου των φιλελευθερών επίσης υποστηρίζει αυτό κείμενο και θα το υποστηρίξουμε για δύο κυρίους λόγους. Πρώτος λόγος ότι δεν αποτελεί απλώ μια ισορροπία μεταξύ πολιτικών ομάδων ή μεταξύ οργάνων, κάτι που είναι σημαντικό, αλλά αποτελεί και ισορροπία μεταξύ συμφερόντων των καταναλωτών και των συμφερόντων των επιχειρήσεων και με τον τρόπο αυτό συνεισφέρει τα μάλλα στην ενιαία αγορά, στην ιστορική αγορά. Δεύτερον, είναι θεμελιώδες για μας ε, και πρέπει να χαιρόμαστε ότι χάρη σε γενική δουλειά έχουμε μια συμφωνία των πολιτικών ομάδων και αποτελεί ένα σαφέ μήνυμα για την κατεύθυνση την οποία θέλουμε να ακολουθήσουμε για την καθημερινή ζωή των καταναλωτών και των επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Um, Ευχαριστώ. Νομίζω ότι δεν ζητά άλλος ε, το λόγο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχουμε εδώ ε, εκπροσώπου του Συμβουλίου και τη Κομισιόν. σω θα καλέσετε την εκπρόσωπο του Συμβουλίου και την ε, εκπρόσωπο τη Κομισιόν. Παρακαλώ, Εκπρόσωπο του Συμβουλίου καταρχήν. Ευχαριστώ. Χαίρομαι πάρα πολύ που περιβρίσκομαι εδώ. Και όπως ε, είπε και ο Υπουργός μου πριν μισή ώρα, στα πλαίσια της ε, συζήτησης ε, για το ενιαίο σύστημα διπλωμάτων βρεσιτεχνίας, ε, όπως και εκείνο είναι σημαντικό και αυτό εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα σα υπενθυμίσω ότι είπα τον Ιανουάριο, όταν πρώτα εκπροσώπησα, όταν τότε εκπροσώπησα την Ουγγρική Προεδρία στην Επιτροπή σα για πρώτη φορά, ότι αυτό αποτελεί κύρια προτεραιότητα για την Ουγγρική Προεδρία, δηλαδή να έχουμε μία Προεδρία φιλική προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και τώρα φτάσαμε στον Ιούνιο και μπορούμε να πούμε ότι πετύχαμε μια συμφωνία για αυτό το πάρα πολύ σημαντικό φάκελο. Ήμασταν επιτυχείς ε, στο να διεξάγουμε μία φιλική προς το Κοινοβούλιο Προεδρία για τους λόγους που αναφέρθηκαν. Πιστεύω ότι η συμφωνία αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική και για τις επιχειρήσεις και για τους καταναλωτές. Αποτελεί μεγάλο συμβιβασμό και σας ευχαριστούμε όλους όσους συμμετείχατε στην επιτευξή του. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και η κυρία Μίσου, μέρος της Κομισιόν. Good morning to Καλημέρα σε όλους. Θα ήθελα μόνο να προσθέσω πως είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη και καλωσορίζω όλες αυτές τις εντατικές συσκέψεις που είχαμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όλοι ήταν αφοσιωμένοι, τελεσφόριζαν οι συζητήσεις και οδηγηθήκαμε στο σημερινό αποτέλεσμα. Οι υπηρεσίε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κρίνουν επίσης πως το σημερινό αποτέλεσμα είναι ιδιαίτερα εξισορροπημένο και για τους καταναλωτές και για τους εμπόρους. Σας ευχαριστούμε για αυτή την τόσο επικοδομητική και αγαστή συνεργασία. Πρόεδρος, θα ήθελα με την ιδιότητα του Πρόεδρου να ευχαριστήσω όλους τους εισηγητές και όλους τους εισηγητές ε, ε, της Υπηρεσίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Κοινοβουλίου που εργάστηκαν σκληρά και τώρα θα ψηφίσουμε για αυτά τα τρία σημεία ομού με ηλεκτρονική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία. αντίστροφα την κάρτα σας αν δεν δουλεύει. Ψήφισαν όλοι. Υπάρχει κάποιος που δεν έχει ψηφίσει. Λείπει μία ηλεκτρονική κάρτα. Πατήστε το κουμπί. Χάσαμε μία ψήφο πέρα, πέρα ψηφοφορίας. 28 ψήφοι υπέρ καμία κατά, τρεις αποχές. Συγχαρητήρια για τους συζητητές και σκιώδους συζητητέ. Uh, τα κείμενα αυτά θα τα προσυπογράψουν οι εκπρόσωποι των πολιτικών ομάδων και θα περάσουν από την Ολομέλεια την ερχόμενη εβδομάδα. Θα περάσουμε τώρα στην ακρόαση. Ελπίζω οι βουλευτέ να παραμείνουν. Αν πρέπει να αποχωρήσετε, παρακαλώ διακριτικά. Γλιστρήστε έξω από την αίθουσα γιατί έχουμε καθυστερήσει λίγο. Ελπίζουμε οι προσκεκλημένοι μα να δείξουν κατανόηση. Ε, θα κάνουμε ένα δίλεπτο διάλειμμα για να βρουν όλοι τις θέσεις τους και αρχίζουμε αυτές αμέσως. Uh, um, λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Οπότε, αν θέλετε να συζητήσετε, παρακαλώ βγείτε εκτός ε, της αιθούσης. Λοιπόν, οι βουλευτές εκεί στα ορεινά να έρθουν ε, λίγο πιο μπροστά. Για να γίνει λίγος χώρος για τους επισκέπτες. Um, uh, λοιπόν, καλώς ήρθατε και πάλι στην ακρόαση. Καλώς ορίζω μας παρακολουθούν και από το διαδίκτυο. Ακούσατε γιατί καθυστερήσαμε, αλλά σας καλωσορίζουμε και online. Λοιπόν, να σας πενθυμίσω Προς όσον αφορά τη μετάδοση στο διαδίκτυο, όταν πατάτε το μικρόφωνο, αυτομάτως η κάμερα θα γυρίζει επάνω σας. Καλώς ορίζω επίσης ε, τον εισηγητή μας ε, για την έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας, ε, τον κύριο Ματία Σελτίνη, ο οποίος θα κάνει και κάποια σχόλια στο τέλος και ευχαριστούμε και την ομάδα του μαζί με τους κοιόδης εισηγητές και βεβαίως ε, πρόκειται για μέρος των ιδεών που θα πάνε στην έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας για τα εξυγχρονισμένα τελωνία. Τα τελωνία είναι σημαντική ευθύνη της ε, Επιτροπής μας και βεβαίως χαιρόμαστε που ακούμε τους ειδικού ε, για τα ζητήματα τα οποία μας απασχολούν. Ο χρόνος πιέζει, οπότε θα δώσω στον κάθε ένα ομιλητή 5 λεπτά. Πρέπει να έχετε νομίζω σε ένα πακέτο όλες ε, τα εντυπωσιακά βιογραφικά τους. Ε, είχατε μια ευκαιρία να τα διαβάσετε. Λοιπόν, αυτό το οποίο προτείνω, δεδομένου του ότι ξεκινάμε λίγο αργά, είναι να μιλήσουμε πρώτα απ' όλα στην πρώτη συνεδρία για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Μετά θα ακούσουμε ερωτήσεις και απαντήσεις και μετά οι συνεδρίες 2 και 3 να τις συνδυάσουμε για να ακούσουμε τους ομιλητές και να κάνουμε στο τέλος ε, μαζί να έχουμε ερωτοαποκρίσεις γιατί ούτως ή άλλως νομίζω πως οι ιδέες αυτών των δύο τμήματων μπορούν να συνδυαστούν και θα πρέπει να ολοκληρώσουμε 12.30 ακριβώς. Αυτά ως χρονοδιάγραμμα. Περνάμε τώρα στο τμήμα ενίσχυση τη ανταγωνιστικότητα, όπου θα έχουμε τέσσερι ομιλητέ. Ο κύριο Μύροσλαβ Ζιελίνσκι, πρώτο, ο διευθυντή ε, της ε, Τελωνιακή πολιτικής νομοθεσίας δασμών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί γνωρίζετε τη επιτροπή μα. Μετά καλωσορίζω την κυρία Σούζαν Ένιε, η οποία είναι υποδιευθυντής ε, συμμόρφωση με νομοθεσία και διευκόνιση στον ε, Παγκόσμιο Οργανισμό Τελωνίων και παίζει σημαντικό ρόλο στα θέματα αυτά. Μετά από την Πολωνία ο Χιμπερτ Γιάντρικ, ο οποίος εργάζεται για την Pricewaterhouse και είναι πρόεδρος της ε, σχετικής ε, επιτροπής για το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Τελωνίων, δηλαδή εντός της εταιρείας, και κάποιος ο οποίος ασχολείται κάθε μέρα με αυτά τα θέματα, ο Keith Bond, ο οποίος είναι υπεύθυνο τελωνιακών θεμάτων για τη UPS ε, στην Ευρώπη και οπωσδήποτε θα μας πει πόσες συναλλαγές περνάνε μέσω της UPS κάθε μέρα για να έχετε έτσι, μια ιδέα της κλίμακας της ε, δουλειάς του και χαιρόμαστε που έχουμε σήμερα την πρακτική του εμπειρία. Πρώτα απ' όλα λοιπόν ο κύριος Ζελίνσκι για πέντε λεπτά. Mr. Chairman. Πρόεδρε, Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίε και κύριοι. Είναι προνομιό μου να υποβάλω την πρώτη παρουσίαση και θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο σε πέντε λεπτά και θα επικεντρωθώ μόνο στην κατάσταση του ξεχρονισμένου τελωνικού κώδικα και τη σχετική αναδιατύπωση. Δεν θα ασχοληθώ με άλλα θέματα, αλλά φυσικά τα τελωνία δεν συνιστάνται μόνο στον ξεχρονισμένο τελωνιακό κώδικα. Έχω και κάποιες διαφάνειες. Μπορούμε να τις δούμε στην οθόνη. sorry. a bit behind with your Ναι, συγγνώμη, έχουμε καθυστερήσει κάπως με τις διαφάνειες σήμερα, αλλά αν θέλετε ξεκινήσετε και θα εμφανιστούν. Μάλιστα, σας ευχαριστώ. Μιλάμε για την διατύπωση του εξυγχρονισμένου τελωνιακού κώδικα. Εδώ έχουμε μια διαφορά γιατί δεν θέλουμε να ξανανοίξουμε τη συζήτηση. Υπάρχουν τρεις κύριοι στόχοι της αναδιατύπωσης του ξεχρονισμένου τελωνιακού κώδικα, το MCC, καταρχήν ε, για πολλούς ε, λόγους επειδή υπάρχει αναγκαιότητα να αναπτύξουμε συστήματα ε, πληροφορικής, έχουμε την ε, αναστολή. Επίσης, έχουμε το θέμα της ευθυγράμμισης ε, του εξυγχρονισμένου του ελληνικού κώδικα με τη συνθήκη της Λισαβόνας και όταν εργαζόμαστε για τις εκτελεστικές πράξεις πρέπει ε, να έχουμε μία διαίρεση μεταξύ κατεξουσιοδότηση πράξεων και εκτελεστικών πράξεων ε, στον MCC. Και έχουμε και κάποιες διορθώσεις ε, που προέκυψαν από το business parcel modeling και από την ανάπτυξη και άλλης σχετικής τελειωνιακής νομοθεσίας. Κατόπιν, τι κάνουμε, προσπαθούμε να περιορίσουμε τις τροποποιήσεις Προσπαθούμε να παραμείνουμε πιστοί στην αρχική πρόθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Κομισιόν όταν ψηφίστηκε το 2008 MCC. Κατόπιν ε, έχουμε ένα φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα. Ξέρουμε ότι χρειάζεται ο ξεχρονισμένο ελληνικό κώδικα για την επιχειρηματική κοινότητα και για την Ευρώπη. Έτσι λοιπόν ε, αναπτύξαμε σε ξεκάθαρα κριτήρια για τις διορθώσεις, καταρχήν αλλαγέ στη διατύπωση. Και αυτό είναι πάρα πολύ απλό. Πρέπει να τροποποιήσουμε εκεί όπου λέμε κοινότητα σε Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκή Κοινότητα σε Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε κάποιες αλλαγές που προκύπτουν από τις διάφορε αλλαγέ στην νομοθεσία. Στη συνέχεια πρέπει να λάβουμε υπόψη το business process modeling. Ε, όταν υιοθετήθηκε ή συζητήθηκε ο MCC πριν από πολλά χρόνια, το business process modeling δεν είχε αναπτυχθεί τόσο καλά. Τώρα έχουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο και ταυτόχρονα όταν καταρτίζουμε τις νομικές διατάξεις βλέπουμε τη διαδικασία και κατόπιν μπορούμε να αποφύγουμε τα λάθη και τις εκπλήξεις. Και φυσικά πρέπει να λάβουμε και υπόψη τα αποτελέσματα αυτής της εργασίας. Κατόπιν, πώς έχει η κατάσταση με το χρονοδιάγραμμα. Είχαμε την επιστολή της 19 η Μαΐου στον πρόεδρο της Επιτροπής ΕΙΜΚΟ και στην Ουγγρική Προεδρία. Στην επιστολή αυτή θέλαμε να εξηγήσουμε, μάλλον θέλαμε να ζητήσουμε πολιτική υποστηρίξη και να έχουμε μια κοινή κατανόηση των αλλαγών. Κατόπιν απευθυνθήκαμε στην Ουγγρική Προεδρία και στις μελλοντικές Πολωνική και Δανική Προεδρίες και Είχαμε μια σειρά ερωτημάτων ε, από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το πολύ σημαντικό θέμα είναι το θέμα της αναδιατύπωσης, recast. Όπως σας είπα, δεν θέλουμε να επαναλάβουμε τη συζήτηση. Και κατόπιν θέλουμε να ολοκληρώσουμε το προπερισκευαστικό έργο για το Business Process Modeling και για τον ε, MCCAP, για τις εφαρμοστικές διατάξεις ε, δηλαδή Το ξεχρονισμένο τελωνιακό κώδικα και κατόπιν ε, πρέπει να λύσουμε μια σειρά θεμάτων. Συζητούμε με την κοινότητα των εμπόρων με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Τι κάνουμε τώρα, κάτι πολύ πολύπλοκο, γιατί συνεχίζουμε να εξετάζουμε τις εφαρμοστικές διατάξεις αλλά ε, προσπαθούμε να διαφοροποιήσουμε και τις διάφορες αρμοδιότητες ε, σε εκτελεστικές πράξεις και σε κατεξουσιοδότηση πράξεις. Έτσι λοιπόν έχουμε διπλό όγκο εργασίας. Θα ήθελα να σας πω ότι είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε δυνατότητα κύψει. Είμαστε έτοιμοι για τις συζητήσεις, θα κρατούμε ενήμερο το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φυσικά. Εξεκολουθούμε να έχουμε την πρόθεση να υιοθετηθεί η πρόταση από το Σώμα των Επιτρόπων ε, μέχρι τα τέλη του έτους, αλλά θέλουμε να αποφύγουμε την εξή κατάσταση. Κομισιόν να στείλει την πρόταση το Δεκέμβριο ή στις αρχές Ιανουαρίου και κατόπιν ε, όλοι να εκπλαγούν. Έτσι λοιπόν ε, πραγματικά θέλουμε να έχουμε μια πολύ καλή επικοινωνία. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Ζελίσκη που μας ε, παρουσιάσατε το πρόγραμμά σας ε, και ο κύριος ε, Σαλβίνη θα μας προετοιμάσει και φυσικά θα μας δώσει και την κατάλληλη ενημέρωση για το θέμα αυτό. Στο πακέτο έχετε και τις διαφάνειες του κυρίου Ζαλίνσκι. Μπορείτε να τη βρείτε φυσικά και στην ιστοσελίδα μας μετά την συνεδρίαση. Κατόπιν θα περάσουμε στην κυρία Ιγνέρ από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τελωνίων θα εμφανιστεί στην οθόνη και θα εμφανιστεί και δική σας δέσμη διαφανειών. Δυστυχώς έχουμε καθυστερήσει. Ευχαριστώ σας δώσω το λόγο. Thank you very much for the invitation. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση σήμερα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τελωνίων χαίρεται που συμμετάσχει στη σημερινή ακρόαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μου ζητήθηκε να εξηγήσω ότι κάνουμε σφαιρικά για τον εξυγχρονισμό των τελωνίων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τελωνιακών υπηρεσιών. Να μιλήσουμε επίσης για τα μέλη μας και για τις εμπορικές συναλλαγές. Είμαστε ένας διεθνής οργανισμός και όταν συζητούμε για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τελωνίων αναφερόμαστε στα 177 μέλη μεταξύ των οποίων και η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα πιο δραστήρια μέλη φυσικά είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη της Ένωσης. Ποια είναι η αποστολή μας, ε, νομίζω είστε εξοικειωμένοι με αυτό, γιατί ποιοι είναι οι στόχοι που επιδιώκει ο Διεθνής Οργανισμός ε, Τελωνίων. Δεν ε, συμμορφώνονται αυτοί οι στόχοι απαραίτητα, δεν ταυτίζονται με τους στόχους Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τη δική μας πλευρά, αυτό που επιδιώκουμε είναι τα 177 μέλη μας να έχουν τη θέση που τους πρέπει στον οργανισμό μας. Ε, η πλειοψηφία αυτών των μελών είναι αναπτυσσόμενες χώρες και αντιμετωπίζουν προκλήσεις διαφορετικές από αυτές που βιώνουμε εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα δείτε ότι ένας από τους στόχους εξακολουθεί να είναι η συλλογή εισοδήματο. Ε, είναι ο πρωταρχικός στόχος των αναπτυσσόμενων χωρών, αλλά ξεκάθαρα Όλες οι δραστηριότητες μας ε, στοχεύουν στην ε, επίρρωση της ανταγωνιστικότητας και αρρωγή προς τα μέλη μας ε, για να χρησιμοποιήσουν τα νέα εργαλεία και το εξυγχρονισμό τελωνιακό σύστημα, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, καθώς και το αναθεωρημένο πρωτόκολλο του Κιώτο μεριμνούμε ώστε να εφαρμόζεται ένα απλουστευμένο, εξυγχρονισμένο τελωνιακό ε, καθεστώς με το ενίο επιχειρησιακό μοντέλο, με τη μονοαπευθυντική θηρίδα και ούτω καθεξής. Ε, θα ρίνουμε την τελωνιακή συνεργασία, οικοδομούμε την εγχώρια δυναμικότητα σε πολλά από τα μέλη μας, καθώς και σε κράτη-μέλη της Ένωσης ε, και προαγάγουμε ε, τις ε, συνεργατικές ε, σχέσεις ανάμεσα στα τελωνία και τους εμπορικούς φορείς. Θα μπορούσαμε να περάσουμε στην επόμενη διαφάνεια. Οι βασικές προκλήσεις, τις οποίες και θα σχολιάσω εν συντομία, διότι συνιστούν κοινέ προκλήσεις και για σας, έγκυται στους βασικούς τομείς που βλέπετε στη διαφάνεια και είπαμε ότι ορισμένοι στόχοι ταυτίζονται με τους στόχους Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι βασικές δραστηριότητές μας λοιπόν σκοπεύουν στην υπεράσπιση των συμφερόντων των μελών μας ε, για τη διευκόλυνση των εμπορικών συναλλαγών, νέες τεχνολογίες, συνεργασία με τους εμπορικούς φορείς κτλ. Επίσης, έχουμε στενή συνεργασία ε, με την ε, ομάδα επαφής για το εμπόριο της Γενικής ε, Διεύθυνσης Ταξούντ και εκπροσωπούνται εδώ στη σημερινή ακρόαση εξάλλου. Συμβάλλουν λοιπόν στις εργασίες μας διότι εκφράζουν τις ανησυχίες που έχουν οι εμπορικοί φορείς ούτως ώστε όταν εκπονούνται τα νέα μέτρα να είναι δυνατόν να εφαρμοστούν διότι πρέπει να καλύπτονται οι ανησυχίες και των τελωνιακών αρχών και των εμπορικών φορέων που καλούνται να εφαρμόσουν τον εξυγχρονισμένο τελωνιακό κώδικα. Είπαμε λοιπόν ότι με τον εξυγχρονισμένο τελωνιακό κώδικα ε, ορισμένοι από τους στόχους μας ταυτίζονται με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης Έχουμε στενή συνεργασία με τα κράτη-μέλη της Ένωσης ως εκ τούτου και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όλος ιδιαίτερος δε με τη Γενική Διεύθυνση Ταξούντ. Μπορείτε να πάτε στην μεθ επόμενη διαφάνεια. Δεν έχω πολύ χρόνο στη διάθεσή μου, αλλά θα ήθελα να σας πω πως ε, το 2008 εγκρίναμε έναν οδικό χάρτη για τα τελωνία ε, τελωνία του 21ου αιώνα. Αυτό είναι ο τίτλος. Γνωρίζετε ποια είναι η μελλοντική στρατηγική των τελωνίων, αναμφίβολα. Εκπονήσαμε αυτό τον οδικό χάρτη σχεδόν ταυτόχρονα με τον εξυγχρονισμένο τελωνιακό κώδικα. Ήταν κάτι απαραίτητο, ούτω ώστε τα τελωνία να εφαρμόσουν τη νέα νομοθεσία μέσα από νέες ε, μεθόδους ε, εργασίας. Ε, έχουμε πρότυπα, πρωτόκολλα, κατευθυντήριες γραμμές, διαρθρωμένες ανταλλαγές απόψεων, συστήματα διαχείρισης κινδύνου, θέματα ασφαλείας κτλ. Ε, ξέρετε, είναι, ήταν πληρέστερη η παρουσίασή μου. Θα σταματήσω εδώ γιατί δεν θέλω να υπερβώ το χρόνο μου. Πάντω, κοιτάξτε τι διαφάνειε ε, και είμαι στη διάθεσή σα ε, για ερωτήσει και ίσω τα θέματα ασφαλεία να τα σχολιάσουν καλύτερα άλλοι ομιλητέ. Πρόεδρο, ευχαριστούμε. Έχουμε και τι διαφάνειέ σα. Είναι πολύ χρήσιμε αυτέ οι πληροφορίε να ακούσουμε για τα νέα εργαλεία που έχετε εκπονήσει στον Παγκόσμιο Οργανισμό Τελωνίων και μα ενδιαφέρει αυτό που είπατε για τον οδικό χάρτη Τελωνία για τον 21ο αιώνα γιατί είναι κομμάτι της δουλειάς μας. Θα περάσουμε τώρα στους επαγγελματίες του κλάδου ε, για να ακούσουμε ποια ζητήματα τους ε, απασχολούν και τι θα πρέπει να συμπεριλάβουμε στις συζητήσεις μας για τον εξυγχρονισμένο τελωνιακό κώδικα. Ο κύριος Γιάντζεστρικ, ε, δεν ξέρω αν προφέρω, παρέφθυρα το όνομά σας μάλλον, τέλος πάντων. Και μετά ο κύριος Βόγκαν. Θα με βοηθήσετε κύριε Χάνης, πώς το προφέρετε, είστε κι εσείς από την Πολωνία. Ε, ε, ε, Γιάτζικ, ε, είναι συνεταιρό στην, Κούπερ, στην παραγωγή Κούπερ στην Πολωνία και αρμόδιο για την φορολογία. Κάθε μέρα συνεργάζομαι με πολλέ εταιρείε που δραστηριοποιούνται στην εσωτερική αγορά και προσφέρω τελωνιακέ συμβουλές. Συνοψίζοντας λοιπόν, θα προσπαθήσω σύντομα να παρουσιάσω την άποψη των επιχειρήσεων για τον ε, εξυγχρονισμένο τελωνιακό κώδικα και πώς θεωρούν πως ε, μπορούν να είναι πιο ανταγωνιστικές στην εσωτερική αγορά αλλά και ευρύτερα σε παγκόσμιο επίπεδο. Πρώτα απ' όλα, ο εξυγχρονισμένος τελωνιακός κώδικας για μένα η μεγαλύτερη ανησυχία που προξενεί είναι πως δεν είναι πάρα πολύ γνωστό στις επιχειρήσεις όταν μιλάμε με, αυτός, με αυτές. Και ο λόγος γι' αυτό είναι πως ε, παρά το ότι ο κανονισμός δημοσιεύτηκε πριν από λίγα χρόνια, είναι πως δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Οπότε το σημαντικότερο κομμάτι, οι εφαρμοστικές διατάξεις ε, δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί. Οπότε, κατ' ουσίαν, δεν μπορεί να αποτελέσει βάση προγραμματισμού για τις επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή. Όσον αφορά την ε, ψηφιοποίηση του τελωνιακού συστήματος και του να υπάρχει μία και μόνη εφαρμογή για τις τελωνιακές εφαρμογές, φαίνεται πως δεν είναι ρεαλιστικό αυτή τη στιγμή, γιατί χρησιμοποιούνται διαφορετικά πληροφοριακά συστήματα π.χ. για δηλώσεις ε, τελωνιακές και ταυτόχρονα η ερμηνεία των διατάξεων από τις διαφορετικές τελωνιακές αρχές ε, επίσης ε, διαφέρει ελαφρώς από την άλλη για να πούμε και τα θετικά ή το καθεστώς του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα φαίνεται πως γίνεται όλο και πιο σημαντικό για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ε, ενιαία αγορά. Επίσης, και αυτό βασίζεται στην πρόσφατη εμπειρία μου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυξάνονται οι επιχειρήσεις που ζητούν ε, να υπαχθούν σε αυτό το καθεστώς και λαμβάνουν ε, αυτό το καθεστώς των εγκεκριμένων οικονομικών φορέων. Δυστυχώς βεβαίω αυτό από μόνο του δεν παρέχει πολλές διευκολύνσεις για όσους έχουν αυτό το καθεστώς. Και η πλειοψηφία των εταιριών που ζητούν ε, το καθεστώς αυτό του εγκεκριμένου φορέα το κάνουν γιατί ανανεώνουν τις άδειέ τους γενικώ και το κάνουν για λόγους απλοποίησης. Ε, δεν υπάρχουν δηλαδή ε, ουσιαστικά με μετρήσιμες διευκολύνσεις για τους κατόχους ε, αυτού του καθεστώτος. Συνοψίζοντας ε, και για να εφηγραμμιστούμε με το θέμα του εργαστηρίου αυτού, την ανταγωνιστικότητα, πώς να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα. Θεωρώ πως ο βασικός στόχος του κανονισμού του τελωνιακού πρέπει να ευθυγραμμίζεται με το βασικό στόχο των επιχειρήσεων, που είναι η ταχύτητα στο σύγχρονο κόσμο. Ταυτόχρονα βεβαίως η ευκολία και η ενιαία εφαρμογή ε, σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά. Και ε, έχω κάποιες σκέψεις, βεβαίως ε, αυτό είναι η φωνή των επιχειρήσεων, το τι θα ήθελαν οι επιχειρήσεις να υπάρχει στο νέο τελωνιακό περιβάλλον υιοθέτηση νομίζω εφαρμοστικών διατάξεων ε, για τον εξυγχρονισμένο τελωνιακό κώδικα νομίζω πως είναι στοιχείο κλειδί για να γνωρίζουν οι επιχειρήσεις ε, πώς θα λειτουργούν στο νέο τελωνιακό περιβάλλον. Πρέπει να έχουν λοιπόν επαρκή χρόνο για να μπορούν να προγραμματίσουν και να προσαρμοστούν οι επιχειρήσεις τους. Το κρίσιμο στοιχείο επίσης είναι το να υπάρχουν περισσότερες ευκολίες για όσους έχουν αυτό το καθεστώς. Μπορεί π.χ. να μην υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης τελωνιακού χρέους, διευκόλυνση πληρωμών και ΦΠΑ εισαγωγών και πιθανώς κάποιες άλλες διευκολύνσεις. Και τέλος, ευρύτερα, όσον αφορά τον υπόλοιπο κόσμο, σημαντικό είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει κάποια δράση για διαπραγματευτεί αμοιβαία αναγνώριση ε, του καθεστώτος αυτού του εγκεκριμένου φορέα όπως έγινε με την Νορβηγία, ε, Ελβετία και Ιαπωνία. Νομίζω λοιπόν πως όλα αυτά θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να είναι πιο ανταγωνιστικές στην ενιαία αγορά και νομίζω πως θα πρέπει όλοι να επικεντρωθούμε στο να έχουμε ε, τις ε, πιο σύγχρονες τελωνιακές ρυθμίσεις στον κόσμο. Σας ευχαριστώ. Μάλιστα, τελευταία ομιλητής τώρα, Keith Vaughan και έχουμε και τις δικές σας ε, διαφάνειες. Mr. Chairman... Πρόεδρε, κύριε. και κύριοι, το Trade Contact Group ε, είναι ένα συμβουλευτικό φορέας που δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να τη βοηθήσει μεταξύ άλλων στη σύνταξη των εφαρμοστικών διατάξεων του MCC. Αποτελείται από ε, τις κυρίες διεθνείς ενώσεις ε, που συμμετέχουν στις διάφορες τελωνικές δραστηριότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το Trade Contact Group είναι ένα φόρουμ, ε, δεν υπάρχει από μόνο του, ούτε έχει εκπροσώπους ή ε, ε θέσεις, οι 24 από τις ενώσεις που εκπροσωπούνται στην ομάδα επαφής για το εμπόριο έχουν καταλήξει σε αυτή την κοινή δήλωση. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεσμεύτηκαν στο στόχο μιας ενίας πανευρωπαϊκής τελωνιακής ένωσης. Ένα τέτοιο όραμα θα προβεί σε εξοικονομήσεις για τα κράτη-μέλη μακροπρόθεσμα και θα καταστήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση πιο ανταγωνιστική για τις επιχειρήσεις. Για να πληρωθεί το όραμα αυτό πρέπει να υπάρχει επαρκής υποστήριξη, συνεπής υποστήριξη σε όλη την Ευρώπη για τους στόχους του MCC και υποστήριξη στους απαραίτη... και διοχέτευση των απαραίτητων πόρων για να ε, δημιουργήσουμε τις διαδικασίες που θα είναι απαραίτητες για όλους τους οικονομικούς φορείς και θα έχουμε και ξεχρονισμό. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να επικεντρωθούμε σε δύο τομείς ανησυχία συγκεκριμένο στο καθεστώς του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα και στον κεντρικό εκτελονισμό το να αποκτήσει κάποιο ένα καθεστώ συγκεκριμένο οικονομικό φορέα σημαίνει ότι θεωρείται η εταιρεία ένα έμπιστο εταίρο των τελωνίων. Ε, δεν, ε, το κόστος για τις επενδύσεις και ε, ο χρόνος που εξοικονομείται είναι κάτι πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν οι εφαρμοστικές διατάξεις ε, του εξυγχρονισμένου τελωνιακού κώδικα ε, θα πρέπει να προσφέρουν ωφέλη στον εμπορευόμενο βάσει στο βαθμό συμμόρφωσης και βάση διαφάνειας. Διαφορετικά όπως έχει τώρα η κατάσταση οι εταιρείε, συγκεκριμένα μικρές και μεσές επιχειρήσεις δεν θεωρούν ότι αξίζουν να καταστούν εγκεκριμένος οικονομικός φορέας και ε, το όλο πρόγραμμα ε, και οι προσπάθειε της Ευρωπαϊκής Ένωσης στήθενται σε κινδυνό. Ο κεντρικό εκτελεισμός είναι κυρίω στοιχείο του MCC όπω θεσπίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό το μέσο θα διευκολύνει τι επιχειρήσει να υλοποιήσει τη διαδικασία του εκτελονισμού σε ένα κράτος μέλος μόνο ακόμη και αν τα πραγματικά ε, φορτία έχουν προορισμό ένα άλλο κράτος μέλος. Σήμερα οι εταιρείε έχουν να αντιμετωπίσουν 27 διαφορετικά συστήματα πληροφορικής και τελωνικές διαδικασίες και ε, το να ε, προσφέρουμε αυτή τη δυνατότητα, δηλαδή να έχουμε ένα μόνο σύστημα, ωφελεί πάρα πολύ και τέτοια ίδια τελωνία αλλά και τον καταναλωτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η σύνταξη των εφαρμοστικών διατάξεων του εξυγχρονισμένου τελωνιακού κώδικα έχει καθυστερήσει πολύ εν μέρη λόγω της τεχνικής και πολύπλοκης φύσης του έργου. Εκατοντάδες σελίδε τεχνικών διατάξεων πρέπει να εξεταστούν από του προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα λειτουργήσουν στην πράξη. Τέτοια πολύπλοκη και σημαντική νομοθεσία πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά. Οι εταιρείε μα είναι πρόθυσμε να προσαρμοστούν σε καθυστερήσει προκειμένου να έχουμε καλή εφαρμογή προκειμένου να πετύχουμε το αρχικό όραμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να υπάρξει πιο επίσημη διαβούλευση με τις επιχειρήσεις που θίγονται περισσότερο από αυτές τις νομοθετικές προτάσεις. Η σημερινή διαδικασία διαβούλευσης θα πρέπει να βελτιωθεί και να ευθυγραμμιστεί κυρίως όλα όλα τα έγγραφα θέσει και τα σχόλια που στέλνουν οι εμπορευόμενοι για τι προτάσει Κομισιόν θα πρέπει να διατίθενται σε όλου του ενδιαφερομένου και του εμπορευομένου και τα κράτη-μέλη και αυτό εγκαίρω. Η πλήρη διαφάνεια είναι ουσιώδη για ορθή εφαρμογή του εξυγχρονισμένου τελωνιακού κώδικα. Είναι σημαντικό και ο MCC και η προτινόμενη νομοθεσία ε, να συνοδευτούν με νέα συστήματα πληροφορικής που θα ε, φροντίσουν και στην ορθή εφαρμογή. Ε, σήμερα βλέπουμε το αντίστροφο, δηλαδή δεν ε, έχουμε διαδικασίες που τελικά εξυπηρετούν τους στόχους του εξυγχρονισμένου τελεωνιακού κώδικα. Η εφαρμογή του εξυγχρονισμένου τελεωνιακού κώδικα δεν πρέπει να εμποδίσει να ε, έχουμε τη σύνταξη νομοθεσία έχοντας ε, κατά νου ε, κάθε εξυγχρονισμό λόγω τη σημερινή οικονομικής κρίσης σήμερα είναι ακόμη πιο σημαντικό να διευκαλύνουμε το εμπόριο, να περιορίσουμε την γραφειοκρατία και το κόστος για τις επιχειρήσεις. Αν υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία, είναι σαφές τώρα ότι όλες αυτές οι πρωτοβουλίες θα πρέπει να προωθηθούν ε, επιγόντω. Ο στόχος του MCC είναι να απλοποιήσει, να εξυγχρονίσει ε, τα τελειωνιακά σύστημα της Τελειωνιακής Ένωσης που είναι σημαντικά για τη μελλοντική ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη της Ευρώπης. Αυτό είναι το όραμα που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ψήφισε για τον εξυγχρονισμένο τελωνιακό κώδικα και αυτό το όραμα συμμεριζόμαστε και εμείς σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και έχουμε, και αντίγραφο και της δικής σας Τώρα στο επόμενο θέμα που προκύπτει από αυτό και προσπαθήσαμε και αυτό να το δούμε, ειδικά όσον αφορά τις προτάσεις της ε, Κομισιόν για αλλαγές στην προηγούμενη στρατηγική που θα πρέπει να εξετάσουμε. Οπότε μέχρι στιγμής έχουν ζητήσει τον λόγο ο κύριος Κρότσμαν και η κυρία Χάντσλικ. Θα του ζητήσω λοιπόν να παρέμβουν. Κύριος Κρότσμαν, ευχαριστώ. Μόλις ακούσαμε πόσο σημαντικό είναι ο εξυγχρονισμένος τελωνιακός κώδικας να ενεργοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν. Το είχαμε πει για το 2013, αναβλήθηκε, ε, αναβλήθηκε μέχρι πότε υπάρχει κάποιος τρόπος να ασκήσουμε πίεση έτσι ώστε το 2014 να εισαχθεί ο εξυγχρονισμένος τελωνιακός κώδικας αναβολή και να τα αφήνουμε ανοιχτό δεν είναι ικανοποιητικό για τους φιλελεύθερους. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήθελα και εγώ μιλήσω εξ ονόματος κυρίας ε, Κορχόλα η οποία λείπει σήμερα δυστυχώς της ε, του συγκεκριτές να αναφέρω κάποια πράγματα. Πράγματι, ο εκτελονισμός είναι πάρα πολύ σημαντικός ε, για την ανταγωνιστικότητα της Ένωσης. Ηλεκτρονικός εκτελονισμός μπορεί να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά μας ε, με το να γίνει πιο σύγχρονος και αποτελεσματικό και να απαντά στι ανάγκε των χρηστών. Όμω, οι καθυστερήσει στον ηλεκτρονικό εκτελονισμό Φαίνεται πως είναι κάτι το μη ρεαλιστικό, καθώς δεν μπορεί να λειτουργήσει πλήρως ε, το σύστημα το ηλεκτρονικό. Κάποιοι λένε πως είναι απλά μια πολιτική απόφαση και δεν χρειάζεται περισσότερος χρόνος για την προετοιμασία του συστήματος. Η κυρία Κόρχολα θα ήθελε να κάνει την εξή ερώτηση. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την προθεσμία του 2013, θα την επιτύχουμε ή όχι. Και ποιος είναι ο κίνδυνος εάν αποφασίσουμε να δώσουμε περισσότερο χρόνο για το έργο αυτό. Και επίσης θα ήθελε να κάνει και μια ερώτηση, κυρία Κορχόλα, για το καθεστώς του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα, δηλαδή ποια θα είναι τα βασικά βήματα που θα πρέπει να γίνουν για να προσελκύσουμε τις επιχειρήσεις να ζητήσουν αυτό το καθεστώς. Αλλά θεωρώ πως απαντήθηκε ήδη αυτό από τον τελευταίο μιλητή, αλλά αν θέλετε να το αναπτύξετε ε, θα ήθελα κάποιες απαντήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Ρούλε επίσης. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Αλλά αυτό το οποίο παρατήρησα εγώ είναι πως υπάρχουν κάποιες αντιφάσεις. Η ομάδα μας, όπως ξέρετε, ενδιαφέρεται να υποστηρίξει την αναβολή γιατί εμείς ε, θεωρούμε πως θα πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα πράγματι που να λειτουργεί και να μην ε, βιαστούμε και να μειώσουμε τις δυνατότητες του πληροφοριακού στήματος. Αλλά αυτό το οποίο μου προξένησε εντύπωση ήταν πως από τις τοποθετήσεις μας είπαν πως θα πρέπει να προσαρμοστούν στο μεταβατικό χρόνο οι διατάξεις, αλλά πως θα γίνουν πιο περιπλοκές, γιατί το βρήκα κάπως ε, περίεργο αυτό το τοποθετήσεις, γιατί δεν ήταν αυτός ο στόχος της αναβολής, ε, να γίνουν πιο πολύπλοκες οι διατάξεις. Το άλλο το οποίο με ενδιαφέρει, κάτι το οποίο ακούω ξανά και ξανά, είναι πως ε, δεν ε, εμπλέκονται οι ενδιαφερόμενοι. Το έχουν πει συχνά αυτό και οπωσδήποτε οι διαδικασίες θα πρέπει να εξυπηρετούν τους εμπλεκόμενους αν δεν ακούγεται η άποψή τους ε, είναι ένα πρόβλημα. Και τελευταίο ερώτημα, το οποίο ακούστηκε και στην πρώτη παρέμβαση και είχαμε ούτως ή άλλως και χθες συζήτηση για τα τελωνία το ζήτημα των λοιπόν απαιτήσεων που υπάρχουν, αυτά τα οποία θέτει η πολιτική ως απαιτήσει στον τελωνιακό κώδικα και οδηγεί σε ένα σύστημα που γίνεται όλο πιο περίπλοκο. Θα ήθελα να μάθω λοιπόν πώς το αντιμετωπίσουμε αυτό. Um, Ωραία. Θα ήθελα να προσθέσω κι εγώ, γιατί και εγώ είμαι σκιώδης εισηγητής για το θέμα. Δύο ζητήματα προκύπτουν σαφέστατα. Το θέμα των εγκεκριμένων οικονομικών φορέων και το θέμα της εφαρμογής του εξυγχρονισμένου τελωνιακού κώδικα και των εφαρμοστικών διατάξεων. Όπως είπε και ο κύριος Βόγκαν, οι εισαγωγεί ή όσοι εμπλέκονται με το εξωτερικό εμπόριο καλούνται να αντιμετωπίσουν 27 διαφορετικά συστήματα. Ε, ενώ είχαμε υποσχεθεί ήδη να λειτουργεί ένα ενιαίο σύστημα. Απευθύνω μία έκκληση λοιπόν. Η νομοθεσία δεν πρέπει να ακολουθεί την τεχνολογία. Το αντίθετο πρέπει να γίνεται με αυτή την αναβολή από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ξέρω να ακολουθούμε αυτό το σωστό προσανατολισμό. Ε, κατόπιν, για τους συγκεκριμένους οικονομικούς φορείς, ε, νομίζω ότι αυτό το θέμα θα πρέπει να ξεχωριστεί, διότι υπάρχουν σαφέστατα εμπορικά πλεονεκτήματα για τη λειτουργία αυτού του συστήματος, ανεξάρτητα με το αν έχουμε ένα ολοκληρωμένο τελωνιακό σύστημα. Έχουμε πρόβλημα μικροφωνισμών. Κύριε Ζελίνσκι, θα τελειώσουμε μέσα. Θα αρχίσουμε με τον κύριο Βόγκαν και θα πάρουμε τους ομιλητές ε, αντίστροφα. Ευχαριστώ. Δύο είναι τα ζητήματα. Ο ΑΕΟ, e ο εγκεκριμένος οικονομικός φορέας, ε, είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό το ζήτημα. Προς το παρόν δεν προσφέρει ωφέλη στις επιχειρήσεις. Και εφόσον έχουν έτσι τα πράγματα, εξετάζουμε προσεκτικά αυτό το ζήτημα και τις προτάσεις για τον εξυγχρονισμένο τελωνιακό κώδικα. Δυστυχώς, σε αυτό το πλαίσιο φαίνεται ότι αυτό που προσφέρει η τωρινή απλούστευση στις επιχειρήσεις είναι ωφέλη που επαναγοράζονται και χρησιμοποιούνται ε, όσο ωφέλη. Ξέρετε τι εννοώ. Εννοώ ότι μπορεί εσύ ως, ε, εμπορικό, ως εμπορευόμενος, αλλά στη συνέχεια μπορεί να αποσυρθεί αυτό και να χρησιμοποιηθεί ως ανταγωνιστικό όφελος από έναν εγκεκριμένο οικονομικό φορέ, γιατί εκπροσωπούμε και μεγάλες επιχειρήσεις και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σας διαβεβαιώ ότι για τις μικρομεσαίες είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα με αυτό το τωρινό καθεστώς. Ε, σημειώθηκε καθυστέρηση σχετικά με την ημερομηνία θέσης εφαρμογής ε, του κώδικα ε, σε σχέση με το, την αρχικά προβλεπόμενη ημερομηνία το 2013. Όμως, χάρη σε αυτή την καθυστέρηση θα κερδίσουμε χρόνο και θα φροντίσουμε ώστε και τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχουν το χρόνο να αναπτύξουν συστήματα που θα λειτουργούν υποστηρικτικά για τον εξυγχρονισμένο κώδικα, διότι φοβούμε ότι τα συστήματα όσοι έχουν τώρα δεν είναι σε θέση να υποστηρίξουν τα καθεστώτα και τις διατυπώσεις που προβλέπονται στον ε, εξυγχρονισμένο κώδικα και δυστυχώς εξαιτίας πείρας θα σας πω ότι χρειάζονται περίπου έξι χρόνια ε, για, από τη σύλληψη της ιδέας σχετικά με το πώς ιδανικά θα έπρεπε να είναι το σύστημα μέχρι ότου να συμφωνήσουν όλοι, δηλαδή ο κλάδος, η Επιτροπή και τα κράτη-μέλη. Ελπίζω λοιπόν ότι με αυτή την καθυστέρηση θα έχουμε χρόνο ούτω ώστε να ιδρύσουμε, να θεσπίσουμε ένα πιο αποτελεσματικό σύστημα που θα λειτουργεί υποστηρικτικά για την νομοθεσία. Ναι, παρακαλώ. Ε, συμφωνώ απολύτως με τον κύριο Βόγκαν. Ως προς ε, την εφαρμογή των νέων εφαρμοστικών διατάξεων του κώδικα, κατά πάσα πιθανότητα είναι πολύ καλύτερη λύση αυτή της αναβολής. Έτσι, οι επιχειρήσεις θα έχουν το χρόνο να ευθυγραμμίσουν τις νέες υποδομές τους ε, ως προς τις ε, εφαρμοστικές διατάξεις. Τα συστήματα πληροφορικής δεν θα είναι έτοιμα μέχρι το 2013 27 διαφορετικά συστήματα πληροφορικής έχουμε προ το παρόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις διασαφήσεις Φερρυπίν για να ενσωματωθούν σε ένα ενιαίο σύστημα. Κατά πάσα πιθανότητα δεν είναι εφικτό να γίνουν ε, αυτά τα πράγματα μέχρι το 2013. Ω προς τα ωφέλη τώρα για όσοι έχουν το καθεστώς του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα, νομίζω το ανέφερα στην παρουσίασή μου, πέρα από το να, είναι, να έχει κάποιος αυτό το καθεστώς, οι επιχειρήσεις ε, χρειάζονται και οικονομικά κίνητρα ε, για να κάνω αυτές τις διατυπώσεις. Ε, Άρση της υποχρέωσης δήλωσης ασφαλείας στις τελωνιακούς σταθμούς ή άλλες διευκολύνσεις για την καταβολή των δασμών ή για τον εισαγωγικό ΦΠΑ, όλα αυτά είναι μέτρα που θα καλωσόριζαν οι επιχειρήσει πέρα από το καθεστώς του οικονομικού φορέα. Αυτά από πλευρά μου. Η κυρία Έγκνερ τώρα μας ενδιαφέρει να ακούσουμε και την άποψη, την ε, παγκόσμια άποψή σα, γιατί εκπροσωπείτε τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τελωνίων. Ε, ε, ναι, ε, ομολογώ ότι δεν είμαι καινούργια σε αυτό το θέμα, γιατί ήμουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είχα ασχοληθεί με το θέμα του ε, εγκεκριμένου οικονομικού φορέα. Λοιπόν, ε, σε παγκόσμιο επίπεδο θα έλεγα ότι γιατί το AEO ανήκει στα δικά μας πρότυπα επίσης ε, και ως προς την εφαρμογή από τα μέλη μας διαπιστώνουμε ότι όλοι αγωνίζονται με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή επιδιώκουν να βρουν τα σχετικά ωφέλη του καθεστώτος ε, και έχουν δημιουργηθεί πολύ καλές σχέσεις ανάμεσα στους εμπορευομένους και έχει επέλθει μια απλούστευση εδώ και ε, πολλά χρόνια. Δύσκολο όμως μπορούμε να έχουμε απτά ωφέλη, είναι ευκολότερο ε, για τα κράτη-μέλη που δεν είχαν καμία διαδικασία απλούστευσης και τα τελωνία τους βασίζονταν στους ελέγχους. Εκεί φαίνεται η διαφορά με το νέο καθεστώς. Καταλαβαίνω ότι όλοι αγωνίζονται, αλλά ίσως ε, στην ομάδα επαφής για το εμπόριο καλό θα ήταν να γίνει ένας κατάλογος όλων των πλεονεκτημάτων ή μάλλον έχει συνταχθεί ο κατάλογος από την ομάδα επαφής για το εμπόριο, δεν είναι μεγάλος ο κατάλογος, αλλά ενδεικτικά αναφέρονται τα ωφέλη που προκύπτουν από το καθεστώς μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχουν και λιγότερο από τα ωφέλη μέσα στον κατάλογο. Θα έλεγα όμως ότι πρέπει να υπάρξουν ότι υπάρχουν απτά ωφέλη για τις ε, τελωνιακές αρχές που χρησιμοποιούν τις διατάξεις ε, διευκόλυνσης των εμπορικών συναλλαγών. Ως προς τα συστήματα πληροφορικής, θα ανέφερα μία πρωτοβουλία στα πλαίσια του οδικού χάρτη, τα τελωνία, δηλαδή για τον 21ο αιώνα, και βάσει αυτού ε, επικουρούμε τα κράτη-μέλη στην εκπόνηση τεχνικών προτύπων για να υπάρχουν και πιο διαρθρωμένες ανταλλαγές απόψεων ανάμεσα στις τελωνιακές αρχές. Ε, πολύ καλό παράδειγμα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι η μόνη, η STS επίσης έχει σχετικά προγράμματα. Αυτές ε, οι ανταλλαγές απόψεων επηρεάζουν τη διαμόρφωση των νέων προτύπων και με τις συζητήσει μα καλύπτουμε και νομικά ζητήματα, ζητήματα διακυβέρνηση, ε, επιχειρησιακά μοντέλα, οικοδόμηση δυναμικότητας, ε, νέε αρχιτεκτονικέ νέα περιβάλλοντα πληροφορικής. αλλά δεν αναπτύσσονται νέα συστήματα, πρότυπα, πρωτόκολλα και ε, κατευθυντήριες γραμμές εκπονούμε. Οπότε, ίσως είναι δύσκολο η νομοθεσία να συμβαδίζει με τα συστήματα πληροφορικής, ε, να σημειώνεται εξελίξη και στους δύο τομείς ε, ταυτόχρονα. Ο κύριος Ελίνσκι μήπως ε, θέλει να παρέμβει, θέλετε τώρα το λόγο, τόσο θα ξαναπάρετε το λόγο μετά, αν θέλετε εν συντομία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να ομαδοποιήσω τις ερωτήσεις. Ένα πολύ σημαντικό θέμα είναι αυτό της αναβολής και τη σχέση που έχει με την μετεξέλιξη των συστημάτων πληροφορικής. Δηλώνω λοιπόν επίσημα ότι δεν υπάρχει καμία πολιτική απόφαση. Οι πολιτικοί θα ήθελαν σήμερα ή αμελητοί να εφαρμόσουν αυτά και σίγουρα πριν το 2013. Όμως οι λύσεις θα πρέπει να είναι και εφικτές. Και ε, το θέμα των, ε, της αποτελεσματικότητας των λύσεων συνδέεται άρρηκτα με το θέμα των συστημάτων πληροφορικής. Άρα ε, καλούμεθα να κατανοήσουμε με ποιο τρόπο μπορούμε να εφαρμόσουμε τον εξυγχρονισμένο τελωνιακό κώδικα ε, σταδιακά. Θα θέλαμε η πρώτη φάση να τεθεί σε εφαρμογή ε, το ταχύτερο δυνατόν, αλλά μόλις ολοκληρωθεί ε, η πρώτη προσπάθεια σίγουρα θα προσκομίσει ωφέλη και στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και θα τονώσει και την ευρωπαϊκή οικονομία. Θα ήθελα να πω ότι τα επόμενα 5-10 χρόνια δεν θα έχουμε ένα ε, κεντρικό σύστημα σύστημα για πολλούς λόγους, για τεχνικούς λόγους, ε, για... Ε, χρειάζονται πολύ ε, πολλοί οικονομικοί πόροι, τα κράτη-μέλη έχουν επενδύσει εκατομμύρια ευρώ και το... για τα συστήματα πληροφορικής τους και τώρα πρέπει να τα μηδενίσουμε όλα και να αρχίσουμε από την αρχή. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Ε, και είναι πάρα πολύ δύσκολο επίσης να συνεπάρξουν και να συλλειτουργήσουν τόσα διαφορετικά συστήματα. Κάποια, ε, κάποιες διατυπώσεις θα γίνονται σε κεντρικό επίπεδο. Ε, ε, θέλουμε να μειώσουμε κυρίως τις επικαλύψεις. αυτός είναι ένας πρώτος στόχος. Δεν θέλουμε να έχουμε τα 27 διαφορετικά συστήματα και καθημερινά να έχουμε 27 διαφορετικές αιτήσει από πλευρά ε, των ε, κρατών μελών. Ε, χάνονται πόροι έτσι και υπάρχουν επικαλύψεις. Αυτά για την αναβολή και τα συστήματα πληροφορικής. Επαναλαμβάνω και πάλι, ότι αν δεν έχουμε ένα ε, ε, ε, σύστημα πληροφορικής που να λειτουργεί εύρυθμα, ο εξυγχρονισμός του λεωνιακού Κώδικας δεν θα αποφέρει τα ωφέλη που αναμένουμε όλοι. Το θέμα τώρα του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα που ενδιαφέρει τους πάντες Έχουμε κάποια καθυστέρηση με τα στατιστικά στοιχεία. Σχεδόν 10.000 είναι ο αριθμός που έχουμε προς το παρόν. Χορηγούνται τέτοια καθεστώτα, δίνονται άδειες και αναγνωρίζεται η αξία του καθεστώτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμη και οι μικρέ επιχειρήσει εφαρμόζουν το καθεστώ του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα. Οι μικρέ, ή μάλλον οι μεσαίες επιχειρήσει επιζητούν τη χορήγηση του καθεστώτος και υποφελούνται από αυτή. Τα ωφέλη, ναι, ε, αναμένονται προ το παρόν, δεν είναι τόσο πολλά. Όμω, στο μέλλον, ε, με τη δομή του εξυγχρονισμένου τελωνιακού κώδικα έχουμε διευκολύνσει, απλουστεύσει, διάφορε νέε διατυπώσει και δεν μπορεί να ισχυριστεί κανεί ότι το, ο εγκεκριμένο οικονομικός φορέας έχει όλες τις εγκρίσεις αυτόματα επειδή είναι εγκεκριμένο οικονομικός φορέας και όλες τις διευκόλυνσεις. Μα εξαρτάται γιατί πράγμα μιλάμε, για τη μεταφορά εμπορευμάτων, για τις ναυτιλιακές εταιρείε κτλ. κτλ. Αν θέλετε ε, αυτόματη έγκριση για όλες τις διατυπώσεις απλούστευσης θα ε, χρειαζόταν ένα ε, μακροσκελέστατο κατάλογο ε, κριτηρίων. Οπότε έχουμε το βασικό καθεστώς του βασικού οικονομικού φορέα και η βασική αρχή έχει ως εξή. Ο AEO δεν χρειάζεται να επαναλάβει τη διατύπωση που καλύπτεται από το καθεστώς του. Ορισμένε φορέ για ενιαίες αποστολές, για τις ε, θαλάσσιες μεταφορές πρέπει να προσθέσουμε κάποια κριτήρια. Αλλά πάντως ε, ο εγκεκριμένος φορέας δεν ασχολείται καθόλου με τα κριτήρια που ε, επιβάλλονται στις αεροπορικές εταιρείε, παραδείγματο χάρη. Θα προκύψουν τα ωφέλη σταδιακά και λένε και περισσότερο. Τώρα για τις διαβουλεύσεις με το εμπόριο ακούσαμε πολλά παράπονα. Μόλις έλαβα μία επιστολή με συγχαρητήρια. Ε, ήταν μία δήλωση από τη συνεδρίαση της ομάδας επαφής για το εμπόριο, που, βάσει της οποίας ε, έχουμε μία άνευ προηγουμένου διαβούλευση με τον κλάδο και ε, στην ομάδα επαφής συμμετέχουν οι εμπορευόμενοι σε, με τηλεδιάσκεψη σε εικονικές τηλεδιασκέψεις, έχουμε εργαστήρια σεμινάρια και πάντοτε συμμετέχει και ο κλάδος. Ε, Βεβαίω. όπως είπε σωστά ο συνάδελφο. δεν υπάρχει κοινή θέση μέσα στην ομάδα επαφής γιατί εκπροσωπούνται διαφορετικά συμφέροντα από διαφορετικούς τομείς ε, του εμπορίου. Ως εκ τούτου δεν δεν είναι εύκολο και πάντοτε θα είναι κάποιοι που δεν είναι ικανοποιημένοι. Θα υπάρχουν κάποιοι που δεν είναι ικανοποιημένοι. Ξέχασα να πω και κάτι ε, ε, δεν ακολουθεί η νομοθεσία την ε, τεχνολογία της πληροφορικής. η νομοθεσία ακολουθεί τις διατυπώσεις. Πώς λειτουργεί η διατύπωση, αυτό εξετάζουμε και μετά ακολουθεί η νομοθεσία και μετά το σύστημα πληροφορικής. Γιατί πρέπει να είναι και τεχνικός εφικτό να γίνει κάτι. Δεν γίνονται όλα. Τέλος. Τα τελωνία δεν σχετίζονται μόνο με την διευκόλυνση, σχετίζονται με τις ελέγχους, με τα έσοδα. Ε, με την ασφάλεια, την προστασία της ε, κοινωνίας, τα πνευματικά δικαιώματα και το καθεξής και ζητώ συγγνώμη που μακρηγόρησα. Ναι, πράγματι. Υπήρχαν πολλά ζητήματα βεβαίω, στα οποία έπρεπε να απαντήσετε. Κάνατε μια τέλεια εισαγωγή για το επόμενο μέρος της συζήτησής μας που αφορά τους ελέγχους και την ασφάλεια. Και βεβαίω για τη συνεργασία, το πώς ε, μπορεί να βελτιωθεί, γιατί νομίζω πως θα τα κάνουμε μαζί αυτά τα δύο. Καλωσορίζω ορίζω επίσης για δεύτερη συνεχή ημέρα τον ε, Δ. Πίτερ Χόμπινγκ, ο οποίος έκανε μία μελέτη για τους συναδέλφους στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών για την τελωνιακή συνεργασία στην περιοχή ασφάλειας και δικαιοσύνης για την διαχείριση των εξωτερικών συνόρων. Ήταν εδώ χτες για να παρουσιαστεί η μελέτη, οπότε παρακολουθούμε τα ζητήματα, αλλά ευχαρίστω εάν θέλετε να αναφερθείτε σε κάποια από τα ζητήματα. Υπάρχουν αντίγραφα της μελέτης αν θέλετε να τα δείτε. Οπότε περνάμε στο κομμάτι το επόμενο και θα ζητήσω να μιλήσει ένας άλλος εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κύριος Καστρισιανάκης, ελπίζω να είπα στο το όνομά σας, Διευθυντής ε, Ασφάλειας, ε, Αποτυχήματα και Κακόβουλες Ενέργειες, Διευκόλυνση Εμπορίου και Διεθνούς Συντονισμού στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχει τον λόγο για 5 λεπτά. Ευχαριστώ. Όπως είπαν και άλλοι ομιλητές, ε, αυτή τη στιγμή βλέπουμε μια, ένα σημαντικό μετασχηματισμό των τελωνίων που φεύγουμε απλά από φορολογικά ζητήματα και πάμε προς την ασφάλεια και την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων. Και το θέμα είναι πως θα μπορέσουμε να έχουμε αφενός ε, την ασφάλεια και την προστασία και αφετέρου την διευκόλυνση του εμπορίου χωρίς να βλαπτεί το ένα από τα δύο. Οπότε το σημαντικό εδώ πέρα είναι το πώς θα εφαρμοστούν μέτρα τα οποία θα επιτυχάνουν και περισσότερη προστασία και περισσότερη διευκόλυνση και επιτάχυνση του εμπορίου. Οπότε σε αυτό το πλαίσιο εργαζόμαστε ανεξαρτήτως ε, καθυστερήσεων ε, στην ε, υιοθέτηση του εξυγχρονισμένου τελωνιακού κώδικα. Ιδιαίτερα όσον αφορά τον τομέα της ασφάλειας, θα ήθελα να αφαιρθώ στην τροπολογία ασφαλείας που εισήχθη πριν από τέσσερα χρόνια και τώρα ε, έχει εφαρμοστεί πλήρως από 1ης ε, πρώτου 2011 και στην ε, αλλαγή αυτή είδαμε την εισαγωγή των εκ των προτέρων δηλώσεων, κανόνων κινδύνου και ανάλυσης κινδύνου και επίσης βεβαίως προβλέπουμε το σύστημα του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα. Ως προς αυτό, όπως είπε και ο Μίρεκ, έχουμε αυτή τη στιγμή γύρω στα 5.800 επιστοποιητικά τέτοιων εγκεκριμένων φορέων και υπάρχουν ωφέλη και στον τομέα της ανάλυσης ε, κινδύνου και ωφέλη διευκόλυνσης και πιθανά ωφέλη όσον αφορά την αμοιβή αναγνώριση με τρίτες χώρες. Όσον αφορά την αλλαγή που επήλθε στην ασφάλεια, πρέπει να σας πω πως παρακολουθούμε την εφαρμογή από 1η Πρώτου 2011, ειδικά ε, υπό το φως των περιστατικών στην Ιεμένη και άλλων περιπτώσεων όπου ε, είχαμε ε, αεροπορικά φορτία. Προσπαθούμε να δούμε πού βρίσκονται οι δυσκολίες και να τις αντιμετωπίσουμε ε, ειδικά όσον αφορά αεροπορικά φορτία, όσον αφορά τα χρονικά όρια, παραδείγματο χάρη για την υποβολή πληροφοριών εκ των προτέρων για να αποφύγουμε, να επιτρέψουμε μάλλον ε, την ε, δυνατότητα στα τελωνία να παρέμβουν πριν φορτωθούν ε, επικίνδυνα, τυχόν επικίνδυνα υλικά και βεβαίως ε, να δούμε και τις διατυπώσεις υποβολής και εξαιρέσεις στον τομέα αυτό. Και αναμένουμε εντός του έτους ίσως να υποβάλουμε μια νομοθετική πρόταση για να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα αυτά. Ένα σημαντικό μέρος αυτού είναι το πώς θα ενισχυθεί είναι ο συντονισμός ε, και η συνεργασία και να συνδυαστούμε βεβαίω και με άλλες υπηρεσίες στα σύνορα που έχουν ε, την ευθύνη της ασφάλειας. Επίσης το θέμα της ασφάλειας της ε, ασφάλειας από κακόβουλες ενέργειες ιτίζεται και με την ασφάλεια από ατυχήματα γιατί υπάρχει το λεγόμενο πλαίσιο το κοινό πλαίσιο διαχείρισης κινδύνου γιατί υπάρχει η πτυχή της ασφάλειας παραδείγματο χάρη στο πλαίσιο της Ιαπωνικής ποινική κρίσης. Ε, να αναφερθώ επίσης στα πνευματικά δικαιώματα. Όπως είπε και ο Επίτροπος ο κύριος Σεμέτα την τελευταία φορά που ήρθε στην Επιτροπή σας, είπε πως έχουμε μια νέα πρόταση για κανονισμό τελωνιακό που παρουσιάστηκε στο Συμβούλιο και Κοινοβούλιο και σημασία έχει να κινηθούμε γρήγορα για να ενισχυθούν οι άμυνες μας όσον αφορά την παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, να ευθυγραμμιστούν οι διαδικασίες και να έχουμε έτσι πιο μεγάλη αποτελεσματικότητα. Τέλος, για τη διεθνή συνεργασία, ενώ στις εθνικές πολιτικές βεβαίως ε, βασιζόμαστε στο ιστορικό επίπεδο, πρέπει να ενισχυθεί και η διεθνή συνεργασία για να επιτύχουμε τους ε, στόχους μας για ασφάλεια και πνευματικά δικαιώματα και στον τομέα αυτών. Στο πλαίσιο συμφωνιών που έχουμε ήδη διαπραγματευτεί ή διαπραγματευόμαστε, προσπαθούμε να ενισχύσουμε αυτή τη συνεργασία, ειδικά η Ελβετία και η Νορβηγία αναφέρθηκαν, καθώς χώρες αυτές αποτελούν τμήμα της του Ευρωπαϊκού Χώρου Τελωνιακής Ασφάλειας συνεργαζόμαστε στενά και με τις υποψήφιες χώρες, τα Δυτικά Βαλκάνια, στο πλαίσιο της διεύρυνσης, στα ανατολικά σύνορα με την Ρωσία, προωθούμε στρατηγικό πλαίσιο τελωνιακής συνεργασίας, καταπολέμησης ε, του λαθρεμπορίου. Όσον αφορά τις ΗΠΑ προσπαθούμε να βρούμε κάποια θέματα όσον αφορά την ασφάλεια και τις αλυσίδες εφοδιασμού. Επίσης για την Κίνα το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων και ασφάλεια από κακόβουλες ενέργειες και η αμοιβαία αναγνώριση είναι σημαντικές και ως προς αυτό νομίζω ότι έχουμε επιτύχει με την Ιαπωνία. Έχουμε επιτύχει την αμοιβαία αναγνώριση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ που μας παρουσιάσατε το πλαίσιο αυτό ο κανονισμός για τη συνεργασία ε, για την επιβολή της νομοθεσίας για τα τελωνία για τα πνευματικά δικαιώματα έχει φτάσει σε αυτή την επιτροπή. Θα διορίσουμε ένα εισηγητή σύντομα. Θέλω να καλωσορίσω ένα διακεκριμένο μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου, τον καθηγητή Χουάν Ραμάλο. Ξέρω ότι το Ελεκτικό Συνέδριο ενδιαφέρεται πάρα πολύ για τα τελωνία, τις τελωνικές διαδικασίες και τους ελέγχους στον ευρωπαϊκό χώρο. Και ήθελα λοιπόν να το καλέσω να μας παρουσιάσει τις απόψεις του σχετικά, ο κ. Ραμάγιο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν ε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ε, πρόσκλησή σας ε, να συμμετέχω εδώ και θα προσπαθήσω να παρουσιάσω την άποψή μου στα πέντε λεπτά που μου έχετε δώσει. Όταν ακούω τα λέγια εξυπνισμένος τελωνιακός κώδικας έρχονται στο νου μου διάφορες ιδέες, διευκόλυνση του εμπορίου, αυτοματημένη διαχείριση κινδύνου, μεγαλύτερη ψηφιοποίηση, ε, ταχύτερος ε, εκτελονισμός ε, και χωρίς χαρτιά. Όμως τίθεται και άλλες ανησυχίες για την προστασία του καταναλωτή, της υγείας του καταναλωτή, προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων, εγγυήσεις, ό,τι αφορά την αλυσίδια φοδιασμού, κατά πολέμηση της ε, παράνομης διακίνησης αγαθών και προστασίας του περιβάλλοντος. Αυτά είναι θέματα ανησυχίας ε, που γενικά ε, ανησυχούν και τους νομοθέτες, τα ενδιαφερόμενα μέρη και γενικά το κοινό, όπως βλέπουμε και από την προσοχή που δίνεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ως μέλος όμως του ελεκτικού συνεδρίου έχω και άλλες σημαντικές ανησυχίες κατά νου όπως ε, την ακαιρεότητα της εισπραξής των εσόδων, την καταπολέμηση ε, της απάτης του λαθρεμπορίου και της ε, φόρο της τήρησης, της συμμόρφωσης με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η κοινή εμπορική πολιτική, η κοινή αγροτική πολιτική και η ορθή λειτουργία της Τελωνιακής Ένωσης και της εσωτερικής αγοράς. Αυτή ήταν ε, η πρώτη πρόθεση της ειδικής έκθεσης του Ελεκτικού Συνεδρίου υπαριθμών είναι του 2010 με το τίτλο «Ελέγχονται αποτελεσματικά οι απλοποιημένες τελωνεϊκές διαδικασίες που εφαρμόζονται στις εισαγωγές» δεν είναι το ότι η έκθεση παραγνωρίζει τους υπόλοιπους στόχους, αλλά στην ίδια την εισαγωγή επαναλαμβάνεται ότι με τον εξχρονισμένο τελωνιακό κώδικα ανοίγει ο δρόμος για την διευκολύνση του εμπορίου και ότι οι νέες απλοποιημένες διαδικασίες αποτελούν ένα στοιχείο κλειδί για την διευκολύνση του εμπορίου. Παρ' αυτά, εφιστούμε την προσοχή των νομοθετών και των ενδιαφερομένων μερών στο εξή ότι πριν να συνεχίσουμε στη στην διαδικασία της απλούστευσης των τελωνικών διαδικασιών θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις ανησυχίες που ανέφερα προηγουμένως. Κατά την άποψή μου, μπορούν ε, να καταργηθούν πρώτεροι ελεγχοί για την εισαγωγή αγαθών ε, όπως ε, ρυθμίζουν οι απλουστευμένες διαδικασίες αν αυτή η έλλειψη ελέγχου αντισταθμίζεται από την υλοποίηση ελέγχων audits στους εμπορευόμενους πριν την άδεια που δίνεται για τη χρησιμοποίηση του απλουστευμένου συστήματος και με exposed ελέγχους στο εμπόρευμα, κατά την παράδοση του εμπορεύματο. Τώρα, αναφέρω και ένα δεύτερο στοιχείο, πώς λειτουργούν τα κράτη-μέλη. Πράγματι, διαπίστωσε το ελεκτικό συνέδριο ότι τα κράτη-μέλη εφαρμόζουν ε, ε, ε πολλές φορές ε, τον έλεγχο ε, στα πλαίσια των απλουστευμένων διαδικασιών. Έτσι λοιπόν οδηγούμαστε, οδηγούμαστε τελικά σε ελέγχους κακής ποιότητας ή ανεπαρκώς τεκμηριωμένους ελέγχους ε, ε, πριν να δοθεί άδεια σε ένα εμπορευμόμενο να χρησιμοποιήσει τις απλουστευμένες διακασίες. Μικρή χρήση ε, της, ε, αυτόματης, της τεχνικής αυτόματης επεξεργασίας για την υλοποίηση των ελέγχων κατά τις απλουστευμένες διαδικασίες. Τρίτον, υπερβολική χρήση των πρακτικών απλούστευσης, κυρίως της απαλλαγής κοινοποίησης ότι η διαδικασία εκτολονισμού και αυτό εμποδίζει να γίνονται κίνδυνοι έλεγχοι με συγχωρείτε βάση αξιολόγηση κινδύνου πριν εισαχθούν τα αγαθά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίση, εξ πόστα έλεγχου των εγγράφων ε, ε, κακή ποιότητα. Και βλέπουμε ότι δεν γίνονται συχνά έλεγχοι, ούτε στοχεύουμε ορθά στις συναλλαγές. Αλλά για τι πράγμα μιλάμε. Πέρα από το ότι οι τελωνιακοί δεσμοί ε, συνιστούν μόνο το 12,2% του ε, κοινοτικού ΕΕΠ ενώ η συμμετοχή στο καθάριστο εθνικό προϊόν είναι της τάξης του 73,4% δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι μόνοι ομοιόμορφοι φόροι σε ευρωπαϊκό επίπεδο που υπάρχουν σήμερα είναι η παραδοσιακή διπόρη. δηλαδή τα, η ε, τελωνιακή δασμή κυρίω και θα πρέπει να έχουμε ομοιόμορφη εφαρμογή σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς ε, στα πλαίσια της Τελωνιακής Ένωσης τα τελωνία, τα τελωνία σε όλο το μήκος και πλάτος των ευρωπαϊκών συνόρων λειτουργούν σαν να είχαμε ένα και μόνο τελωνία. Δηλαδή έχουμε ισότιμη μεταχείριση των οικονομικών φορέων χωρίς να λαμβάνεται υπόψη που υλοποιείται η τελεωνιακή επιχείρηση. Από τη σκοπιά αυτή είναι σημαντικό να διαπιστώσουμε, να παρατηρήσουμε ποιες είναι οι χώρες που προβαίνουν σε περισσότερες εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από αυτές τις εισαγωγές ε, ποια ποσοστό, σε ποιο ποσοστό ακολουθείται η απλουστευμένη διαδικασία. Καταρχήν το 74% όλων των εισαγωγών του 2009 υλοποιήθηκε υπό την απλουστευμένη διαδικασία. Δεύτερον, έχουμε ουσιαστική διαφορά μεταξύ των κρατών μελών σε ό,τι αφορά τη χρήση των απλουστευμένων διαδικασιών. Καθώς τρία κράτη-μέλη, Γερμανία, κάτω χώρες και Ηνωμένο Βασίλειο, υλοποιούν το 85% των απλουστευμένων διασαφήσεων. Εισαγωγής. Αυτό το 2009. Αλλά ταυτόχρονα αυτές οι τρεις χώρες ε, ε, μόνο ε, συνιστούσαν το 48% των ίδιων πόρων. Όπως σας είπα, η τελωνιακή δραστηριότητα μέσα στο παραδοσιακή της λειτουργία για τη συλλογή, για την ίσπραξη των ίδιων πόρων έχει επίσης σημαντικές συνέπειες για την εσωτερική αγορά. Γιατί οι ε, οικονομικοί φορείς ε, πληρώνουν λιγότερους δασμούς ή, ή, αν πληρώνουν λιγότερους δασμούς ή αν υποτιμούνται οι αξίες που δηλώνονται έχουν τελικά οικονομικό πλεονέκτημα. Το ίδιο ισχύει και για λοιπούς ε, φόρους ε, που συλλέγονται, όπως είναι ο ΦΠΑ ή η ειδικη φορη κατανάλωσης. Παρ' όλα αυτά, προκειμένου να αποφύγουμε οποιαδήποτε στρέβλωση στην εσωτερική αγορά και να εγγυθούμε ένα θεμητό ανταγωνισμό πρέπει να έχουμε αποτελεσματικούς ελέγχους που θα προσανατολίζονται στους παραδοσιακούς ίδιους πόρους επί των εισαγωγών χρησιμοποιώντας αυτοματοποιημένες τεχνικές διαχείρισης των κινδύνων συμπεριλαμβανομένων και των απλουστευμένων διαδικασιών εισαγωγής που όπως σας είπα αποτελούν σήμερα το 74% του συνόλου των εισαγωγικών διασαφήσεων. Σας ευχαριστώ. Uh, Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήμουν επικέστατος για το χρόνο αγόραυσης, ε, γιατί ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας είπατε. Έχετε δώσει και τεκμηρίωση και περάσατε ένα σαφέστατο μήνυμα και σίγουρο η συγητής θα το λάβει υπόψη του. Τώρα θα περάσουμε στις οργανώσεις που εμπλέκονται άμεσα στον τομέα των τελωνίων. Ε, και στο παρελθόν έχουμε συμμετάσχει σε συζητήσεις γιατί ευθυνόμαστε και για το θέμα της ασφάλειας των προϊόντων κυρίως σε συνδυασμό με την οδηγία για την προστασία των καταναλωτών. Καλωσορίζω τον κύριο Έλστερ που είναι σύμβουλος στην ε, Γενική Διεύθυνση ε, για τα τελωνία ε, συμμετέχετε και λειτουργείτε καθημερινά μέσα στην αγορά. Θα μας μιλήσετε για την ασφάλεια των προϊόντων. Οι διαφάνειές σας είναι έτοιμες. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι, αξιότιμοι βουλευτέ, χαίρομαι που έρχομαι σήμερα να σα μιλήσω. Θα ήθελα να σα ρίξω λίγο παγωμένο νερό, ε, ας το πω έτσι. Δεν είναι και τόσο εξυγχρονισμένα τα τελωνία μας φοβούμε, αλλά βάζουμε τα δυνατά μας. Συγγνώμη για την ψυχρολουσία, αλλά θα αρχίσω μιλώντας ε, για ε, την ασφάλεια των προϊόντων, όπως είπατε, μετά από μία σύντομη εισαγωγή θα μιλήσω για τις βασικές προκλήσεις στο τέλο παρουσίασή μου. Επόμενη διαφάνεια. Όπως ακούσαμε, ε, βασίζεται στους φόρους οποιαδήποτε τελωνιακή αρχή, αλλά όλο ένα και περισσότερο ε, χρησιμοποιούμε και νέους περιοριστικούς όρους για τη διεξαγωγή των ελέγχων, διότι όπως ακούσαμε, έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα στα τελωνία. Ε, οι δασμοί δεν είναι το βασικό μας έσοδο και βρήκαμε άλλους τομείς για να μην βαριόμαστε καθημερινά. problems for Λοιπόν, ε, μετεξελίσσεται το εμπόριο με καταιγιστικούς ρυθμούς ε, και μέσα στους νέους κανονισμούς είναι σαν να ψάχνουμε ψήλους τάχυρα. Ε, θα ήθελα να ε, μιλήσω πιο συγκεκριμένα για την ανάλυση κινδύνου και διαχείριση του ζητήματο τη ασφάλεια. Επόμενη διαφάνεια. Ποια είναι τα ζητήματα με τα οποία ασχολούνται σήμερα τα τελωνία. Βλέπετε πόσο δύσκολο είναι να αντιμετωπίζουμε ταυτόχρονα όλα αυτά τα ζητήματα. Είμαι Einstein επίσης, ξέχασα να σας το πω και έχω φτιάξει αυτό το μαθηματικό τύπο Ε, αν ε, ε, τα τελωνία συνεργαστούν καλύτερα με τις αρχές επιτήρησης αγοράς θα έχετε αποτελεσματικότητα στη Δευτέρα, enforcement και αποτελεσματική εφαρμογή του νόμου δηλαδή. Οι αρχές επιτήρησης αγοράς όταν πρέπει να αποσύρουν ένα προϊόν πρέπει να απευθυνθούν σε χίλια τουλάχιστον καταστήματα για να αποσύρουν ένα προϊόν γιατί δεν υπάρχει καλή συνεργασία με τις τελωνιακές αρχές. Οι αρχές επιτήρησης αγοράς, λοιπόν, οι MSA, ε, σε αντίθεση με τα τελωνία, λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο, 7 ώρες την εβδομάδα και ασχολούμαστε με τις εφαρμοτικές διατάξεις και όχι τους νόμους. Ε, δεν ασχολούμαστε με το αν θα απελευθερωθούν τα αγαθά σε ένα λιμένα παραδείγματο χάρη. Εμεί ε, πιο πολύ κρίνουμε την κατάσταση ω έχει και δυσαρεστούμε συχνά τα τελωνία. Ε, πρόκειται για μια νομική πρόκληση για μας. Τρόπον την ένα λεπτό να πάμε στην επόμενη διαφάνεια, διότι ο τελωνιακός ε, κωδικός κώδικας ε, και ο παλιός και ο εξυγχρονισμένος ε, είναι ατελής ως προς την ασφάλεια των προϊόντων και την προστασία των καταναλωτών. Λογικό είναι βέβαια αυτό, διότι τα τελωνία ε, δεν μπορούν να καλύψουν όλους τους περιορισμούς και τις απαγορεύσεις. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη, για να έχουμε νομική βάση για κάθε έλεγχο που διεξάγουμε, χρειαζόμαστε συνεργασία. Κάποια οργάνωση πρέπει να μας βοηθά, να μας προσφέρει, αν θέλετε, την νομική βάση για να διεξάγουμε τον έλεγχο. Αυτό είναι το χρυσό τρίγωνο, όπως το αποκαλώ εγώ, των τελωνίων. Έχουμε τη διασάφηση, γίνεται ο έλεγχος από τις αρχές επιτήρησης αγοράς, έχουμε τους διαχειριστές. Όταν λοιπόν υπάρξει, ε, διαπιστωθεί μη συμμόρφωση με τις νομοθετικές διατάξεις, ε, η αρχή επιτήρησης αγοράς ε, ανακοινώνει τα ευρήματα ε, του ελέγχου βάσει της νομοθεσίας και μας ε, ενημερώνει αν υπάρχει κάτι που βρωμάει, κάτι ύποπτο με κάποια ε, αποστολή αγαθών και κρατούνται στις αποθήκες κατόπιν τα εμπορεύματα και η διάρκεια όλης αυτής της διαδικασίας είναι τρεις μέρες για να Έχουμε μια ομάδα εμπειρογνωμών που συστάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μια ομάδα εργασία ε, για να ε, ε, ενισχυθεί η συνεργασία, να υπάρξει καλύτερη κατάρτιση και να συνεργάζονται καλύτερα οι τελωνιακέ αρχέ με τι αρχέ επιτηρήσει αγορά. Ποιο είναι το πρόβλημα, όταν έχουμε την ίδια αντίληψη περί κινδύνου. Οπότε, θα πρέπει να εξηγήσουμε στι αρχέ επιτήρηση αγοράς ε, τι ε, ε, συνιστά κίνδυνο για τα τελωνία. Δεν μιλάμε μόνο για τα εμπορεύματα, μπορεί να είναι κίνδυνος μόνο και μόνο το ότι εισέρχονται τα εμπορεύματα στην επικράτεια τη της Ένωσης. Επόμενη διαφάνεια. Προτείναμε να υπάρχει ένα γενικό κομμάτι για τις κατευθυντήριες γραμμές και ένα ειδικό κομμάτι ε, σχετικά με την ασφάλεια των προϊόντων ως προς τους ε, τελωνιακούς ελέγχους. Ε, θα έχουμε μία checklist, ένα κατάλογο για τους ελέγχους που μπορούν να χρησιμοποιούν οι αρχέ επιτήρηση αγορά όταν περνάνε στου φυσικού ελέγχου. Επίση, πληροφορίε για την ανάλυση κινδύνου που θα χρησιμοποιούν οι τελωνιακέ αρχέ. Τέλο, θα ήθελα να σα μιλήσω για τι προκλήσει που αντιμετωπίζουμε. Χρειαζόμαστε καλύτερη ανάλυση κινδύνου, καλύτερα συστήματα αποτίμησης ε, του κινδύνου. Η ασφάλεια λοιπόν των προϊόντων και η προστασία των καταναλωτών δεν έχει συνδεθεί ακόμη με τους εγκεκριμένους οικονομικούς φορείς. Δεν υπάρχουν σχετικά κριτήρια. Η εγκεκριμένη επιχείρηση λοιπόν δεν λαμβάνει σοβαρά υπόψη το θέμα της ασφάλειας. Επίσης, το πεδίο εφαρμογή του κανονισμού 765 του 2008 είναι ε, κάπως ασαφές. Δεν δίνεται απάντηση για όλους τους τομείς, γιατί και αυτό είναι επιβλαβές για τα τελωνία, διότι χρειάζονται ε, σαφείς ε, απαντήσεις. Επίσης, χρειάζεται ευαισθητοποίηση του κοινού και σταματάω εδώ. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε. Αυτά τα οποία είπατε, νομίζω πως τον είστε αρκετά σημαντικά ζητήματα, όπως ξέρετε ενδιαφερόμαστε και για την επιτήρηση της αγοράς στην Επιτροπή μας. Υπάρχει εδώ πέρα και η Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και θα ξέρετε πως ο Επίτροπος, ο κύριος Ταγιάννη, είναι επικεφαλής μιας ομάδας που θα πάνε στην Αμβέρσα, όχι στο Ρότερνταμ, την ερχόμενη εβδομάδα που νομίζω είναι το μεγαλύτερο λιμάνι κοντέινερ στην Ευρώπη για να εξετάσει αυτά τα ζητήματα οπότε νομίζω πως μπορείτε να πάτε κι εσείς μαζί του Τώρα, για να δούμε τι γίνεται με τους ανθρώπους που κάνουν τους ε, ελέγχους. Ε, με χαρά ορίζω τον ε, κύριο Ζωγράφο, ο οποίος είναι πρόεδρος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Τελωνιακών, που ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα, για να μας δώσει την δική του σκοπιά για το τι πρέπει να κάνουμε. Κύριε Ζωγράφο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ θερμά την ΙΜΚΟ για την τιμητική πρόσκληση. Φυσικά θα τοποθετηθώ ως κεντρικός εκπρόσωπος 20.000 περίπου εκτελονιστικών εταιριών τελωνιακής αντιπροσώπευσης και ως αρμόδιος κάτοχος μιας σημαντικής πολύχρονης εμπειρίας. Το διακύβευμα προκειμένου των πολιτικών αποφάσεων που ελήφθησαν και του αντίστοιχου έργου που υλοποιήθηκε συνίσταται κατά την άποψή μου στο ακόλουθο στρατηγικό τρίπτυχο. Ασφάλεια και προστασία στη διακίνηση των αγαθών, ανταγωνιστικότητα, διαφάνεια και μέγιστη οικονομία στι απαιτούμενε διαδικασίε, ασφαλή και εγγυημένη ίσπραξη των κατά δασμών και φόρων. Το πλέγμα των συστημάτων που καθιέρωσε ο κανονισμό 450 το 2008 περιγράφει και αποτυπώνει σε προωθημένο βαθμό την αντιμετώπιση, διεκπαιρέωση και λειτουργία στην καθημερινή τελωνιακή πραγματικότητα των ζητημάτων που προκύπτουν από την υιοθέτηση του προαναφερθέντος στρατηγικού τριπτύχου. Προφανώ, το μόνο που μέχρι στιγμή δεν ικανοποίησε είναι η εναρμόνιση του βηματισμού ανάμεσα στον κάθε εθνικό και διεθνή χώρο του εμπορίου και τον χώρο, τεχνικά και θεσμικά, των τελωνιακών και άλλων υπηρεσιών που εκπροσωπούν οι εθνικές διοικήσεις και τα κεντρικά ευρωπαϊκά όργανα. Οι πρώτοι ζητούν κυρίως ταχύτητα, αντιγραφειοκρατική νοοτροπία και αποτελεσματική ανταγωνιστικότητα. Οι υπηρεσίες όμως πέραν αυτών πρέπει να μεριμνούν και για την σύνομη και αποτελεσματική λειτουργία των διαδικασιών που στοχεύουν στην ίσπραξη των προβλεπωμένων φόρων και την εξάλληψη της απάτης και του λαθρεμπορίου. Αυτό προφανέστατα είναι το νέο διακύβευμα ο νέο στόχο, τι λεπτέ πλευρέ του οποίου πρέπει να εντοπίσουμε και να εξοραίσουμε μέσα στα επόμενα χρόνια. Συμφωνούμε και προσυπογράφουμε τη θέση του Επιτρόπου κυρίου Σεμέτα ότι δεν πρέπει να ασχοληθούμε με τα θεμέλια και τι βασικέ κατευθύνσει που ορίζονται από τι διατάξει του κανονισμού 450. Γιατί θα χάσουμε πολύτιμο χρόνο και θα αποχρωματίσουμε τον χρήσιμο χαρακτήρα του. Αντίθετα, πρέπει να εισφέρουμε σε ιδέε που θα ενισχύσουν μέσω των ηλεκτρονικών προσαρμογών την εφαρμογή του. Ο εμπορικό κόσμο, από τη μια πλευρά, και οι τελωνιακέ διοικήσει, από την άλλη, προσμένουν τη μέγιστη υπευθυνότητα και προβλεπτικότητα. Όταν φτάσουμε στο τέλο, θα πρέπει να εγγυημένα να έχουμε πετύχει του στρατηγικού μα στόχου, έτσι όπω αυτοί ετέθησαν το 2008 από το γράμμα και το πνεύμα τη τελική απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου. Οι στόχοι αυτοί, πέραν των άλλων, θα πρέπει και μέσω των ελέγχων να μεριμνούν για τα ακόλουθα. Ασφάλεια και προστασία. Οπωσδήποτε πρέπει να εγγυηθούμε τα υψηλότερα επίπεδα τόσο της ασφάλειας κατά τη διακίνηση των εμπορευμάτων, κυρίως απαγορευμένων υλών, όπλων κτλ., όσο και της προστασίας των πολιτών σε θέματα υγείας σχετικά με τα είδη διατροφής και ευρεία κατανάλωσης. Επιβάλλεται αυστηρή φροντίδα και ειδική μέρημνα για τήρηση των νόμων που απαιτητικά διέπουν τη σύγχρονη διαβίωση. Υγιής ανταγωνιστικότητα και οικονομία. Είναι κανόνε απαράβατοι και σεβαστοί για να μπορέσουν εμπόριο και δημόσια διοίκηση να οικοδομήσουν ένα βιώσιμο και ισχυρό μέλλον για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει κάθε ενέργεια που του υπηρετεί να ενισχύεται και κάθε συμπλεγματική, αναχρονιστική σκέψη να απομακρύνεται. Εγγυημένη ίσπραξη δασμών και φόρων. Η ύπαρξη ενό καλώ νοούμενου δημοσιονομικού φόβου θεωρώ ότι είναι το background και η προπόθεση στο πνεύμα των οποίων εξυπηρετούνται θετικά οι αποτελεσματικοί έλεγχοι. Φυσικά δεν θέλω ούτε καν να υπονοήσω μεσαιωνικού επίπεδου συστήματα και νοοτροπίε. Αντίθετα, Αναφέρομαι σε έξυπνε και αποτελεσματικέ μεθόδου, όπου η εμπειρία, η γνώση και ο εξοπλισμό των σύγχρονων τελωνιακών υπηρεσιών διασφαλίζουν. Η φράση τη Ταξούντ «Τα τελωνία βλέπουν αυτό που εσείς δεν βλέπετε» πιστεύω ότι δίνει με πολιτισμένο και σύγχρονο τρόπο το νόημα και τις μεθόδους λειτουργίας των σημερινών ευρωπαϊκών τελωνίων. Ταυτόχρονα, η διαρκή συνεργασία των εθνικών τελωνιακών υπηρεσιών και η χρήσιμη συνεχής πληροφόρηση με ανταλλαγή και διασταύρωση ηλεκτρονικών μηνυμάτων θα αποτελέσουν κορυφαίο και πλήρως αξιοποιήσιμο μέσον έγκαιρου εντοπισμού και αφοπλισμού όσων προσπαθήσουν να εξαπατήσουν τις αρχές υποκλέπτοντας δασμούς και φόρους και περιορίζοντας τους κοινωνικούς πόρους υπό των Ευρωπαίων πολιτών. Ίσως θα ήταν χρήσιμο και αποδοτικό να δημιουργηθεί ένας λεπτομεριακός ηλεκτρονικός χάρτης των τελωνιακών κινήσεων στην Ευρώπη από αυτόν θα ξεκινούν και σε αυτόν θα καταλήγουν σαν δρόμοι αμοιβαία προσέγγισης και επικοινωνίας όλα τα στοιχεία όλων των τελωνιακών πράξεων που θα εκτελούνται καθημερινά στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένας κεντρικός εγκέφαλος μνήμης και πληροφόρησης θα καθοδηγεί και θα γνωστοποιεί σε κάθε αρμόδιο όλες τις φάσεις των κινήσεων των εμπορευματικών συναλλαγών μέχρι την ίσπραξη των δασμών και φόρων. Θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι τα πρόσωπα που θα κάνουν χρήση των συστημάτων πρώτον έχουν τι τεχνικέ και επαγγελματικέ γνώσει για να διεκπαιρεώνουν με ορθότητα και φερεγγιότητα τι θελωνιακέ εργασίε. Και δεύτερον, θα συμβάλλουν με τα ηλεκτρονικά του μέσα στην διεισδυτική και ξεκάθαρη ολοκλήρωση των ελέγχων. Η σημερινή ανασταλτικότητα για οικειοποίηση τη ιδιότητα του ΑΕΟ δεν πρέπει να αποθαρρύνει και να απογοητεύει. Πιθανότατα δεν έχει γίνει ευρύτερα αντιληπτό ο θεσμικό του ρόλο και αυτό μπορεί να οφείλεται στο δυσνόητο περιεχόμενό του πρέπει να εκλαϊκευθεί και να διαφημιστεί ώστε να προσελκύσει ενδιαφερόμενους με γρηγορότερου ρυθμούς. Ο συμπληρωματικό τη τελωνιακή δραστηριότητα ρόλο των διαπιστευμένων τελωνιακών αντιπροσώπων, συμβαδίζοντα σε θεσμικέ και λοιπέ προποθέσει με αυτόν του ΑΕΟ, εγκεκριμένου οικονομικού φορέα, αποτελεί ενισχυμένη εγγύηση και προστιθέμενη αξία στην προσπάθεια των αρχών για εύρυθμη αντιγραφειοκρατική και αποδοτική λειτουργία ίσπραξη των δασμών και φόρων σε κάθε γωνιά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό η αναβαθμισμένη και θεσμοθετημένη δραστηριοποίησή του θα αποβεί δυνατό εργαλείο προ αξιοποίηση. Η, η εφαρμοσμένη ηλεκτρονική του κατάρτιση πρέπει να χρησιμοποιηθεί από τι τελωνιακέ αρχέ σαν μια διαρκή online πρόσβαση που σαν καθρέπτη θα διευκολύνει του ελέγχου ακόμα και μετά την παρέλευση σημαντικού χρονικού διαστήματος. Το καθεστώς της αυτορύθμισης, σε συνδυασμό με τη διαρκώς ανοιχτή τελωνιακή πρόσβαση, αποτελεί εγγύηση για εξαφάνιση της απάτης και της φοροδιαφυγής. Για να λειτουργήσει όμως αυτό το σύστημα, θα πρέπει οι τελωνιακοί αντιπρόσωποι που θα το εξασφαλίσουν να διαπιστευτούν με αυστηρές προϋποθέσεις. Οι κωδικοί κλειδιά που θα τους δοθούν θα ανοίγουν επίσης τις πόρτες μόνο στα αρμόδια πρόσωπα που έχουν θεσμοθετηθεί να διεκπεραιώνουν ελέγχους. Τέλος, προσαρμοσμένα ηλεκτρονικά συστήματα μπορούν να υλοποιούν αυτή την αμοιβαία και χρήσιμη επικοινωνία. Ο εξχρονισμένο κοινοτικό τελωνιακό κώδικα και το σημερινό σχέδιο διατάξεων εφαρμογή του πρέπει να είναι η αποτύπωση τη συγκερασμένη βούληση εμπειρογνωμόνων και εμπορικού κόσμου. Α δουλέψουμε και συνεργαστούμε για μια ενωμένη Ευρώπη, ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο, ακμάζουσα σε ανθρώπινε υπηρεσίε και προσφορέ και ευημερούσα σε οικονομικό και βιωτικό επίπεδο. Για την καθιέρωση και εφαρμογή των προαναφερομένων, ο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήταν και θα παραμείνει ιστορικό. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Ζωγράφο. Θα προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις σας, στις προσδοκίες σας. Λοιπόν, όπως είπα, περνάμε κατευθείαν στους επόμενους τρεις ομιλητές και μετά θα γίνει μια κάποια γενική συζήτηση με τους βουλευτές γιατί νομίζω πως υπάρχει ένα κοινό νήμα που διατρέχει αυτά τα ζητήματα και είναι η σημασία της συνεργασίας θα νομίζω πως θα μπορέσουν να μιλήσουν και οι επόμενοι ομιλητές λίγο παραπάνω, αλλά μείνετε παρακαλώ εντός των 7 λεπτών. Έχουμε τον κύριο Φρανκ Χάιμαν, υπεύθυνο για τις σχέσεις με το εμπόριο από τα Ολλανδικά Τελωνία και Ρισπέντιφ, ε, υποδιευθυντής πολιτικής ε, ειδικών φόρων κατανάλωσης ε, και διαδικασιών και Frank Calvert από την Microsoft θα μας μιλήσει για την τεχνολογία καθώς είναι αρμόδιος για την τεχνολογική στρατηγική και συχνά μιλήσαμε για τον εξυγχρονισμό, ας ακούσουμε και από αυτή την σκοπιά. ξεκινήσουμε τον κύριο Χάιμαν. η διαφάνειες σας όπως βλέπετε προβάλλονται ήδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας δίνετε την ευκαιρία να καταθέσουμε την άποψή μας επί του θέματος. Πρώτα απ' όλα για την ε, συνεργασία, θα μιλάτε για συνεργασία μεταξύ των τελωνιακών αρχών. Μπορεί να είμαι σύντομο. Τα τελωνία στην Ευρώπη είναι μια μεγάλη οικογένεια. Καμία άλλη υπηρεσία νομίζω δεν ε, επικοινωνεί τόσο εύκολα μεταξύ 27 κρατών μελών όσο τα τελωνία. Και υποστηρίζονται βεβαίως και από το πρόγραμμα της Κομισιόν Τελωνία 2030 και έτσι έρχεται όλο και πιο κοντά η οικογένειά μας και νομίζω πως η συνάδελφος από το Ηνωμένο Βασίλειο θα αναφέρει κάποια πράγματα για την συνεργασία με το εμπόριο, οπότε εγώ θα σας πω ποια είναι η κατάσταση στις προτάσεις που έχουμε. μιλήσαμε για τους συγκεκριμένους φορείς, ακούστηκαν ήδη πολλά. Πρώτα απ' όλα πρέπει να δούμε τους στόχους του εξυγχρονισμού. Θέλαμε μια απλοποίηση των τελωνιακών διαδικασιών και της νομοθεσίας, να γίνουν ε, να υπάρχουν απλοποιήσεις για τους εμπόρους, να διευκολύνουμε το νόμιμο εμπόριο, να μειωθεί το διοικητικό βάρος, να αυξηθεί η ασφάλεια ε, και να γίνει πιο ανταγωνιστική η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τώρα, εάν δείτε τις προτάσεις τις οποίες έχουμε, πράγματι υπάρχει ένα σύστημα εγκεκριμένων φορέων. Τα δε ωφέλη του, όπως υπόθηκε, είναι κάπως περιορισμένα. Ε, ακόμα και αν το συγκρίνετε εδώ και δύο χρόνια τι έχει γίνει, πρέπει για απλοποιημένες διαδικασίες να εκπληρώσει κάποια κριτήρια ο έμπορος, αλλά πριν δεν χρειαζόταν αυτό, οπότε για κάποιους ε, εμπόρους ε, το καθεστώς συγκεκριμένου ε, φορέα θεωρείται ένα παραπάνω εμπόδιο αντί για μια διευκόλυνση. Και αν δούμε το τι υπάρχει στον εξυγχρονισμένο τελωνιακό κώδικα, αν δούμε το σύστημα διαχείρισης εγγυήσεων για να παρακολουθούμε πανευρωπαϊκά αυτέ για να υπάρχουν ήδη οι πόροι της Ένωσης αυτή τη στιγμή υπάρχει τελωνιακή επιτήρηση το ερώτημα το οποίο έχουμε είναι πως ε, θα χρειαστεί ένα μεγάλο πληροφοριακό σύστημα το θέμα είναι υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Υπάρχουν τόσοι πολλοί ήδη πόροι που δεν μπορούν να συλληγούν λόγω του τωρινού συστήματος εγγυήσεων. Εφαρμόζουμε το σύστημα αυτό των εγγυήσεων πριν από λίγα χρόνια για τα διερχόμενα εμπορεύματα και για τις υπόλοιπες διαδικασίες θεωρούμε πως δεν υπάρχει τέτοιο μεγάλο πρόβλημα ότι θα πρέπει να γίνει μια καλή μελέτη αξιολόγησης αντικτύπου. Κατόπιν εξετάσαμε άλλη μια πρόταση του εξυγχρονισμένου συστήματος για την προσωρινή αποθήκευση. Έχουμε αυτή τη στιγμή απλές διαδικασίες εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να έρθουν τα αγαθά. Δηλαδή αυτή τη στιγμή φτάνει ένα αεροπλάνο, έχουμε μια εύκολη διαδικασία προσωρινής αποθήκευσης για να φύγουν τα αγαθά από το αεροπλάνο ή το πλοίο και να πάνε σε μια προσωρινή αποθήκευση. Γιατί, Γιατί τα μέσα μεταφοράς, πλοία και αεροπλάνα πρέπει να κινούνται και δεν μπορούν να παραμείνουν επιτόπου αγκυροβολημένα για να τελειώσουν τελωνιακές διαδικασίες. Με τις τωρινές προτάσεις βλέπουμε πως η προσωρινή αποθήκευση γίνεται τελωνιακή διαδικασία και αυτό βεβαίως επιβάλλει πολύ διοικητικό βάρος στο εμπόριο και θα μπορούσε να μειώσει την ταχύτητα εισερχόμενης και εξερχόμενης κυκλοφορίας. Και αυτό το οποίο βλέπουμε είναι πως υπάρχει ένα ασφαλές πλαίσιο διαδικασιών που υιοθετήθηκε από τον ΠΟΕ πριν από λίγα χρόνια, αλλά στον εξυγχρονισμένο τελωνιακό κώδικα δεν βλέπουμε να υπάρχει ευθυγράμμιση με τους στόχους του πλαισίου αυτού. Δηλαδή, να γνωρίζουμε π.χ. τα ευρήματα τρίτων τελωνιακών διοικήσεων από τρίτες χώρες Ε, θεωρούν πως υπάρχουν ευρωπαϊκά εγρήματα. Οπότε θα μπορούσαμε να έχουμε μια κάποια ευθυγράμμιση. Και υπάρχουν και κανόνε όπως σας είπα, ασφάλεια από κακόβλε ενέργειες και ατυχήματα που είναι απολύτως απαραίτητα. Αλλά αυτό το οποίο αντιμετωπίζουμε είναι πως υπάρχει μεγάλο βάρος που επιβάλλεται στο εμπόριο για να δίνει διάφορα δεδομένα και μιλάμε για το 100% του εισερχόμενου εμπορίου ενώ κατ' ουσίαν αναζητούμε το 0,1% που είναι το παράνομο εμπόριο. Οπότε θα μπορούσαμε να έχουμε μια διαφορετική προσέγγιση. Αυτό το οποίο βλέπουμε επίσης είναι πως οι προτάσεις αυτές τυποποιούν τα πάντα. Η τυποποίηση είναι καλή για να συνεργάζονται τα ευρωπαϊκά τελωνία, αλλά υπάρχουν διαφορετικά μέσα μεταφορές. Ο κόσμος των πλοίων είναι διαφορετικός από τα αεροπλάνα και τα φορτηγά. Και η θέση των χωρών είναι διαφορετική. Στην Ολλανδία, όπως είπατε, είπατε θα πάτε στο Ρότερνταμ. Το Ρότερνταμ ε, μετακινεί εκατομμύρια εμπορευματοκιβώτια και είναι κάτι το λίγο διαφορετικό από ένα φυλάκιο χερσαίων συνόρων που μπαίνουν λίγα φορτηγά τη μέρα. Οπότε όταν θα τυποποιήσουμε τον εξυγχρονισμένο τελωνιακό κώδικα θα πρέπει να αντιμετωπίσει Όλε αυτέ τι διαφορετικέ καταστάσει και θα τι αντιμετωπίζει ω μία. Οπότε εμεί έχουμε μια οποτε εμει εχουμε εμπειρία για το πώ θα αντιμετωπίζουμε του μεγάλου όγκους εμπορευμάτων που πρέπει να μετακινηθούν γρήγορα. Και αυτό το οποίο θα θέλαμε είναι βεβαίω να δούμε αυτέ τι συγκεκριμένε καταστάσεις. Τώρα για τα ηλεκτρονικά τελωνία. Αυτή τη στιγμή έχουμε 27 διαφορετικά συστήματα, μορφές δεδομένων και ε, σημεία πρόσβασης και βεβαίως επενδύουν εκατομμύρια τα τελωνία. Χρειάζεται λοιπόν μια πιο έξυπνη προσέγγιση για να μην έχουμε υπερβολικές επενδύσεις σε πληροφορική και ε, ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα για να ξέρουμε το τι θα θέλουμε να επενδύσουμε και εμείς και ε, οι εμπορευόμενοι. Τώρα κοιτάζοντας ε, τους ε, μη φορολογικούς κανόνες. Δυστυχώς έχουμε μείνει στο 2003 όταν λέγαμε πως θέλουμε να έχουμε μόνο ηλεκτρονικά μηνύματα και όμως έχουμε οδηγίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ασχολούνται με συστήματα που βασίζονται στο χαρτί. Θέλουμε καλύτερη επικοινωνία. Ε, λέτε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά της, αλλά όχι να ανταγωνιζόμαστε στο εσωτερικό, θα πρέπει να ενωθούμε οι Γενικές διευθύνσει Κομισιών, τα κράτη-μέλη και εσεί. Ε, Θέλουμε λοιπόν μια καινοτόμο προσέγγιση, περισσότερο ανταγωνισμό για το νόμιμο εμπόριο, για να βρεθεί μια καλή βάση για νέες ιδέες ε, τελωνιακών διευκολύσεων, π.χ. κεντρικό κεντρικός και να έχουμε καλύτερες καινοτόμες ιδέες, ε, πρωτοποριακές, ε, για να δούμε βεβαίως ε, τι βρίσκεται μέσα στο κάθε κυβότιο. Γιατί αυτός ο οποίος ξέρει τι βρίσκεται μέσα στο κάθε κυβότιο είναι ο εξαγωγέας και εκεί πέρα ακριβώς θα πρέπει να επικεντρωθεί η νομοθεσία. Έργα δε όπως το πρόγραμμα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μας δίνουν την ευκαιρία με χρηματοδότηση, να κάνουμε κοινή έρευνα με του εμπορευόμενου για τι νέε δυνατότητε. και στην τελευταία διαφάνεια βλέπετε πω, αν δεν αλλάξουμε τώρα, βλέπετε ποιο θα μπορούσε να είναι το μέλλον. Αναμένουμε να αυξηθεί ε, να αυξηθούν οι διευκολύνσει με τον εξυγχρονισμένο του ελληνικού κώδικα. Αλλά αν δεν γίνει αυτό, θα μπορούσαμε να καταλήξουμε με χαμηλότερο επίπεδο διευκολύνσεων από ό,τι αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ για την προσοχή σα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Χαϊμάν. Αισθάνομαι κάπως στεναχωρημένος που έχασα ένα μέρος της παρουσίασή σας, αλλά είμαι σίγουρος ότι οι συγγητές μας παρακολούθησαν με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Λοιπόν, να περάσουμε στην κυρία Σπέντιφ για να μας παρουσιάσει τη δική της προοπτική για την ενδυνάμωση του εσωτερικού συντονισμού. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε. Εγώ έχω στείλει την παρουσίασή μου και ο τίτλος είναι Why Bother, γιατί να ασχολούμαστε, γιατί δεν θέλω να κάνουμε ε, κάποιες ε, υποθέσεις που να τις θεωρούμε δεδομένες. Θα κάνω κάποιες παρατηρήσεις για το σημερινό περιβάλλον και ελπίζω ότι ε, θα στείλω ένα μήνυμα που θα λάβετε για το πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε τα επόμενα χρόνια. Λοιπόν, εδώ βλέπετε παρόμοια σημεία με αυτά που είπαν και προλαλήσατε. Έχουμε τους διάφορους κινδύνους ε, που αντιμετωπίζουν οι τελωνιακές δικήσεις ε, και βλέπετε ότι πρόκειται για μια επιχείρηση που πρέπει να διαχειρίζεται κινδύνους. Αυτό είναι τα τελωνία. Εδώ έχουμε φορολογικούς, οικονομικούς, κοινωνικούς ε, και φυσικούς κινδύνους αλλά από ό,τι γνωρίζετε δεν είναι εύκολο ε, να το υλοποιήσουμε όλο αυτό, τους ελέγχους. Περισσότερο είναι τέχνη παρά επιστήμη. Εδώ μιλάμε για διακίνηση αγαθών, δεν μιλάμε για κυκλοφορία ανθρώπων. Πολύ συχνά εξηγούμε ότι μας ενδιαφέρουν τα αγαθά και όχι οι άνθρωποι και βέβαια έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους γιατί αυτοί διακινούν τα αγαθά, όχι για κανέναν άλλο λόγο. Αλλά αν ε, καταστήσουμε αυτό σαφές, νομίζω ότι το επόμενο σημείο της παρουσίασης έχει να κάνει ε, με τις εντάσεις που μπορεί να δημιουργήσουν αυτοί οι κίνδυνοι για τα τελωνία Νομίζω ότι ο κύριος Καστρισιανάκης ανέφερε τη θέμα της έντασης μεταξύ της διευκόλυνσης και της ε, ασφάλειας. Νομίζω ότι αυτά τα δύο τα συμπεριλαμβάνουμε όλο και περισσότερο στις διαδικασίες έτσι ώστε να μπορούν να συνεχίσουν ε, την, ε, το εμπόριο οι επιχειρήσεις και εμείς να μπορούμε να προβούμε στον έλεγχο. Λοιπόν, το επόμενο στοιχείο που θέλω να αναφέρω είναι πολιτικού χαρακτήρα ε, βλέπουμε εδώ πώς συμπεριλαμβάνονται διάφορα υπουργεία ε, και ποιος μπορεί να πει ποιο είναι το υπουργείο που έχει τη μεγαλύτερη προτεραιότητα. Σε αυτή τη διαφάνεια βλέπετε το θέμα των διασαφήσεων. Εδώ βλέπετε ότι μέσω ενό και μόνο διοικητικού εγγράφου προστατεύουμε τα συμφέροντα όλων αυτών των φορέων. Εμείς δηλαδή προσπαθούμε να συντονίσουμε όλα αυτά τα συμφέροντα στη διέλευση των συνόρων. Επίσης συνεργαζόμαστε πολύ στενά με άλλες τελωνιακές αρχές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τελωνίων, το να σκεφτόμαστε παγκόσμια είναι στο αίμα μα. Ε, Επίση, ενδιαφερόμαστε τι συμβαίνει και στον ΠΟΕ, στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και συνεργαζόμαστε αποτελεσματικά μαζί του. Τώρα, βλέπετε εδώ τον όρο business, επιχειρήσει με παγιά γράμματα. Γιατί νομίζω ότι εδώ πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σοβαροί. Αν θέλουμε να προωθήσουμε το διεθνέ εμπορίο και τον ανταγωνισμό στην Ευρώπη, πρέπει να είμαστε πολύ ε, πιο ανοιχτοί στη συνεργασία με τι επιχειρήσει και να τι εμπλέκουμε στο πώ ε, σχεδιάζουμε το μελλοντικό επιχειρησιακό μας μοντέλο. Λοιπόν, θα, για να, να, αναφερθώ και σε μια μελέτη που έγινε σήμερα. Ε, έλεγε η μελέτη αυτή ότι είναι εξυγχρονισμένη τα τελωνία, αλλά δεν νομίζω ότι έχουμε φτάσει στον εξυγχρονισμό που θέλουμε. Πρέπει να δούμε τι κάνουμε σήμερα. Ε, νομίζω ότι πρέπει να αναπτύξουμε μία μεγαλύτερη αμοιβαία κατανόηση και να συνεργαστούμε. Πρέπει οι κυβερνητικές αρχές να προσπαθήσουν να κεφαλοποιήσουν όσα διαθέτουν ήδη. Πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών και μεγαλύτερη ανταλλαγή διάφορων δεξιοτήτων δεν θα πρέπει να δαπανούμε χρόνο για τις οργανωτικές δομές ούτε τα τελωνία να κάνουν το ίδιο πράγμα σε 27 κρατημέλη. Ε, εδώ δεν θέλουμε να πούμε ότι πρέπει να γίνονται τέτοια πράγματα σε μια χώρα, αλλά θέλουμε να εργαστούμε για να καταλήξουμε σε πρότυπα αριστεία και για να κατανοήσουμε τα μοναδικά μα περιβάλλοντα και να κεφαλοποιήσουμε επί αυτή τη ποικιλομορφία. Τώρα, το μήνυμα εδώ είναι Έχουμε σχέση με τις επιχειρήσεις, μας αρέσει να συνομιλούμε με τις επιχειρήσεις, αλλά ότι μπορούμε να τα πάμε καλύτερα. Θέλουμε μια προσέγγιση από την οποία όλοι θα βγαίνουν κερδισμένοι και το μήνυμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι να σα ζητήσουμε βοήθεια. Θεωρούμε ότι μπορείτε να μας βοηθήσετε ε, στο να συμμετέχουμε και εμείς στη χάραξη πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, υπάρχουν ε, ε, ε, ουσιαστικά πάρα πολύ έλεγχοι εγγράφων στα σύνορα. Αυτό μας καθυστερεί. Ε, κατανοούμε τι καθοδηγεί τις διάφορες πολιτικές που μας ζητούν να το κάνουν αυτό αλλά θέλουμε να συζητήσουμε σήμερα, να προσπαθήσετε κι εσείς να κατανοήσετε τι κάνουν τα τελωνία. Είναι μοναδικό το καθήκον μας, έτσι λοιπόν θα ήθελα να αναγνωρίσετε το ρόλο μας. Υποστηρίζουμε τις νόμιμες ε, επιχειρήσεις, αλλά μας αρέσει να πιάνουμε και τους κακούς. Σας ευχαριστώ. Well, Σας ευχαριστούμε. Είτε ήσασταν σαφέστατοι βρήκατε και την ευκαιρία να μας υπενθυμίσετε τον απότερο στόχο της ακρόασης. Ξ' των συναδέλφων μπορώ να σας πω ότι συμμετείχα στι έρευνε που κάναμε σε διάφορα μέρη του κόσμου, μεταξύ των οποίων και η Κίνα και η Ινδία και στην ε, Τσεχία. Νομίζω ότι είναι όντως ε, πολύ σύνθετο το πρόβλημα. Και τα θέματα συνεργασία που γύρεται είναι εξαιρετικά εύστοχα και σίγουρα θα τα σχολιάσει και ο εισηγητή μα. Θα ήθελα να σα θυμίσω ότι πρόκειται για πολιτική πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αλλιώ δεν θα ήμασταν υποχρεωμένοι να το κάνουμε. Αυτό, ε, είναι, πρόκειται για πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου. Αλλιώ αυτό που κάνουμε είναι να εξετάζουμε νομοθετικέ ε, πράξει. Και εσεί ε, από την πλευρά σα διαδραματίστε το ρόλο σα στα πλαίσια τη διαβούλευση. Α περάσουμε τώρα στην τεχνολογία. Με χαρά συνήθω έχουμε κάποιον από την Microsoft. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχει η συνέλευση για την ψηφιακή κοινωνία που διεξάγεται αυτή τη στιγμή ε, και αυτό το λέω για να καταδείξω ότι σε οποιαδήποτε οργάνωση, οποιοδήποτε μέρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, το θέμα τη τεχνολογία έχει ιδιαίτερη σημασία. Ο κύριο Κάλιβαρ θα κάνει την τελευταία παρουσίαση σημερινή ακρόαση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμοι βουλευτέ, κυρίε και κύριοι, ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να σα προσφωνήσω σήμερα. Α δούμε το εμπόριο από την οπτική γωνία τη ε, Microsoft, ε, μια διεθνή εταιρεία. Βασιζόμαστε λοιπόν στο εμπόριο στη συνεργασία. Οι αγοραστές ε, βρίσκουν, οι πολιτές βρίσκουν τους αγοραστές και γίνονται οι εισαγωγέ κάθετο εξαγωγέ Μέσα από διοικητικέ, οικονομικέ, εμπορικές διαδικασίες. Αν δούμε τα πράγματα από την πλευρά τη πληροφορική. όλα αυτά είναι διαφορετικά συστήματα. Όλες οι οργανώσεις έχουν δικό του σύστημα και το σύστημα πρέπει να συνάζει με τον κανονισμό και θα πρέπει λοιπόν να συμμορφώνονται όλοι με τις νομοθετικές ε, διατάξεις. Ε, τώρα σε παγκόσμιο επίπεδο η Microsoft καλείται να λάβει υπόψη όλα αυτά τα στοιχεία και από ρυθμιστικής, κανονιστικής πλευράς όπως είπε και η συνάδελφός μου εδώ ε, Τίδονται διάφορα ζητήματα. Ο εξυγχρονισμένο τελωνιακό κώδικα, τα διάφορα συστήματα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, μιλήσαμε για τον εγκεκριμένο οικονομικό φορέα. Υπάρχουν και άλλε και άλλοι κυβερνητικοί φορεί που έχουν άλλου κανονισμού και εμεί οφείλουμε να συμμορφωθούμε. Τα συστήματα πληροφορική διευκολύνουν τη ροή των δεδομένων την επαναχρησιμοποίηση δεδομένων ανάμεσα σε διαφορετικά συστήματα. Μιλήσαμε για τα συστήματα ανάλυση κινδύνου. Κοιτάξτε, το πλαίσιο ανάλυση κινδύνου είναι ένα σύστημα που θα μπορούσε να ε, επωφεληθεί τα μάλλον από τι νέε διατάξει ε, για να υπάρχει καλύτερη ροή των πληροφοριών και καλύτερη επαναχρησιμοποίησή του. Ε, λοιπόν, εμεί στέλνουμε εμπορεύματα σε 147 διαφορετικέ χώρε, υλικό καθώ και λογισμικά πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε να προστατεύουμε και τα περιουσιακά μας στοιχεία. Ε, έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό για τις επιχειρήσεις ε, και ε, δηλαδή τα συστήματα πληροφορικής πρέπει να συμβάλλουν τόσο ώστε να προστατεύονται και τα πνευματικά δικαιώματα των προϊόντων που εμπορευόμαστε. Ε, το σημαντικό είναι να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε, ε, να επικοινωνήσουν μάλλον μεταξύ τους όλα τα υφιστάμενα συστήματα πληροφορικής, όχι μόνο μέσα στην Ευρώπη αλλά και ανά τον κόσμο. Εμείς έχουμε δικά μας συστήματα, αλλά έχουμε δημιουργήσει και ένα τμήμα εμπορίου μέσα στην Microsoft ε, που θεωρεί ότι η συνεργασία είναι ακρογωνίως λήθος της λειτουργίας της Microsoft. Ερχόμαστε σε επαφή με όλες τις τελωνιακές διοικήσεις, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, εργαζόμαστε στενά με οργανισμούς όπως ο Παγκόσμιο Οργανισμός ε, Τελωνίων και κάνουμε τα πάντα ώστε τα συστήματα πληροφορική να συνάδουν ε, με τους συγκεκριμένου κανονισμούς και με τις απαιτήσει από πλευρά εμπορευομένων, από τη δική μα δηλαδή, και από πλευρά των τελωνιακών αρχών. Αποστέλουμε εμπορεύματα σε ολόκληρο τον κόσμο αφημερών ε, και χρειαζόμαστε έγγραφα σε όλε τι πιθανέ γλώσσε. Τώρα, σε σχέση με τι εξελίξει στην Ευρώπη και τον εξυγχρονισμένο κώδικα, ε, έχουμε εντοπίσει διάφορα εμπόδια που ανακύπτουν και διάφορε λύσει που θα μπορούσαν να διευκολύνουν την ευχερέστερη χρήση ε, των νέων τεχνολογιών και των συστημάτων πληροφορική. Πρώτον, και νομίζω ότι το ανέφεραν ε, οι περισσότεροι αμιλητές, ε, το πρόβλημα είναι η διαφορά των συστημάτων. Δηλαδή, για την διασάφηση εισαγωγή στη Γερμανία έχουμε διαφορετικό σύστημα ΦΠΑ. Οπότε, από πλευρά διατυπώσεων υπάρχει ήδη πρόβλημα γιατί είναι διαφορετικέ οι διασαφήσει. Τώρα, από πλευρά τεχνολογία υπάρχει επίση πρόβλημα δεν είναι διαλειτουργικά τα συστήματα πληροφορική. Ε, δηλαδή, από την πλευρά του εμπορευομένου θα πρέπει να μπορέσετε να μπείτε και να λειτουργήσετε βάσει ενός συστήματος που όμως δεν είναι διαλειτουργικό με το δικό σας. Ε, νομίζω ότι σε αυτό κρύβεται και η λύση. Ε, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τελωνίων έχει κάνει κάποια θετικά βήματα και έχει αναλάβει πρωτοβουλίες όπω ε, το ενιαίο διοικητικό έγγραφο, το, την ευρωπαϊκή απόδειξη. Όλα αυτά μα βοηθούν ούτω ώστε να επιτύχουμε καλύτερη διαλειτουργικότητα των συστημάτων πληροφορική και να γίνεται καλύτερα και αποτελεσματικότερα η ανταλλαγή των πληροφοριών ανάμεσα στι τελωνιακέ αρχέ και τι επιχειρήσει. Η ολοκλήρωση του συστήματο είναι εξαιρετικά δραπανηρή. Σε ορισμένες σε ορισμένε χώρε χρειαζόμαστε συγκεκριμένη πραγματογνωμοσύνη και λογισμικά για να μπορέσουμε να εμπορευτούμε με μια χώρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ω προ τη συνεργασία, ε, ήδη έχουμε μπλακεί στη συζήτηση για τον εξυγχρονισμένο κώδικα και έχουμε καταθέσει τι απόψει μα, αλλά όπω και οι λοιποί ομιλητέ, θα θέλαμε περισσότερε ευκαιρίε ε, για να σα τροφοδοτούμε με περισσότερε πληροφορίε, ε, για να δούμε τι περιμένετε από του εμπορικού φορεί στα πλαίσια του εξυγχρονισμένου κώδικα, να αντιστρέψουμε την κατάσταση, ποια είναι τα θετικά στοιχεία χάρη σε ποια στοιχεία μπορούμε να προχωρήσουμε και ε, τι μπορούμε να διευκολύνουμε με τον εξυγχρονισμένο κώδικα. Ο στόχο είναι να έχουμε ε, ένα νέο ηλεκτρονικό τελωνιακό περιβάλλον ε, που θα διευκολύνει τη συνεργασία. Η εναρμόνιση και η τυποποίηση των δεδομένων και των διατυπώσεων έχει ιδιαίτερη σημασία. Σα μίλησα ήδη για το module για τα δεδομένα του Παγκοσμίου Οργανισμού Τελωνίων. πολύ ενδιαφέρουσα λύση. Από πλευρά εμπορευμένων, αυτό που θέλουμε να αποκομίσουμε εμεί είναι το εξή. Με ανταγωνιστικό τρόπο να πορευόμαστε στην περιοχή της Ευρώπης με διαφάνεια, με ασφάλεια όπως ακούσαμε από τους ομιλητές μας. Ανησυχούν πολύ φυσικά τα πνευματικά δικαιώματα και η προστασία τους, αλλά το πλέον σημαντικό για μας είναι η μείωση του κόστους, η περικοπή του κόστους, διότι θέλουμε να εμπορευόμαστε με χαμηλό κόστος και χρησιμοποιώντας ένα διαλειτουργικό σύστημα. Ευελιξία επίση. Δεν πιστεύουμε ότι όλε οι λύσει κάνουν για όλου, και το είπε και ένα προλαλή σα ότι υπάρχουν διαφορετικά μεγέθη επιχειρήσεων στα κράτη-μέλη, πολύ διαφορετικέ ανάγκε, οπότε το ίδιο το τελωνιακό σύστημα για ένα, μια περίκλειστη μικρή χώρα δεν μπορεί να λειτουργήσει για μια μεγαλύτερη χώρα και το ίδιο ισχύει και για του εμπόρου. Ε, μιλήσατε για τι μικρομεσαίες επιχειρήσει. Οι μεγάλοι διεθνείς ε, εμπορικοί φορεί έχουν διαφορετικέ ε, τεχνολογικέ ανάγκε και διαφορετικό δυναμικό σε σχέση με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, τώρα, τι έχει θεσπιστεί ήδη, μας μιλήσατε για το τι ισχύει στους λιμένες, οι διάφορες εταιρείε έχουν δικά τους συστήματα και επιτρέπεται έτσι η ροή των πληροφοριών και οποιοδήποτε τέτοιο βήμα έχει γίνει νομίζω θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη και να ενισχυθεί. Επίσης σας είπα ε, προηγουμένως ότι έχουμε ένα εμπορικό τμήμα και ασχολούμαστε επισταμένα με την κατάρτιση προσωπικού και ανάπτυξη ανάπτυξη ε, ικανοτήτων. Συνεργαζόμαστε με πολλού φορεί ε, και ε, επίση ένα άλλο θέμα που μα απασχολεί είναι η χρήση των νέων τεχνολογιών. Γιατί έχει προχωρήσει η τεχνολογία, ο ιδιωτικό τομέα έχει υιοθετήσει, παραδείγματο χάρη, τη μονοπευθυντική θηρίδα που βασι... με έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιείται το υπολογιστικό νεφο, το cloud computing. Αυτό δημιουργεί νέε δυνατότητε σχετικά με την χρήση των νέων τεχνολογιών τη πληροφορική για τη διευκόλυνση του εμπορίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ε, ομιλητές για τις ενδιαφέρουσες αυτές ε, παρουσιάσεις. Έχουμε και το υλικό σας, να το εξετάσουμε. Υπάρχει λίγος ε, χρόνος, πρέπει βεβαίως 12.30 να τελειώσουμε. Οπότε υπάρχει λίγος χρόνος για συζήτηση. Η κυρία Χαντσλίκ έχει ήδη κάποιες ερωτήσεις και ο κύριος Σαλβίνη θα κάνει κάποια δήλωση. Δεν ξέρω αν οι άλλοι συνάδελφοι έχουν ερωτήσει. Α ξεκινήσουμε με την κυρία Χάντσλικ. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και όλους τους ομιλητές. Οι ήταν πολύ ενδιαφέρουσες. Έχω άλλο ένα ερώτημα πάλι εξ ονόματος κυρίας Κόρχολα και απευθύνομαι προς όλους τους ε, ομιλητές. Χωρίς ε, δικαιοσύνη εναντίον και ίσως όρους ανταγωνισμού ε, ως προς τους ανταγωνιστές μας, η ευρωπαϊκή βιομηχανία θα υποφέρει όσον αφορά τους υπόλοιπους ανταγωνιστές της στον κόσμο, γιατί οι υπόλοιποι βεβαίως δεν θεωρούν τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε ως δεσμευτικούς ή αρκετά ε, σαφής. Για πολλά προϊόντα λοιπόν είναι εύκολο να λυθεί αυτό το πρόβλημα με την επιτήρηση Τη ε, αγορά, ε, τη στιγμή κατά την οποία μπαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένα προϊόν. Βεβαίως μια ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ τελωνιακών διοικήσεων και αρχών επιτήρησης αγοράς είναι κρίσιμη. Οπότε αυτό το οποίο θέλει να ρωτήσει η κυρία Κορχολά είναι το εξή. Θεωρείτε πως μια τέτοια ενισχυμένη συνεργασία λαμβάνει χώρα ήδη. Μπορείτε να μας δώσετε συγκεκριμένα παραδείγματα τέτοια συνεργασίας για να έχουμε ένα πλαίσιο αναφοράς για το μέλλον. Και το δεύτερο ερώτημα της συναδέλφου. Κάποια κράτη-μέλη είναι κόμβοι ε, διαμετακομιστικοί από τρίτες χώρες. Γι' αυτό η αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ τελωνιακών αρχών και αρχών υποπτίας της ε, αγοράς ε, θα μπορούσε να έχει πολλά ωφέλη όχι μόνο για αυτές τις χώρες αλλά για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρείτε πως ε, θα μπορούσαμε να έχουμε παραδείγματο χάρη ε, να κάνουμε ένα τεστ και να έχουμε το ίδιο προϊόν σε πέντε διαφορετικά σημεία εισόδου και να δούμε πώς μπορεί να οργανωθεί αυτή η συνεργασία. Θεωρείτε πως υπάρχει δυνατότητα να γίνει κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσετε τον λόγο για να κάνω τις ερωτήσεις εξ ονόματος και τους Ευχαριστώ. Θα δούμε ποιος άλλος θέλει να κάνει ερωτήσεις, αλλά θα ζητήσω και από τον Δόκτρα Χόμπιν να σχολιάσει γιατί για το ζήτημα της συνεργασίας ανέφερε κάποιες πτυχές συνεργασίας στους συνοριακούς ελέγχους. Καλό θα ήταν λοιπόν να ακούσουμε και τη δική του άποψη. Ποιο άλλο λοιπόν θέλει να κάνει ερώτηση στην Κομισιόν, κύριε Σαλβίνη. Μα, Ναι, να εκφράσω μια σκέψη. Έχουμε μπροστά μας σκληρή δουλειά, γιατί τουλάχιστον στο ίμιση των παρεμβάσεων άκουσα ότι η αναστολή που ζητείτε ε, από την Κομισιόν ε, είναι καθήκον και δεν ε, είναι κάτι κακό γιατί δεν θα θέλαμε τελικά να επιβάλλουμε μία τροποποίηση που αντί να διευκολύνει τη ζωή των εμπορευομένων θα τους δυσκολέψει και επίσης ε, θα πρέπει ουσιαστικά να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ και κρατών μελών αλλά και εμπορευομένων. Άκουσα και από, άλλους, και από κάποιους άλλους ότι πρέπει να διασφαλίσουμε επίσης και τα συμφέροντα των μεμονωμένων κρατών μελών αλλά και την προστασία των καταναλωτών ταυτόχρονα διασφαλίζοντας ότι δεν καθιστούμε πιο πολύπλοκη τη ζωή των ε, επιχειρήσεων που εμπορεύονται νόμιμα. Τώρα, μια ερώτηση για τους πόρους για το κόστος της επικαιροποίησης του προσωπικού, για την κατάρτιση του προσωπικού και για την αύξηση του προσωπικού. Θα ήθελα να καταλάβω δεδομένη της οικονομικής κατάστασης πολλών κρατών μελών πώς ε, θα καλυφθεί αυτό το κόστος ε, για την ε, κατάρτιση του προσωπικού και για την επικαιροποίηση ενώ έχουμε σήμερα 27 διαφορετικά συστήματα έτσι λοιπόν ε, μου έρχεται κατά νου η αμφιβολία ότι πέρα από ε, οποιαδήποτε τυπική αναστολή μήπως ε, μπαίνουμε και σε κάποια ουσιαστικά θέματα γιατί διαφορετικά διακινδυνεύουμε να έχουμε ένα έγγραφο το οποίο τελικά αντί να μας διευκολύνει και να μας οδηγεί στην εναρμόνιση θα καταστήσει τα πράγματα πιο δύσκολα. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, αναμένουμε λοιπόν τις συστάσεις σας. Άλλοι συνάδελφοι, να κάνω εγώ μια ερώτηση πριν δώσω το λόγο μετά ότι θα δώσω την ευκαιρία στα μέλη του πάνελ να σχολιάσουν και στον κύριο Χόμπιν για το θέμα των ορών πληροφοριών. Α, κυρία Ρούλε, συγγνώμη, δεν σας είδα. Και εγώ θα είμαι σύντομη. Θεωρώ πως υπήρχαν κάποιες αντιφάσεις ε, σε αυτά τα οποία ακούστηκαν Αφενός είπατε πως είναι αναγκαίο κάποια πράγματα να γίνουν πιο απλά. Από την άλλη όμως από την Ολλανδία ακούστηκε η κριτική πως ε, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη τυποποίηση και δεν υπάρχει πάντα βάση για αυτή την τυποποίηση. Ε, εκεί πέρα εγώ αυτό το βλέπω σαν αντίφαση. Και μετά θέλω να πω πως ε, έχω την εντύπωση πως περιμένουμε πάρα πολλά από αυτό τον τελωνιακό κώδικα, ίσως υπερβολικά πολλά πράγματα και θα πρέπει να είμαστε κάπως πιο ρεαλιστές από όλες τις πλευρές. Γιατί μόνο έτσι θα έχουμε επιτυχία. Αυτά έτσι ως παρατηρήσεις. Θεωρώ πως κομμάτι του προβλήματος είναι και πολύ υψηλέ ε, προσδοκίες. Ναι. Ευχαριστούμε. Υπάρχουν και άλλα βεβαίως τέτοια σχόλια που θα τα δούμε. Εγώ ήθελα να αναφερθώ σε αυτό το οποίο ακούστηκε στη συνεργασία, για τη συνεργασία με τις επιχειρήσεις. Και σημαντικό ήταν όταν επισκεφθήκαμε διάφορα τελωνία. Ήταν το ζήτημα των νέων μέσων αξιολόγησης κινδύνου. Νομίζω ο κ. το ανέφερε, ο κ. Σέλστα. Πως ε, ειδικά το πρόβλημα πως οι αρχές επιβολής ε, θα πρέπει να ξέρουν ποια, αρχεία, ποια φορτία με πρέπει να ανοίξουν και ενδιαφέρον είναι πως ε, βεβαίως θα πάω μετά ε, στη συνάντηση των αρχών που παρακολουθούν την ασφάλεια των προϊόντων γιατί γιορτάζει η ομάδα του στα 20 χρόνια. Αλλά θεωρώ πως θα έπρεπε οι επιχειρήσεις να δίνουν στοιχεία σε αυτά τα μέσα αξιολόγησης κινδύνου, γιατί θα βοηθούσε γενικότερα και θα ήταν και προς το συμφέρον των επιχειρήσεων να φροντίσουν ε, έτσι ώστε προϊόντα μη ασφαλή που παροβιάζουν πνευματικά δικαιώματα να σταματάνε στα σύνορα και με με προξενεί εντύπωση το γεγονό πω δεν ε, συμμετέχουν τόσο οι επιχειρήσει. Σχετίζεται με την εσωτερική οργάνωση των επιχειρήσεων. Η μόνη επιχείρηση εδώ πέρα είναι η Microsoft από ό,τι βλέπω, που ανέφερε κάποια ζητήματα. Οπότε ο κύριο Κόλμπερτ θα ήθελε ίσω να σχολιάσει πω, τι κάνει η Microsoft για τις πληροφορίε που δίνει. για ζητήματα επιβολής ε, Θα ήθελα λοιπόν να μάθω ποιε είναι οι υποθέσει με τις αρχές. Η κυρία Σπέντιφ μας έδειξε ε, τη διαφάνεια όπου υπήρχαν 23 διαφορετικές αρχές. Υποψιάζομαι λοιπόν οι άνθρωποι που ασχολούνται με τις αποστολέ αγαθών σε επιχειρήσει δεν έχουν τις επαφές ίσως που θα έπρεπε να έχουν. Οι δε μεγάλε εταιρείε έχουν τι δικέ του εσωτερικέ τις λειτουργίε που δεν είναι τέλος πάντων αντικείμενό μας. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο θα ήθελα να κάνω λοιπόν να ζητήσω από τον Δ. Χόμπινγκ που ακούει τόση ώρα υπομονετικά να κάνει μια σύντομη παρέμβαση. Θα παρακαλέσω μετά ο καθένας να τοποθετηθεί για ένα λεπτό γιατί χρειάζεται χρόνος ε, για να ολοκληρώσει και ο εισηγητή. Θα σας πούμε όταν τελειώνει ο χρόνο. Ο Δ. Χόμπινγκ πρώτα απ' όλα. Ναι, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Πρόεδρε. Πολύ σύντομο ε, θα είμαι. Θέλω να αναφερθώ σε ένα σημείο το οποίο έθιξαν και πολλοί ομιλητέ, αλλά και ο κύριο Σελβίνη. Είναι το θέμα των χρημάτων. Ακούσαμε ότι πολλές από τις ε, καλές βελτιώσεις ε, που έχουν σχεδιαστεί αναστέλλονται και λόγω έλλειψης σπόρων και άκουσα από 7 μιλητές ότι περισσότερες από τους σπόρους αυτούς που χρειάζονται για τη χρηματοδότηση προέρχονται από τα κράτη-μέλη. Εγώ δεν εργαζόμαι μόνο στα τελωνία, αλλά και από την άλλη πλευρά, δηλαδή στο χώρο Σέγγεν. Και αν δείτε πάνω από το φράχτη, θα δείτε ότι υπάρχουν ε, πολλά διαθέσιμα χρήματα. Έχουμε το ταμείο, το συνεργατικό ταμείο για τη Σέγγεν, το οποίο δίνει 1,5, έχει 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ για την περίοδο μέχρι το 2013. Έχουμε λοιπόν ε, πολλούς σπόρους που έχουν χορηγηθεί για την ανάπτυξη του Eurosur. Νομίζω λοιπόν ότι θα ήταν καλό αν και οι πολιτικοί συνειδητοποιήσουν ότι και τα τελωνία ε, επιτελούν αποστολή τήρησης της ασφάλειας και ίσως θα έπρεπε να πάρουν και ένα κομμάτι της πίτας και από την άλλη πλευρά. Αυτή είναι η πρότασή μου, προσέξτε το. Ναι, είναι ίσω μια ευπρόσδεκτη πρόταση. Αν δεν μπορούσαμε να πετύχουμε κάτι, θα το συζητήσουμε με του συναδέλφου από την Επιτροπή Προπολογισμού. Λοιπόν, α προχωρήσουμε. Α ξεκινήσουμε από το τέλο, από τον κύριο κάλβερτ και θα καταλήξουμε στον κύριο Καστρεσινάκη. Παρακαλώ, ένα λεπτό έχετε. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Εγώ ως διεθνής εμπορευόμενος, εκπρόσωπος διεθνής εμπορευμένου της, ε, ενδιαφέρεται η επιχείρησή μου να αυξήσει την ασφάλεια, να προστατεύσει τα πνευματικά δικαιώματα και έχει δημιουργήσει ένα τρόπο εργασίας, ανάπτυξης συστημάτων για την ε, υποστήριξη αυτών των στόχων, αλλά και ως εταιρεία συμμετέχουμε ενεργά στον ΠΟΕ, στον ΠΟΤ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και προβαίνουμε και στην ανταλλαγή βελτιστών πρακτικών και στην οικοδόμηση δυνατοτήτων. Τώρα, για την ερώτησή σα για την ανταλλαγή πληροφοριών, πιστεύουμε ότι το πλαίσιο τη διαχείριση των κινδύνων πράγματι είναι ένα στοιχείο συνεργασίας. Εκεί βλέπουμε ότι οι ιδιωτικέ εταιρείε μπορεί να έχουν στη διάθεση του πληροφορίε, μπορεί να τις πουλήσουν έναντι αντιτίμου και αυτό μπορεί να συνδυαστεί με άλλες πληροφορίες που να είναι χρήσιμες για τα τελωνία ή για τον ΠΟΤ. Μπορούμε να έχουμε και μοντέλα intelligence, ε, στρατηγικό πληροφοριών. Φυσικά εμείς είμαστε πρόθυμοι να συμμετάσχουμε και να παρέχουμε αυτές τις πληροφορίες έτσι ώστε να λειτουργεί το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνου αποτελεσματικά. Και να έρθω και στην αρχή της διαλειτουργικότητας, δηλαδή ανταλλαγή πληροφοριών. Ο τρόπος ανταλλαγής πληροφοριών από τη σκοπιά της ασφάλειας, ε, αλλά και από άλλες σκοπιές, είναι κάτι που θέτει προκλήσεις, γιατί έχουμε διαφορετικές απαντήσεις ασφαλείας. Ε, εμείς ε, από αυτή την σκοπιά, ως εμπορευόμενοι δηλαδή, έχουμε ένα πρόβλημα εκεί, αλλά προσπαθούμε να συμμετέχουμε ενεργά. Η κυρία Σπέντιφ, ε, θα αναφερθώ σε δύο τομείς για το θέμα της συνεργασίας με τις επιχειρήσεις. Νομίζω ότι έχετε απόλυτο δίκιο. Και εμείς θεωρούμε συχνά ότι οι επιχειρήσεις ε, δεν ε, είναι τόσο ενωμένες όσο εμείς ε, υποθέτουμε σε εσωτερικό επίπεδο. Δεν είναι τόσο οργανωμένες. Και επίσης, να σας πω ότι τα τελωνία δεν κάθονται στο Συμβούλιο για να συμμετάσχουν εκτός αν πάει κάτι λάθος. Νομίζω ότι η διαχείριση των κινδύνων είναι ο τρόπος να τετραγωνίσουμε τον κύκλο. Είναι ο τρόπος να κινηθούμε στο μέλλον για να βρούμε τους ψήλους τάχυρα αλλά πάντοτε πρέπει να προωθείτε με τις στρατικές πληροφορίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα να στηρίξω και εγώ αυτό το οποίο είπε ο κύριος Σχόμπινγκ πως τα τελωνία έχουν πολύ ευρύτερη δουλειά από την ανταγωνιστικότητα. ασχολούμαστε και με την ασφάλεια και στο ευρωπαϊκό επίπεδο μπορεί να γίνουν ακόμη πολλά πράγματα στο συντονισμό και τη χρηματοδότηση αυτού του τομέα για πιθανές αντιφάσεις αυτά τα οποία είπα περί τυποποίησης υπάρχει διαφορά μεταξύ τυποποίησης και εναρμόνισης. Πρέπει να δράσουμε ενωμένοι ως ευρωπαϊκά τελωνία, αυτό είναι η εναρμόνιση, αλλά τα μέσα τα οποία χρησιμοποιούμε ε, δεν θα πρέπει να είναι, θα πρέπει να είναι τυποποιημένα, αλλά να υπάρχουν ε, διαφορετικές δυνατότητες ανάλογα με το μέσο μεταφοράς και τις δυνατότητες επιμελητίας του καθενός. Καθώς ο κύριος Καλβέρτ εκπροσωπεί μεγάλη εταιρεία, ε, είπε πως είναι δυνατόν να υπάρχουν ε, διαφορετικές λύσεις και όχι μόνο μία τυποποιημένη. Μάλιστα. Βεβαίως και η διαλειτουργικότητα είναι εδώ πέρα ένα ζήτημα. Ο κύριος Ζωγράφος. Πέρα για τους ελέγχους και σε αυτό το τομέα θα μείνω. Έχω τη γνώμη ότι γενικά τα τελωνία στην Ευρώπη, πέρα την Ευρώπη, αλλά κυρίως στην Ευρώπη, βρίσκονται σε αρκετά ευαίσθητη και κρίσιμη θέση. Από τη μια μεριά καλούνται να διευκολύνουν με τις απλουστεύσεις και όλες τις λοιπές διαδικασίες στην ταχεία και σωστή διεκπαιρέωση των τελωνιακών ε, εργασιών και γενικότερα στη μεταφορά για τη διακίνηση των αγαθών και, και σωστά. Και από την άλλη πλευρά καλούνται επίσης να φροντίζουν για να περνούν σωστά εμπορεύματα, υγιείς τροφές, μία απαγορεύσιμα και μία κατάλληλα υλικά στον κόσμο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να εισπράττονται φυσικά και δασμοί και οι φόροι. Επιτρέψτε μου να επιμείνω ότι ο σωστός, κατάλληλος, με τα μέσα τα σύγχρονα, έλεγχος είναι απολύτως απαραίτητος. Χωρίς σωστούς ελέγχους θα βρεθούμε σε πολύ δύσκολη θέση και σαν κοινωνία και σαν υπηρεσίες, αλλά γιατί όχι και σαν ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν θα εισπράττει τα χρήματα τα οποία πρέπει μέσω του λαθρεμπορίου, μέσω της απάτης, μέσω της φοροδιαφυγής. Νομίζω σωστή και ευέλικτη έλεγχη και γνωρίζει πολύ καλά η αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης τι εννοώ, είναι απαραίτητη για να διασφαλίσουμε στο μέλλον κανονικές, σωστές, αποδοτικές και γρήγορες τελωνιακές διαδικασίες. Ε, Elster. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ θα αναφερθώ στα ερωτήματα της συνεργασίας και του τεστ που αναφέρατε. Κάποιες χώρες που έχουν πολύ καλή... Υπάρχουν χώρες που έχουν πολύ καλή συνεργασία μεταξύ τελωνίων και αρχών ε, παρακολούθησης αγοράς όπως π.χ. η Ολλανδία και η Γαλλία αλλά αλλού στην Ορβηγία ας πούμε υπάρχει μεγαλύτερη απόσταση γιατί οι αρχές επιτήρησης της αγοράς αντλούν ε, τη χρηματοδότησή τους από τη δική τους δραστηριότητα και όχι από κάτι που σχετίζεται με τα σύνορα. Οπότε εστιάζονται στην αγορά και όχι στα σύνορα. Οπότε όλος ο οργανισμός ε, είναι αλλού προσανατολισμένος. Και καμιά φορά πρέπει να αντλήσουμε διδάγματα πριν ε, συνεργαστούν οι δύο οργανισμοί. Τέλος πάντων για τεστ, όπως είπατε, εισαγών. Νομίζω πως αυτές τις μέρες ε, η ProSafe κάνει τεστ για την εισαγωγή αναπτύρων και μπορούμε άρα να έχουμε κάποιες απαντήσεις ε, στο ερώτημά σας και να δούμε το τι κάνει η κάθε χώρα με τις ε, εισαγωγές. Uh, Ο κύριος Ραμάλου. Καταρχήν, λοιπόν, ενία δίκηση όχι μόνο για την ε, εφαρμογή του κοινού τελωνιακού ελέγχου, αλλά να συνδέεται και με 27 κράτη. Αυτό απαιτεί μία επίσης ενία ρύθμιση και οι ιδιαιτερότητε, ε, όπως υπόθηκε πριν τους χάρη στο λιμόνι του Ρότερνταμ, δεν πρέπει να ρυθμίζονται από τις χώρες, αλλά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ρυθμίσει τι γενικέ, αλλά και τι ειδικέ διαδικασίε ε, για τι διάφορε περιστάσει που μπορούν να προκύψουν. Τώρα, παγκόσμια ανταγωνιστικότητα έχουμε την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον υπόλοιπο κόσμο, όχι μεταξύ των διάφορων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνολό της. Τρίτο. Συμφωνώ με τη διευκόλυνση του εμπορίου, αλλά δεν μπορεί να είναι εις βάρος ε, διαφορετικής μεταχείρισης μεταξύ των διάφορων χωρών. Σας ευχαριστώ. Και τώρα ο κύριος Καστιστριανάκης για την Κομισιόν. Απλώς ε, θέλω να ελέγξω αν ε, κάποιοι από τους προηγούμενους θέλουν το λόγο για κάτι από όσα ακούσαμε πριν τον κύριο Καστιστριανάκη. Ένα λεπτό έχετε. Yes, Μάλιστα. Ε, ε, ε, έθεσε μία ερώτηση κάποια κυρία, αλλά έχει αποχωρήσει το μεταξύ. Θα βγάλω το καπέλο του μέλου της ομάδας επαφής για το εμπόριο. Έτσι εκπροσωπώ την εταιρεία μου μιλώντας τώρα. Λοιπόν, η κυρία αυτή μας μίλησε για τους συνοριακού ελέγχους. Οι έλεγχοι γίνονται πλέον στα σύνορα. Αλλά ο γόρδιος δεσμός στην Ευρώπη είναι ότι έχουμε δύο διαφορετικά σύνορα και οτιδήποτε έχει σχεδιαστεί για τις επιχειρήσεις υποτίθεται ότι καλύπτει την, τα θέματα ασφάλειας ε, και προστασίας ε, στο σημείο άφηξη, στο πρώτο, στον πρώτο σταθμό που μπορεί να είναι σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ένωσης και κατόπιν ακολουθεί η αποστολή, την όλη διαδικασία μέχρι τον τελικό προορισμό. Όλες οι αποστολές που αναλαμβάνουμε δηλαδή ε, υπάγονται σε δύο διαφορετικές αναλύσεις κινδύνου. Με τον εξυγχρονισμένο κώδικα έχουμε τη δυνατότητα τεσσάρων σημείων διεξαγωγής ε, ανάλυσης κινδύνου. Πρόεδρος. Μα θέσατε και ένα άλλο ένιγμα και άλλο ένα γόρδιο δεσμό στο με αυτό που είπατε. Ο κύριος Σαλβίνη σίγουρα ε, θα το σχολιάσει αυτό το θέμα. Ας ακούσουμε τον κύριο Καστριτσιανάκη από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής πριν ολοκληρώσουμε. Ίσως ε, θέλετε να σχολιάσετε κάποια από τα ζητήματα που σχολιάστηκαν και ο κύριος Σαλβίνη μετά θα πάρει το λόγο για τις καταληκτικές ε, παρατηρήσεις. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι θα συμφωνήσουν όλοι πως για τα θέματα ασφάλειας και προστασίας και το πρώτο σημείο εισόδου Εκεί είναι το σημείο που πρέπει να διεξαχθεί ο έλεγχος για την ε, διαχείριση, ανάλυση και διαχείριση κινδύνου. Τρεις παρατηρήσεις θα ήθελα να κάνω, η συντομία. Σχετικά με τους ε, περιορισμούς, την ασφάλεια και την ε, διυπηρεσιακή συνεργασία, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεξεργαζόμαστε ένα σετ βελτίστων πρακτικών και προσπαθούμε να εκπονήσουμε κατευθυντήριες γραμμές για τις τελωνιακές διοικήσεις σχετικά με το πώς να ε, αναβαθμίσουν την αποτελεσματικότητά τους και ελπίζουμε να τα έχουμε καταφέρει μέσα στο 2011. Επίσης, η χρήση του ε, κοινού συστήματος διαχείρισης κινδύνους Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενθαρρύνουμε τη χρήση του, ώστε οι τελωνιακές αρχές να μπορέσουν να ανταλλάσσουν ευκολότερα πληροφορίες σχετικά με το κίνδυνο και τις ε, διακρατήσεις ε, εμπορευμάτων από τους τελωνιακούς σταθμούς. Αυτό που άκουσα και βρήκα ενδιαφέρον είναι πώς θα μπορούσε να εμπλακεί ο κλάδος, ο ιδιωτικός τομέας στην όλη προσπάθεια. Νομίζω ότι θα έπρεπε όλοι να το σκεφτούμε, δηλαδή σε ποιο βαθμό αυτό είναι καλή ιδέα και εφικτή κυρίως. θα τα χρησιμοποιούμε ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον συνεργασία με άλλου διεθνού οργανισμούς, ε, σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τελωνίων και φυσικά όλε οι υπηρεσίε τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής επεξεργάζονται αυτό το θέμα. Κατόπιν, για του συγκεκριμένου οικονομικού φορεί. και πάλι εδώ θα έλεγα ότι ε, το, είναι νέο το σύστημα, καινούργιο το σύστημα, δεν έχουμε μακρά ε, εμπειρία. Θα μπορέσουμε υπό το φως της εμπειρίας μας σε κάποια στιγμή να εξετάσουμε τα αποτελέσματα μας απασχολεί το θέμα της αμοιβαίας αναγνώρισης σχέσεις μας με τις τρίτες χώρες ε, η ΕΠΑ, ΕΕ, η Ιαπωνία, Καναδάς, ε, Νορβηγία, Ελβετία είναι χώρες που σίγουρα ε, είναι στον κατάλογο αυτό. Τώρα σχετικά με την ερώτηση αν χρειαζόμαστε όλες αυτές ε, τις ε, πληροφορίες για τη διαχείριση κινδύνου, δηλαδή οι πληροφορίες προάφηξης. Ε, αυτή την ερώτηση θέσατε, τις χρειαζόμαστε όλες αυτές τις πληροφορίες από πλευρά σας. Λοιπόν, θα απαντούσα το εξή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε πολυεπίπεδη προσέγγιση για τη διαχείριση του κινδύνου, να συνδυάσουμε διάφορα στρώματα και να μην επαφιέμεθα σε ένα μόνο εργαλείο το σκανάρισμα 100% παραδείγματος χάρη. Επίσης πρέπει να δούμε εγκαιρός ε, τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι μπορούμε να εντοπίσουμε το εμπόρευμα ε, και φυσικά ε, το ποιος το συσκεύασε. Οι πληροφορίες λοιπόν που παρέχονται είναι απαραίτητες και θα έπρεπε να αναπτύξουμε περαιτέρω το σύστημα και να το βελτιώσουμε. Να βελτιώσουμε αυτά τα εργαλεία διαχείρισης του κινδύνου για να χρησιμοποιούνται από κοινό, από όλα τα κράτη-μέλη και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουμε και ε, τις πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών, ε, των εθνικών υπηρεσιών ε, πληροφοριών ε, σε αυτή τη διαδικασία. Θα σταματήσω εδώ. Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε όλους για τη συμβολή σας στη σημερινή ακρόαση. Ευχαριστούμε τον κύριο Σαλβίνη γιατί ηγείται των προσπαθειών από πλευρά του Κοινοβουλίου. Θα του δώσω λοιπόν το λόγο για να κάνει κάποιες καταληκτικές παρατηρήσεις και μετά θα ανακοινώσουμε το χρονοδιάγραμμα των εργασιών μας. Ευχαριστώ. Αναμένοντας να βρω το μαγικό ραβδί το οποίο ουσιαστικά θα συνδυάσει μαγικά όλες ε, τις ιδέες. Έτσι δεν θα σας πω ότι ε, χαίρομαι που είμαι από το Μιλάνο και που δεν έχετε έξοδο στη θάλασσα. Ε, τέλος πάντων, ε, χαίρομαι πάρα πολύ που εδώ ακούσαμε διάφορες ιδέες και από τους εμπεριβομένους αλλά και από εκπρόσωπους της, πολιτικής. της πολιτικής. Έχουμε χρόνο το καλοκαίρι για να καταθέσουμε το έγγραφο δεν ε, ε, θα αναφέρω στο τώρα λεπτομερό σε όλες αυτές τις ιδέες που αναφέρθηκαν στο ότι πρέπει να ενερμονίσουμε αλλά όχι να τυποποιήσουμε γιατί είναι δύσκολο να περάσουμε από το 27 σε ένα σύστημα. Σας ευχαριστώ για όλες τις ιδέες ε, και είναι πολύ πιο σημαντικές αυτή τη στιγμή γιατί πρέπει να κατορθώσουμε να έχουμε ένα συνθετικό κείμενο αλλά νομίζω θα τα καταφέρουμε και με τη βοήθεια του Προέδρου αλλά και της γραμματείας. Λοιπόν, να κλείσω λέγοντας ε, καταρχήν, ε, και αυτό είναι για το ευρύτερο ε, ακροτηριό μα ότι όλες οι παρουσιάσει θα μπουν στην ιστοσελίδα έτσι όλοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στις διαφάνειες που μας στείλετε έχουμε και αντιγραφά της ε, μελέτη του κυρίου Χόμπινγκ αν θέλετε μπορείτε να την πάρετε φεύγοντας ε, αφορά το ρόλο του Λεωνίου και τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων υπάρχουν και αντίγραφα του newsletter τη Επιτροπή μα και βέβαια αν θέλετε ευχαριστώ να εγγραφείτε για να λαμβάνετε τακτικά το αντίγραφο και το ηλεκτρονικό ε, αντίτυπο σας προσφέρει και σύνδεση ε, live. Σας ευχαριστώ όλους που ήσασταν εδώ Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε μαζί σας. Ο κύριος Σαλβίνη θα εκπονήσει την έκθεσή του και θα την ολοκληρώσει μέχρι τι 19 Σεπτεμβρίου. Έχει καιρό, έχει χρόνο στη διάθεσή του. Κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών σας θα σκέφτετε όλα αυτά που τίποτα. Δεν ξέρω αν θα είναι στη θάλασσα ή όχι, θα το δει ο ίδιο. Έχουμε 23 Σεπτεμβρίου προθεσμία για τις τροπολογίες και θα ψηφίσουμε τον Οκτώβριο στην Επιτροπή. Αν έχετε περαιτέρω σκέψεις, ε, παρακαλώ να ε, μας τις στείλετε και ε, ελπίζω σήμερα να σας δώσαμε και την ευκαιρία να γνωριστείτε όσοι δεν γνωριζόσασταν από πριν, έτσι ώστε να συνεργαστείτε και στο μέλλον. Έτσι λοιπόν, ολοκληρώνεται εδώ η συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Η επόμενη πλήρη συνεδρίαση της Επιτροπής μας θα είναι στις 11 Ιουλίου. Και ο Πρόεδρος ευχαριστεί ευγενικά τους διερμηνείς. Ευχαριστούμε και εμείς. Αντίο. Έχουμε τον ε, Υφυπουργό της Πολωνίας που θα παρευρεθεί για πρώτη φορά στη συνεδρίασή μας ε, ασκώντας ε, την εκπεριτροπής Προεδρία και εκπροσωπούνται στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας.